Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι, καλωσορίζω ήδη ε, ενώπιόν μας τον Επίτροπο, τον κύριο Μοέδας. Πριν του δώσω όμως το λόγο, θέλω να τον ευχαριστήσω για την υπομονή. Ε, να παρακαλέσω σύντομα τον κύριο Μαρινέσκου να μας δώσει μια σύντομη επισκόπηση για τον πρώτο τριμερή διάλογο για την Όλαφ, δηλαδή τα πρώτα θέματα που θίξατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you, Chair. So Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είχαμε την πρώτη συνεδρίαση του Τριμέρου διαλόγου. Ε, συζητήσαμε τα πρωτα έξεπτα άρθρα. Επιτύχαμε σε δύο-τρία από αυτά, για τα υπόλοιπα όχι. Έχουμε κάποιες συζητήσεις Ε, σχετικά με τα αιτήματα του Κοινοβουλίου για την εισαγωγή των παρατυπιών και να αλλάξουν και κάποια ονόματα ε, και χαρακτηρισμοί σχετικά με τις έρευνες που γίνονται εσωτερική και εξωτερική. Αυτά ήταν τα βασικά θέματα που μας απασχόλησαν. Γενικά νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε. Ήδη έχω προγραμματίσει τεχνικές τέτοιες συνεδριάσεις, άλλες δύο με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, από Δεκέμβρη. Ε, ελπίζω να έχω καλύτερα νέα να σας πω. Αυτά. Και φυσικά έχουμε και εσωτερικές συνεδριάσεις με τους συναδέλφους του Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ερωτήσεις έχετε στο συνάδελφο Μαρινέσκου. Βλέπω όχι. Λοιπόν, σου ευχόμαστε πάρα πολύ καλή επιτυχία και καλή τύχη. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Οπότε, επανερχόμαστε στην απαλλαγή, που είναι το σημείο 15, ε, λέει η Πρόεδρος. Ε, καλωσορίζω από το ελεκτικό συνέδριο τον κύριο Μιχάηλ Σκόσλοφς, που είναι ορμόδιος για το θέμα αυτό στα πλαίσια του ελεκτικού συνεδρίου. Ε, που ασχολείται με τα θέματα ορίζων και λοιπά, δηλαδή έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία και επιστήμης και χαίρομαι που ήρθε και ο Επίτροπος ο κύριος Μουέδερς, για να συζητήσουμε τα προγράμματα που έχετε να διαχειριστείτε και που είναι στη δική σας ευθύνη. Είναι από τα ε, ε επιτυχέστερα που έχουμε. Και γιατί καθυστέρησα, ε, γιατί έτρεχα και αγωνιζόμουν για το ορίζον 2020 στα πλαίσια ε, της διαδικασίας του προϋπολογισμού που ελπίζω να ολοκληρωθεί την Παρασκευή υπέρ της επιστήμης, της έρευνας και της καινοτομίας. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Κόσλοφς και μετά στον Επίτροπο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, αγαπητέ Επίτροπε, ε, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς, ε, να σας πω ότι χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ και μπορώ να καλωσορίζω και τα νέα αλλά και παλιά μέλη της Επιτροπής σας που επανεξελέγησαν και να επαναλάβω και πάλι την προσήλωση και τη δέσμευση του ελεκτικού συνεδρίου ε, να σας βοηθάει και την Επιτροπή σας και το Κοινοβούλιο. Στην κατηγορία 1α, οι δαπάνες υποστηρίζουν τις φιλοδοξίες, ηγετικές φιλοδοξίες που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ε, πολλούς τομείς πολιτικής. Καταλαμβάνει μεγάλο τμήμα του προπολογισμού ε, και ακόμα περισσότερο στο μέλλον, ακόμα μεγαλύτερο. Από τη σκοπιά ε, του συνεδρίου οι τακτικές δαπάνες και συμμορφούμενες με τους κανόνες είναι πολύ σημαντικές για να αξιοποιήσουν όσο γίνεται καλύτερα τα κράτη-μέλη τους πόρους που τους διατίθενται. Γι' αυτό χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να σας παρουσιάσω τα αποτελέσματα ε, του ελέγχου μας για το 2018. Καταρχάς, πολύ σύντομα να σας πούμε τι κάνουμε είχαμε τέσσερις ε, βασικούς τομείς, ας πούμε, κεφάλαια ε, για τη δήλωση εξοπιστίας. Το πρώτο είναι κάτι που κάνουμε κάθε χρόνο, στάνταρ, που είναι ουσιαστική ε, δοκιμή και έλεγχο των υποκείμενων συναλλαγών. Είχαμε 130 συναλλαγές και βλέπετε και από την παρουσίαση πώς κατανέμονται αυτές οι συναλλαγές σε διάφορες δαπάνες. Στη δεύτερη ενότητα ε, αξιολογήσαμε τους ε, λογιστικούς ελέγχους Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκ των υστέρων για τον ορίζοντα 2020 και πώς ε, αυτό θα μεταφραστεί στο μέλλον. Εδώ αναθεωρήσαμε, αξιολογήσαμε 20 ελέγχους, έτσι δειγματοληπτικά, που έχει κάνει εκ των υστέρων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, αφορούσε αυτό τις πληρωμές και τις εκαθαρίσεις των λογαριασμών ε, της σχετικής χρονικής περίοδου. Στο τρίτο κεφάλαιο που ήταν πολύ σύντομο αναθεωρήσαμε τις ε, εκθέσεις πεπραγμένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ετήσιες διαφόρων γενικών διευθύνσεων και στη συνέχεια συλλέξαμε στοιχεία από το πρώτο κεφάλαιο σχετικά με την αποδοτικότητά του στο πρώτο module. Τα ευρήματά μας μπορείτε να τα δείτε στην αντίστοιχη έκθεση, στο αντίστοιχο κεφάλαιο. Ποια είναι τα βασικά μας τώρα συμπεράσματα, αποτελέσματα. Εκτιμήσαμε το επίπεδο σφάλματος για την κατηγορία 1α στο 2% για όλη την περίοδο. Δηλαδή παραμένει το σφάλμα σε επίπεδα που αξιολογούνται. Και σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, έχει πέσει μεν και αυτό το καλωσορίζουμε, αλλά πιστεύουμε ότι τα μέτρα απλούστευσης και ιδιαίτερα στον ορίζοντα 2020 θα μπορούσαν να είχαν συνεισφέρει προς την κατεύθυνση αυτή, προς τη βελτίωση αυτή. Έρχομαι τώρα στα γενικά συμπεράσματα. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι είναι υψηλού κινδύνου ο τομέας των δαπανών στην έρευνα και παραμένει η βασική πηγή σφαλμάτων. Παρά τις βελτιώσεις υπάρχει ακόμα χώρος για ενδεχόμενα σφάλματα και, και χωράει η βελτίωση σίγουρα. Νομίζω ότι θα συνεχίσουμε προς την κατεύθυνση αυτή να εργαζόμαστε ε, της βελτίωσης μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, όπως σας είπα, στα πλαίσια του δεύτερου κεφαλαίου, κοιτάξαμε τι γίνεται με τον λογιστικό έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην παρούσα φάση καταλήξαμε ότι δεν μπορούμε να βασιζόμαστε στους λογιστικούς ελέγχους που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όπως σας είπα, Ελέγξαμε 20 υποθέσεις δειγματοληπτικά και στις 10 από αυτές για διάφορους λόγους ε, καταλήξαμε ότι δεν μπορούμε να βασιστούμε στους εκ των υστέρων ελέγχους Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρά το συμπέρασμα αυτό, έχουμε την πρόθεση να επαναλάβουμε ε, ε, αυτή την άσκηση ε, για τη δήλωση αξιοπιστίας του 2019 για να έχουμε περισσότερα στοιχεία όπου θα βασίσουμε την εκτίμησή μας. Πάντως είναι σαφές ήδη ότι για το οικονομικό έτος 2019 δεν θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε την παλιά μέθοδο. Σε ό,τι αφορά τις πληροφορίες που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, αυτές επιβεβαιώνουν και τα ευρήματά μας και τα συμπεράσματά μας. Έχουμε τώρα στις βασικές συστάσεις μας. Τι προτείνουμε ε, να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα, τα λέμε και σε εσάς. Να έχει πιο στοχευμένους ελέγχους μικρομεσαίων επιχειρήσεων όταν έχουν κάποιες αξιώσεις αποζημίωσης και να γίνεται καλύτερη ενημερωτική εκστρατεία από πλευράς Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό έχει, κάνει, έχει να κάνει με το γεγονός ότι βρήκαμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα όσες για πρώτη φορά συμμετέχουν ε, σε τέτοια προγράμματα του Horizon 2020, τείνουν να κάνουν περισσότερα σφάλματα από εταιρείε που ε, ήδη λαμβάνουν χρηματοδότηση ή ε, έχουν λάβει στο παρελθόν. Δεύτερη σύσταση. Για το επόμενο ε, πρόγραμμα πλαίσιο της έρευνας καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, απλουστεύσει περαιτέρω ε, τους κανόνες για τον υπολογισμό του κόστους λειτουργίας, το κόστος προσωπικού μάλλον, γιατί εκεί έχουμε βρει πάρα πολλά σφάλματα. Και τέλος, η τρίτη σύσταση αφορά τον ορίζοντα 2020 πάντα και την αξιολόγηση που κάναμε των εκ των ελέγχων ως προς την τεκμηρίωση, ε, τη, συνέχεια, τη συνέπεια των δειγμάτων και την ε, αναφορά, καθώς επίσης και την ποιότητα των διαδικασιών λογιστικού ελέγχου. Νομίζω ότι μπορώ να σταματήσω εδώ την παρουσίασή μου και με χαρά να ακούσω οποιασδήποτε ερωτήσεις και σχόλια για να γίνει συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Thank you so much for your very... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύτιμη η δουλειά σας και τώρα θα δώσω το λόγο στον Επίτροπο, ε, τον Επίτροπο μας τον κύριο Μέδας για να απαντήσει για τις διάφορες ερωτήσεις και συστάσεις που έγιναν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Uh, σας ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμα μέλη, Κύριε Κοσλόφ, είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι εδώ ήταν πρέπει να σας πω ένα από τα ωραία σημεία της ε, θητείας μου να είμαι κοντά σας μια φορά το χρόνο. Χαίρομαι που ήρθα εδώ, βλέπω κάποιους από το παρελθόν, καλωσορίζω ε, τα καινούργια μέλη και πρέπει να σας πω πως είναι σημαντικό το θέμα για εμένα και σέβομαι πάρα πολύ τη δουλειά που κάνετε μια και εξασφαλίζετε πως όλα θα πάνε καλά. Η δουλειά σας είναι πάρα πολύ σημαντική για τον τρόπο με τον οποίο ε, αξιοποιείτε τα ευρωπαϊκά κονδύλια και διασφαλίζετε τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας εύχομαι λοιπόν καλή θητεία. Και να σας πω πως κάθε χρόνο έχω έρθει και σας έχω πει κάποιες ιστορίες. Ιστορίες που εξηγούν για ποιο λόγο τα κονδύλια αυτά είναι τόσο σημαντικά για τόσους ανθρώπους. και γιατί χρειαζόμαστε να συνεχίσουμε έτσι και στο μέλλον. Λοιπόν, το πρώτο που θα θυμηθώ πέρσι είναι το βραβείο Νόμπελ που δόθηκε στον καθηγητή Πίτερ Ράτκλιφ για την ιατρική. Και όταν του τηλεφώνησαν, του τηλεφώνησε ένας Άνταμ Σμιθ. Δεν είναι ο οικονομολόγος, αλλά είναι από την Επιτροπή των Βραβείων και τον ρώτησε τι κάνετε κύριε καθηγητά και είπε αυτή τη στιγμή ψάχνω ένα, μια επιχορήγηση συνέργειας και μόλις είχε πάρει το Νόμπελ. Δηλαδή το πρώτο που είπε είναι πως θέλει μια επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δουλειά του Ράτκλιφ είναι καταπληκτική. Αν δείτε τι γίνεται με τον καρκίνο και δυστυχώς όλες οι οικογένειές μας έχουμε και στο περιβάλλον μας τόσο πολλούς ανθρώπους που υποφέρουν αυτή την τρομακτική ασθένεια και ήρθε και είπε ψάχνω κάτι διαφορετικό. Θέλω να ε, μελετήσω το οξυγόνο στα κύτταρα και εξετάζοντας το επίπεδο οξυγόνου σε ένα κύτταρο μπορώ να ελέγξω καλύτερα και να λύσω το πρόβλημα Γιατί όταν λείπει οξυγόνο από ένα κύτταρο, έχει τελείως διαφορετική συμπεριφορά από ένα το οποίο έχει επαρκή ε, επίπεδα. Οπότε, βρήκε ένα καινούριο τρόπο για να αντιμετωπίσει τον καρκίνο, την ανεμία και πάρα πολλά ακόμα θέματα. Το άλλο ήταν τι κάναμε ε, τον Οκτώβριο. Εμείς είπαμε 6 εκατομμύρια συνεισφορά για μια δοκιμή εμβολίων στο Κονγκό ε, κατά του έμπολα. Και είναι ένα παράδειγμα το οποίο δίνω πάντοτε γιατί θυμόσαστε το 2014 πόσο δύσκολα ήταν τα πράγματα. Τώρα συνεχίζουμε να χρηματοδοτούμε γιατί και πάλι έχει ξεσπάσει ασθένεια ε, στο Κονγκό και θέλω να σας πω και μια ιστορία για την καινοτομία και για τις εταιρείε ε, που είναι πίσω τους. Αυτή τη στιγμή το πιλωτικό που κάναμε στο Συμβούλιο για την Καινοτομία είχαμε πολλές επιτυχίες. Πέρσι συναντήσαμε πάρα πολλές επιχειρήσεις και είναι δύσκολο να ε, πω ποια είναι η πιο καινοτόμα, αλλά έχουμε μία καινούρια η οποία έχει ε, φτιάξει ε, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, όχι μακριά από την ε, αγορά που πολλούν τα προϊόντα, αλλά κοντά σε αυτή την αγορά. Έχουν λοιπόν κάποια, κάποιες μικρές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες είναι μικρές, είναι αστικές και είναι δίπλα στο σημείο πώληση. Οπότε είναι πολύ μικρότερη ρήπανση από τη μεταφορά των προϊόντων. Εμείς χρηματοδοτήσαμε και μέσω αυτού κατάφεραν να μοχλεύσουν 88 εκατομμύρια ευρώ από επενδυτές. Ένας από τους λόγους ήταν γιατί πραγματικά πιστεύουν πως αν χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα βιώσιμο ε, project και γι' αυτό τους εμπιστεύτηκαν. Μετά θέλω να πω και κάποια πράγματα για το ελεγκτικό συνέδριο. Να σας πω πως για αυτή τη φορά Ε, συμπίπτω με τα αποτελέσματα της έκθεσής τους που είπε πως ε, το προϋπολογισμός έρευνας και τεχνολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέτος, την προηγούμενη χρονιά, δαπανήθηκε πιο ορθολογικά από ό,τι περασμένα έτη. Αυτό. Δεύτερον, το ποσοστό σφάλματος. Θυμάμαι να έχω έρθει εδώ πριν από κάποια χρόνια και ήμασταν στο 5,6%. Και πρέπει να σας πω ότι πονούσε η καρδιά μου. Ήμουν σαν όμουν νευρικός, ε, κοιτούσα τη Μαρτίνα από το ελεγκτικό συνέδριο ε, και σήμερα έχω έρθει με κάτι τελείως διαφορετικό. Αισθάνομαι λοιπόν πολύ καλά. Δεν έχουμε τελειώσει. Χρειάζεται περισσότερη απλούστευση. Γιατί αυτό που βλέπουμε φέτος είναι ότι η απλούστευση του Horizon 2020 έκανε τη διαφορά. Δηλαδή μία απλούς τύπος ε, είναι η καταποκοπή ε, για τις επιχορηγήσεις, η ηλεκτρονική ε, υπογραφή των συμβάσεων, η μία εφάπαξ πληρωμή, όλα αυτά φέραν τη διαφορά. Και θα συνεχίσουμε, θα συνεχίσουμε στο δρόμο της απλούστευσης. Και αυτό είναι ένα από τα θέματα τα οποία είναι σημαντικά. Τώρα, Μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ναι, κάνουν πολλά σφάλματα. Έχουν αυτή την τάση. Αλλά θα συμφωνήσω μαζί σας και έχουμε κάνει αυτή τη συζήτηση. Χρειαζόμαστε καινούριου ανθρώπου, καινούριε μικρομεσαίε. Δεν θέλουμε να δούμε τα χρήματα στου ίδιου και στου ίδιου. Αλλά είναι καινούργοι, δεν ξέρουν του κανόνε τόσο καλά όσο οι παλαιότεροι. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να συνεχίσουμε με έναν τρόπο που θα κατανοούν τους κανόνες, δηλαδή περισσότερη επικοινωνία, διαφορετικού είδους επικοινωνία, ε, εκστρατείες ενημέρωσης που στοχεύουν αυτές τις νέες ε, περιπτώσεις, γιατί τους θέλουμε και θέλουμε να εξασφαλίσουμε πως ξέρουν τους κανόνες. Επίσης, το ελεγκτικό συνέδριο συνιστά αυτές τις ε, ε, παρατηρήσεις που κάνουμε να τις κάνουμε και για την, εκ για την στρατηγική εκ των υστέρων ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό βέβαια δεν επηρεάζει το ποσοστό σφάλματος. Παρόλα αυτά, καλό είναι να αναλύονται τα συμπεράσματα και να αναλαμβάνονται τέτοιου είδους έλεγχοι και να συνεργαστούν περισσότερο με το ελεγκτικό συνέδριο εδώ. Τέλος, συνιστά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μοιράσει και να μοιραστεί τα αποτελέσματα της έρευνας. Και αυτό θα το κάνουμε και εμείς σίγουρα. Τέλος, χρειαζόμαστε τη δική σας βοήθεια για το μέλλον. Εμείς κάναμε ό,τι απλούστευση μπορούσαμε. Τώρα θα πρέπει να δούμε το Horizon Europe, θα είναι πια πιο εύκολη δομή, θα είναι ένα στοχευμένο εργαλείο με εταιρικέ σχέσεις, με μια mission-based προσέγγιση, δηλαδή ανα ε, συγκεκριμένη αποστολή. Και νομίζω ότι στα πέντε χρόνια ε, μπορώ να πω έκανα είναι κάτι το οποίο μπορούμε να συνεχίσουμε αν συνεργαστούμε όλοι μεταξύ μας έτσι ώστε να έχουμε πραγματικές επιπτώσεις στη ζωή των καθημερινών ανθρώπων αλλά και των ερευνητών. Ας συνεχίσουμε λοιπόν να συνεργαζόμαστε και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Thank you so much. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, πάρα πολύ καλή δουλειά σας. Τώρα όμως ε, πρέπει να κάνω κάποιες ερωτήσεις, ακόμα και αν είστε τελευταία φορά στην Επιτροπή Ελέγχου Προβλημών αλλά ήταν πάρα πολύ ευχάριστο που αναφέρετε τα συναισθήματα σας όταν η Μαρτίνα έκανε ερωτήσεις και με τότε ποσοστό σφάλματος πάνω από 15%. Έχω λοιπόν κάποιες ερωτήσεις και πρώτα απ' όλα μία παράκληση. Η πρώτη μου παράκληση αφορά το ότι ζητήσαμε να μας καταθέσετε ένα κατάλογο όλων των μελετών που έχουν ανατεθεί και έχουν δημοσιευτεί ή και όχι. Ε, δεν πρέπει να το κάνετε τώρα, αλλά το έχουμε ζητήσει. Το δεύτερο, οι επιπρόσθετες διαδικασίες ελέγχου, single audit approach. Αυτές οι διαδικασίες του ελεγκτικού συναδρίου σε κάποια, κάποιους φακέλους ε, διαπίστωσαν ελλείψεις σε τεκμηρίωση δειγματοληπτικούς ελέγχους και κατάθεση εκθέσεων, όπως επίσης και στην ποιότητα των διαδικασιών ελέγχου. Και το ελεγκτικό συνέδριο είπε ότι τότε δεν μπορούσε να βασιστεί στη δουλειά που είχε ήδη γίνει. Γι' αυτό λοιπόν με ενδιαφέρει ε, το τι προτίθεται ε, να κάνει η Κομισιόν, τι μέτρα για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και για να βελτιωθεί η αξιοπιστία της δουλειάς των άμεσα θυγόμενων εθνικών αρχών και επίσης και πώς μπορεί να βελτιωθεί η δυνατότητα να έχουν και να διασφαλίζουν ε, σωστούς ελέγχους με βάση τα διεθνή πρότυπα. Πώς είναι δυνατόν να βελτιωθεί λοιπόν αυτή η δυνατότητα των δημόσιων αρχών. Και μετά και ένα άλλο ερώτημα που αφορά καταρχήν στις μεγαλύτερες προκλήσεις και κατά πόσον υπάρχουν χώρες που δημιουργούν περισσότερα προβλήματα, μήπως ε, στα κράτη-μέλη υπάρχουν ε, κάποια θέματα ε, που προβάλλονται πολύ περισσότερο και αν ποια είναι ακριβώς αυτά. Δεύτερο ερώτημα, η δουλειά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η συμβουλευτική σε αυτά τα εθνικά σημεία επαφής είναι πολύ σημαντικό πώς να χορηγούν τις συμβουλές η ε, πρώτη τι ε, υποβάλλονται σε αιτήσει ε, θα πρέπει να έχουν καλή, καλές συμβουλές. Και είπε ο κύριος Επίτροπος ότι δεν θέλουν να έχουν πάντα τους ίδιους υποψήφιους, αλλά να υπάρχουν και νέοι ε, που υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά, αλλά συνήθως αυτοί είναι και εκείνοι που κάνουν τα περισσότερα λάθη. Γι' αυτό λοιπόν ερωτώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι ακριβώς προτείνει έτσι ώστε να βελτιωθεί η συμβουλευτική ικανότητα των εθνικών σημείων επαφής και να μας πείτε επίση ποια είναι κατά την άποψή σας τα περισσότερα προβλήματα σε σχέση με αυτά τα εθνικά σημεία επαφής. Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη και ε, σε σχέση με την αποδοχή της, ε, του όγκου της ε, παροχή συμβουλών, γιατί αυτό που παίζει ρόλο είναι κατά πόσον ένας ετών ε, γνωρίζει ότι υπάρχουν αυτά τα εθνικά σημεία επαφής. Αυτά τα σημεία επαφής είναι σωστά μοιρασμένα σε μια επικράτεια, έχουν τους απαραίτητους εμπειρογνώμονες και κατά την άποψή σας ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα οποτεδήποτε θέμα παροχής συμβουλών. Και επίσης, ε, τι ρόλο θέλει να παίζει η Επιτροπή έτσι ώστε αυτές τις ε, συμβουλές να τις βελτιώσει έναντι των ε, εθνικών σημείων επαφής, έτσι ώστε όλοι να μπορούν να παρουσιάζουν υψηλή ποιότητα. Ε, μετά υπάρχει ένα θέμα που, υπάρχει, που έχει σχέση με τα widening measures της συμμετοχής. Αυτό είναι ένα μέτρο για την προαγωγή των κρατών μελών ε, χωρίς πανεπιστήμια αριστείας. Τι ακριβώς είναι αυτό. Ε, δεν χρειάζεται να μας τα πείτε όλα προφορικά, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει να γνωρίζουμε είναι τι ακριβώς κάνει η Επιτροπή για να πείσει τα κράτη-μέλη τα οποία δεν έχουν καθόλου πανεπιστήμια αριστείας. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στο ίδιο το κράτος μέλος. Ίσως γιατί τον ενδιαφέρει, δεν έχουν χρήματα ή δεν έχουν το απαραίτητο προσωπικό. Ποια είναι τα βασικά αίτια και τι ακριβώς μπορεί να κάνει η Επιτροπή έτσι ώστε να μεριμνήσει, ε, να γνωρίζει ε, τι ακριβώς συμβαίνουν με τα μέτρα, το twinning, tinning, ε, ευρωπαϊκή συνεργασία και επιστήμη και τεχνολογία, ε, πώς μπορεί ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προάγει τα πανεπιστήμια αριστείας και την έρευνα αριστείας σε όλα τα κράτη-μέλη. Επίσης, μπορείτε να μας πείτε κατά πόσον τα μέτρα τα οποία έχετε λάβει έχουν οδηγήσει σε ιστορίες επιτυχίας ή μήπως έχετε κάποιες ενδείξεις ότι θα υπάρχουν τέτοιες επιτυχημένες περιπτώσεις στο μέλλον. Κατόπιν το Horizon Europe. Στο μέλλον ε, το 35% των κονδυλίων θα διατίθεται για το κλίμα. Και ε, αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή γίνεται δουλειά για τη μέθοδο. Και διαπιστώσαμε στον προπολογισμό ότι κάποια μέτρα όπως νανοτεχνολογία, βιοτεχνολογία, στη μέθοδο βρίσκονται στο 0%. Ενώ σε άλλες περιπτώσεις έχουμε το 100% ε, και όπου, εντάξει δεν είμαι σίγουρη αν είναι το 100% ή αν είναι μόνο το 80%. Κατά την άποψή σα όσον αφορά τη μέθοδο, τι ακριβώ θα αλλάξει και δεύτερον, ε, ποια είναι ε, τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να ληφθούν ε, για να επιτευχθεί το 35% για πράσινες τεχνολογίες ή για σχετικά μέτρα στην επιστήμη, την έρευνα, έτσι ώστε ή δυνατόν να υπάρξουν νέα προγράμματα. Και τέλος και μία τελευταία ερώτηση που αφορά στα μεγάλα έργα υποδομών η Γενική Διεύθυνση ε, προτίθεται ε, την εξάντε, τον εξάντε έλεγχο για μεγάλα προγράμματα υποδομής ε, κατά το επόμενο χρονικό διάστημα αυτά τα προβλήματα να αντιμετωπίσει με καινοτόμε μεθόδους. Αυτό το καινοτόμε δεν το κατανοώ ακριβώς. Τι ακριβώς σημαίνει καινοτόμες μέθοδοι ελέγχου και πώς ακριβώς διαχωρίζονται αυτές οι καινοτόμες μέθοδοι από τις παλιές. Αν ε, δεν μπορείτε να απαντήσετε σήμερα προφορικά για κάτι από όλα αυτά που ερώτησα, μπορείτε να απαντήσετε ε, εκ των υστέρων σε γραπτή μορφή. Παρακαλώ κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. για ε, όλες αυτές τις εξαντλητικές ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να ε, τις απαντήσω και όσες δεν μπορέσω γραπτός. Για τις μελέτες πρώτα απ' όλα και τον κατάλογο των μελετών, μόλις ε, ζήτησα ε, από το Γενικό Διευθυντή να βεβαιωθεί ότι έχουμε όλες τις απαντήσεις για τις μελέτες που αναθέσαμε και πληρώσαμε ως Γενική Διεύθυνση. Ποιες είναι, πόσες είναι. Μπορεί να μην έχετε ακόμη πλήρη απάντηση, αλλά θα σας διαβιβαστεί γραπτός και θα το αναλάβω εγώ προσωπικά να γίνει και οι υπηρεσίες ε, το επιτελείο του Γενικού Διευθυντού. Ε, κάνατε μια δύσκολη ερώτηση σχετικά με το τι μπορούμε να κάνουμε για να ε, έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις ε, για πραγματική αξιοπιστία των εθνικών ελεγκτικών αρχών. Όταν ανέλαβα νόμιζα ότι θα μπορούσα με ένα μαγικό ραβδάκι να τα αλλάξω όλα. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε. Αλλά τι έμαθα. Δύο τρόποι υπάρχουν. Πρώτον, να επενδύσουν περισσότερο σε εθνικό επίπεδο για την ε, ενημέρωση και το δεύτερο είναι η απλούστευση. Και σε αυτή την πενταετία στην αρχή ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα γιατί οι περισσότερες ε, συναλλαγές που έψαχνε ε, το ελεκτικό συνέδριο ήταν από το πρόγραμμα πλαίσιο πέντε για την έρευνα. Αλλάξαμε λοιπόν έκτοτε. Ε, είναι σφάλματα. Πραγματικά κάτι κάνει λάθος ο κόσμος. Δεν προσπαθεί να εξαπατήσει κανέναν. Δεν είναι σκεμμένο. Είναι γνήσια λάθη. Σφάλματα. Ε, δεν τήρησαν το χρονοδιάγραμμα ή δεν ξέρω το έμεσο κόστος το ανέφεραν με τρόπο λανθασμένο. Ε, αποφασίσαμε λοιπόν να κάνουμε ε, μια απλούστευση με ένα καταποκοπή ποσό για τα έμεσα κόστη και αυτό έλυσε αυτόματα πάρα πολλά προβλήματα. Θα σας έστελα λοιπόν αυτό το μήνυμα της συναδέλφου Μαρία Γκαμπριέλ ότι η απλούστευση είναι κάτι το οποίο είναι διαρκές, δεν μπορεί να το σταματήσει. Θα πρέπει τώρα να δώσει συνέχεια σε αυτό. Αλλά δεν μπορείς να αλλάξεις και τα πάντα, γιατί αν αλλάξεις τα πάντα δεν απλουστεύεις. Ε, προφανώς, χρειάζεται προσοχή εδώ. Θα έλεγα λοιπόν επικοινωνία σε εθνικό επίπεδο. Κάναμε πολλά προς αυτή την κατεύθυνση. Και επικοινωνία τι εννοώ. Όχι από εμά, αλλά και μεταξύ των χρηστών. Οι εταιρείε, τα πανεπιστήμια ε, μπορούν να μας διδάξουν ε, οι ίδιοι πώς κάνουν κάποια πράγματα. Για τα διάφορα κράτη-μέλη τώρα, πιστεύω ότι στατιστικά και θα επανέλθω με περισσότερες πληροφορίες. Το Horizon 2020 ε, αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για τις χώρες που γνωρίζουμε, που έχουν τα μεγάλα ερευνητικά κέντρα, κέντρα καινοτομία, όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Ισπανία, η Γαλλία κτλ. Ε, οι περισσότερες λοιπόν συναλλαγές είναι σε αυτές τις χώρες και υπάρχουν και άλλες ε, χώρες ε, με λιγότερες συναλλαγές, εξού και τα δείγματα. Πάντως, για να είμαι ειλικρινής, δεν πιστεύω ότι σήμερα θα βλέπαμε μεγάλες αλλαγές. Όχι μεταξύ των κρατών, αλλά μεταξύ των ιδρυμάτων. Δηλαδή, αν, αν είσαι στην Ισπανία ή στην Πορτογαλία ή στη Μάλτα ή στην Κύπρο, ε, πανεπιστήμιο, ε, ε, αριστείας, ξέρεις πώς γινόνται αυτά τα πράγματα, αλλά όταν είσαι πιο περιφερειακό πανεπιστήμιο, ένα πανεπιστήμιο που πρώτη φορά συμμετέχει στα προγράμματά μας, ε, είναι μεγαλύτερες δυσκολίε, Γιατί προφανώς όταν ασχολείσαι με κάτι για πρώτη φορά, το ίδιο ισχύει με τι εταιρείε. Αυτό δεν έχει τόσο πολύ περιφερειακό χαρακτήρα, αλλά έχει να κάνει με το επίπεδο τη εταιρεία ή του πανεπιστημίου στα πλαίσια ε, του πεδίου εφαρμογή των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Επίσης, μας ε, ρωτήσατε για τη διεύρυνση και θέλω να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο στους τριμερείς διαλόγους, όπως ξέρετε, είχαμε αυτή την ιδέα στην πρότασή μας να διευρύνουμε, να διπλασιάσουμε ε, τα χρήματα που κατευθύνονται εκεί και το Κοινοβούλιο μας βοήθησε στον τριμερή διάλογο γιατί επίεσε το Συμβούλιο προς την κατεύθυνση αυτή και τώρα έχουμε προσημειώσει αυτό το 3% του όποιου προϋπολογισμού προκύψει ε, και αυτό είναι κάτι το οποίο απολυτελεί και μεγάλη αλλαγή στο μέλλον. Δεν βλέπω την πρώην συνάδελφο Κορίνα Κρέτσου, που ξέρω ότι είναι μέλος της Επιτροπής σας. Έχουμε συνεργαστεί πολύ σε αυτά τα θέματα για τις συνέργειες μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων και του Horizon 2020. Και νομίζω ότι εκεί είναι το μέλλον. Πώς θα έχουμε περισσότερες συνέργειες ε, ε, η σφραγίδα αριστείας είναι ένα θαυμάσιο παράδειγμα και η κυρία Κρέτσου και εγώ ε, χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Μετά μου κάνατε μια ερώτηση, δεν έχω την πλήρη απάντηση σε αυτή, γιατί σε κάποιους τομείς, κλάδους όπως είναι η βιοτεχνολογία, έχουμε λιγότερα κονδύλια και κάπου αλλού περισσότερα. Ξέρετε τι αλλάξαμε αυτή τη στιγμή για το Horizon Ευρώπη, το διάδοχο πρόγραμμα. Ε, ότι ε, γενικά είχαμε μια προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω στο 5ο, 6ο, 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και το Horizon 2020. Έχουμε ομάδες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αποφασίζουμε τελικά που θα δοθούν τα κονδύλια. Ενώ τώρα η μεγάλη διαφορά με το διάδοχο πρόγραμμα, το Horizon Europe, είναι τελείως διαφορετικό. Είναι μια συμπαραγωγή καθόμαστε μαζί με τους ε, ε, ενδιαφερομένους, εμπλεκομένους ε, και το συζητούμε, όχι μόνο επειδή το ζητούν οι ίδιοι, μαζί με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε κάθε ένα από τους τομείς θα έχουμε έναν αρμόδιο. Σήμερα μπορείτε να έχετε τρεις ή τέσσερις γενικές διευθύνσεις που είναι αρμόδιες και θα πρέπει να συνεννοηθούν πρώτα-πρώτα μεταξύ τους. Αυτό το λέμε συμ... δημιουργία ή συμπαραγωγή και θα είναι κάτι που θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη συνέπεια και συνοχή στη μεθοδολογία. Με ρωτήσετε και κάτι που δεν ξέρω να σας απαντήσω για την καινοτόμο, τον καινοτόμο λογιστικό έλεγχο. Τι είναι αυτό. Λυπάμαι πάρα πολύ. Θα πρέπει να μάθω κι εγώ τι είναι για να σας απαντήσω. Τι εννοούν μάλλον οι υπηρεσίες. ότι επικοινωνούμε καλύτερα, ότι θα έχουμε περισσότερους επιτόπου, θα προσπαθήσουμε να ενημερώσουμε, να εκπαιδεύσουμε τις εταιρείες, ιδιαίτερα ε, ε, για τον εξωτερικό έλεγχο, αυτό που κάνουν οι ιδιωτικές εταιρείες, ε, το λογιστικό έλεγχο, να εργαζόμαστε περισσότερο μεταξύ τους και για την απόδοση τους. Και μία από τις συζητήσεις που έχουμε εκεί με το ελεκτικό συνέδριο είναι ακριβώς αυτό το θέμα της απόδοσης. Εκεί είναι η καινοτομία. Μπορεί να έχω μηδενικό δείκτη φάλματος, αλλά δεν ξέρω αν ο Σερ Πίτερ Ράτκλιφ που πήρε το Νόμπελ ε, ε, ε, έκανε λάθη συμπληρώνοντας το έντυπο της αίτησης, πάντως το Νόμπελ το πήρε. Σίγουρα θα πρέπει να γίνονται τα πράγματα σωστά, αλλά να δούμε και τι κάνουμε, όχι μόνο πώς το κάνουμε. Ε, ίσως από εκεί προκύπτει η λέξη καινοτόμος. Θα το ψάξουμε και θα σας πούμε. So, thank you very much for the first... Σας ευχαριστώ πολύ για τις πρώτες απαντήσεις. Θα δούμε λοιπόν ε, αυτά τα καινούρια και πολύ καινοτόμα μέτρα. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Πένκοβα από τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ επίσης και τον κύριο Κοσλόφ που Παρουσία στην έκθεση και τον Επίτροπο Μόιδας που απάντησε στις δικές μας ερωτήσεις. Έχω να ρωτήσω τα εξής που ξεπερνούν τα γραπτά σχόλια που μας έχετε στείλει. Θα σας εξηγήσω λοιπόν. Η πρώτη ερώτηση και η δεύτερη σχετίζονται με την απάντηση 81 μπορείτε να μας δώσετε πληροφορίες για το ποσοστό ε, σφάλματος σε σχέση με, τα, με τη δέσμευση κονδυλίων που, έχει, που έχουν αναλυφθεί, με τις μέσεις που έχουν αναλυφθεί. Αυτό για το Horizon 2020. Και το δεύτερο που είναι παρόμοιο, ποσοστό εκτέλεσης παρακαλώ, δηλαδή που να έχει πληρωθεί στους τελικούς αποδέκτες το, για το Horizon 2020 από το 2018 και μέχρι σήμερα. Επίσης, η μέθοδος και τα βήματα για να μειώσετε τη μεγάλη γεωγραφική έλλειψη ισορροπίας για να στηρίξετε και τους ερευνητές στα πλαίσια του Horizon 2020 με αριθμό ερευνητών από κάθε κράτος μέλος. Θα σας δώσω κάποια παραδείγματα για να καταλάβετε γιατί σας ρωτάω. Είναι η ερώτηση 82. Από το Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε στηρίξει πάνω από χίλιους ερευνητές από τη Γερμανία, πάνω από 800, από το Βέλγιο σχεδόν 200 και μετά έχουμε χώρες όπως η Ελλάδα, 27, Βουλγαρία ένας, Σλοβακία ένας. Θέλω λοιπόν να καταλάβω αν υπάρχουν κάποια βήματα ή σχέδια για να ξεπεράσετε αυτή την έλλειψη ισορροπίας, γιατί δεν μοιάζει να είναι η κατάλληλη αυτή τη στιγμή. Εξαιρετικές ερωτήσεις. Να πω πρώτα απ' όλα πως για την ερώτηση 81 θα σας στείλω αν έχετε ερωτήσεις ε, τις ε, πληρωμές που έχουν εκτελεστεί έχετε τον πίνακα στις απαντήσεις που λέει 2014 1,3 δις 5,1 στο 15 και τα λοιπά το 18 όπου φτάνουν τα 31 και κάτι δις. Στην σελίδα 39 των απαντήσεων έχετε τις πληρωμές που έχουν εκτελεστεί, δηλαδή αυτές οι οποίες φτάνουν στον τελικό αποδέκτη. Μετά, διαβάζοντας αυτό που ρωτούσατε, την ερώτηση 82, είπατε η Κομισιόν λέει ότι από το 4 μέχρι το 18, 5.250 ε, κορυφαίοι ερευνητές έχουν χρηματοδοτηθεί μέσω του Horizon 2020 δώστε μας πληροφορίες από ποιες χώρες. Εδώ θα ζητήσω από την υπηρεσία να ξαναδεί τον πίνακα, γιατί νομίζω ότι είναι αδύνατον στη Βουλγαρία να είχαμε ένα άτομο. Νομίζω αυτό είναι μόνο το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας. Η απάντηση που δόθηκε και αυτή τη στιγμή αντιδρώ εν θερμό και γι' αυτό το λέω έτσι ανοιχτά, θεωρώ πως εδώ αναφερόμαστε μόνο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνα ή στο Horizon 2020. πολύ ψηλότερα τα νούμερα. Για τη Βουλγαρία τα γνωρίζω καλά. Και νομίζω το ίδιο συμβαίνει και με άλλες χώρες. Και θα σας πω γιατί είναι αυτό το Ευρωπαϊκό ε, Συμβούλιο Έρευνας. Γιατί για την Πορτογαλία που την γνωρίζω καλύτερα από οτιδήποτε άλλο, ε, ε, είναι αυτά ακριβώς τα νούμερα. Οπότε θα σας στείλουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά. Για τη διεύρυνση θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο έτσι ώστε οι προτάσεις μας για να υπάρχει συνέργεια με τα διαφορετικά ταμεία να λειτουργήσει, να λειτουργήσουν. Η πρόεδρος το γνωρίζει εδώ και 4-5 χρόνια. Λέμε πως θέλουμε να εργαστούμε περισσότερο με και μέσω των διαφορετικών ταμείων. Αυτό που κάναμε τότε με την ε, Κορίνα Κρέτσου, να δημιουργήσουμε μια σφραγίδα που θα λέει άριστο ε, project και μετά ε, επειδή υπάρχουν υπογραφές δύο επιτρόπων να ξαναμπαίνουν στην αξιολόγηση και τελικά να μην γίνεται τίποτα. Οπότε μία από τι προτάσει που κάναμε ήταν να έχουμε μια πιο αυτοματοποιημένη διαδικασία όπου κάποιο ο οποίο έχει περάσει από αυτά τα φίλτρα του Horizon 2020 να μπορεί να απευθυνθεί στα εθνικά ταμεία ή στα ε, ε, διαρθωτικά ταμεία ή σε κάποια άλλα ταμεία και να μπορεί να χρηματοδοτηθεί αμέσω. Αλλά εκεί θα ζητήσω τη βοήθειά σα στο μέλλον. Πάντως θέλουμε πραγματικά να διευρύνουμε ένα σημαντικό κομμάτι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Επίτροπε. Η Ματίνα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Καταρχήν ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δουλειά που κάνατε τα τελευταία πέντε χρόνια. Σας ευχαριστούμε για τις ε, διεξοδικές απαντήσεις σας και χαίρομαι πάρα πολύ που ε, τα τελευταία πέντε χρόνια μαζί αλλάξαμε το θέμα των αποδόσεων, την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, ακόμα και αν ακόμα υπολείπονται αρκετά. Ε, ίσως θα ήταν καλό να ακούσουμε από εσάς προτάσεις για το τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα ως Επιτροπή. Να μην μιλάμε μόνο για τα ποσοστά ασφάλματος, αλλά να δούμε και θετικά παραδείγματα, να είμαστε πιο θετικοί έναντα της έρευνας και της καινοτομίας. Φοβάμαι ότι αυτό είναι ένας πολύ δύσκολος τομέας για να παρουσιάσει κανείς συγκεκριμένα παραδείγματα. Η έρευνα είναι μια μακρά διαδικασία, άρα δηλαδή θα ήταν ενδιαφέρον να μας πείτε ε, τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε τα επόμενα πέντε χρόνια σε αυτή την Επιτροπή. Ίσως αυτή να είναι η τελευταία σας παρουσία εδώ στην Επιτροπή και, και λυπάμαι ε, πολύ Γι' αυτό φιλοσοφικές λοιπόν ερωτήσεις μου. Πρώτον, ε, τι γίνεται ακριβώς με την ε, ε, απόδοση, πώς μπορούμε να πείσουμε καλύτερα τους Ευρωπαίους πολίτες για το τι ακριβώς κάνουμε. Να επενδύσουν στην έρευνα και την καινοτομία. Ο κύριος Μπίνιγκμαϊρ, είχαμε σήμερα την ανανέωση, την ανανέωση της θητείας πολλών υποψηφίων, ο κ. Μπίνιγκμαϊρ είπε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Η απόδοση πρέπει να είναι το αποτέλεσμα του διαλόγου. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί η κατουσία εννοούσε ότι πρέπει να υπάρχουν κάποιες πρώτες εξηγήσει για το τι ακριβώς προτίθεται να κάνει η Επιτροπή με την χρηματοδότηση και μόνο αν έχει κανείς ε, το στόχο, μόνο μετά μπορεί να αξιολογήσει την απόδοση και αυτό είναι λογικό. Όμως κάτι λείπει σε αυτό το διάλογο, γιατί μερικές φορές με βάση τα αποτελέσματα των, του Λεκτικού συνεδρίου, ε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, και όσοι πρωτοκάνουν αίτηση, αυτοί είναι και εκείνοι που κάνουν τα περισσότερα λάθη, τα σφάλματα. Άρα δηλαδή Υπάρχουν ακόμα αρκετά που μπορούν να γίνουν σε αυτό το διάλογο ανάμεσα στους δικαιούχους, τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώς μπορούμε όλα αυτά να τα λύσουμε για να έχουμε καλύτερη απόδοση. Η δεύτερη ερώτησή μου έχει σχέση με την πρώτη. Δηλαδή, για να επιτύχουμε απόδοση χρειαζόμαστε την κατάλληλη χρηματοδότηση. Εσείς τι πιστεύετε για τις περικοπές στο επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και στο επόμενο πρόγραμμα Horizon. Αυτός ο στρατηγικός σχεδιασμός πώς μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά τις συνεργασίες και τις εταιρικές σχέσεις. Και τελευταία μου ερώτηση, όταν μιλάμε για έρευνα και καινοτομία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μερικές φορές ξεχνάμε ότι δεν πρόκειται μόνο για ευρωπαϊκά κονδύλια. Γνωρίζουμε ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια είναι μόνο ένα μικρό κομμάτι ε, γενικότερα της χρηματοδότησης για την έρευνα και την καινοτομία στην Ευρώπη. Ε, όταν μιλάμε για τη χρηματοδότηση του Horizon Europe, μιλάμε για 8 μέχρι 10% του συνόλου των κονδυλίων για την έρευνα και την καινοτομία στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τα επόμενα έτη. Άρα δηλαδή πρέπει να γίνουν περισσότερες εθνικές επενδύσεις. Τι πρέπει να κάνουμε ως Κοινοβούλιο και Επιτροπή έτσι ώστε να δώσουμε κίνητρα στα κράτη-μέλη να επενδύουν περισσότερο στην έρευνα και την καινοτομία. Ε, πώς μπορούμε να φέρουμε τα κράτη τη μελη σε αυτό το 3% που είναι ο στόχος 3% του ΑΕΠ, που είναι ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λυπάμαι ε, που ήταν φιλοσοφικής φύσεως η ερωτήση μου, αλλά νομίζω ότι μετά από αυτά τα πέντε χρόνια ε, μπορείτε να δώσετε απαντήσεις. Δεν ήταν μόνο φιλοσοφική, λέει η Πρόεδρος. Ε, Πίτρο, σε ευχαριστώ, Πρόεδρε και αξιότιμα μέλη. Σε ευχαριστώ, Μαρτίνα, για τις ερωτήσεις. Έτσι είναι πάντα προκλητικές ε, ερωτήσεις με την έννοια ότι με προκαλούν να σκεφτώ και να απαντήσω. Τι κάνουμε για την επιτροπή σας και τα λοιπά. Τι, μάλλον εσείς τι μπορείτε να κάνετε για μας. Κοιτάξτε. Καμιά φορά μπορείτε να προσκαλείτε εδώ στην επιτροπή σας και κανέναν επιστήμονα ή κανέναν καινοτόμο για να σας λέω από πρώτο χέρι τι γίνεται. Ξέρω ότι είναι θέμα χρόνου και πώς θα το αξιοποιείτε το χρόνο σας, αλλά σκεφτείτε το γι' αυτό. Ο Μπεν Φερίγκα μένει εδώ κοντά στην Ολλανδία, ε, ο νομπελίστας. Ε, αγαπάει την Ευρώπη και είπε ότι δεν θα έπαιρνα τον Νόμπελ αν δεν είχα πάρει κονδύλια από την Ευρώπη προηγουμένως. Ε, και θα χαρεί πολύ να ε, έρθει εδώ και είναι καλό να έχετε επαφές με επιστήμονες. Καλέστε το σε μια δεξίωση για τα Χριστούγεννα. Δεν χρειάζεται να είναι ολόκληρη συνεδρίαση επίσημη. Ε, και καλό θα ήταν, νομίζω καλή ιδέα, αν έχετε χρόνο, καμιά φορά να βλέπετε και επιστήμονες αυτού και αυτούς τους νέους ε, επιχειρηματίες. Γιατί σκέφτομαι και τον Μπόιαν Σλάτ, έναν άλλο νεαρό Ολλανδό, που έφυγε από το Πανεπιστήμιο για να πάει να καθαρίσει του ωκεανού. Και έχει ε, φτιάξει αυτή την εταιρεία που λέγεται ε, Oceans Cleanup. Και για όλους εμάς ε, είναι πολύ σημαντικό και έρχομαι στο επόμενο. Τι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο για να έχουμε περισσότερη επαφή με τους πολίτες. Ξέρετε, ότι κάτι το οποίο είχα σκεφτεί στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ε, επιστήμη που να βασίζεται, ε, να εμπνέεται από μία αποστολή. Δηλαδή, έχετε πέντε τομείς εσείς για αποστολές της επιστήμης. Αυτή είναι η ε, δυνατότητα να συνδέεστε με τους πολίτες. Και η εκλεγμένη πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής μίλησε για τον καρκίνο. Έχουμε μια αποστολή για τον καρκίνο, αλλά δεν αρκεί αυτό. Θα πρέπει και ο κόσμος να καταλαβαίνει τι κάνετε για τον καρκίνο. Γιατί αν πούμε ότι ψάχνουμε τον καρκίνο, ωραία. Και από εκεί και πέρα ο κόσμος πώς θα ε, αισθανθεί ότι τον αφορά. Για να καταλάβει ο πολίτης ότι η Ευρώπη κάνει κάτι γι' αυτόν. Αν δείτε λοιπόν αυτές τις αποστολές, είπαμε, ξέρω εγώ, οι δέκα πρώτες πόλεις στην Ευρώπη που θα έχουν φύγει τελείως από τον άνθρακα. Ο κόσμος θα το καταλάβει. Χρειάζεται λοιπόν αυτή η σύνδεση επικοινωνιακά με τους πολίτες. Ή να πούμε, σε δέκα χρόνια από τώρα δεν θα πεθαίνει κανείς από καρκίνο. Ξέρουμε ότι τον καρκίνο δεν μπορούμε να τον θεραπεύσουμε. Αλλά τουλάχιστον να μην πεθαίνει κάποιος από καρκίνο. Δεν ξέρω, μπορεί να μην είναι σε 10 χρόνια, να είναι σε 5 και σε 20. Αλλά ο κόσμος αυτό θα το καταλάβει. Έτσι συνδεόμαστε με τους πολίτες και αυτές είναι οι αποστολές ε, και τα εργαλεία που έχετε στη διάθεσή σας για να αγωνιστείτε. Μιλήσατε για τους ε, νέους, νέους ερχόμενους στο σύστημα. Εδώ υπάρχει μια αντίφαση. Θέλουμε νέους να μπαίνουν ε, στις επιδοτήσεις, ε, ξέρουμε ότι κάνουν περισσότερα σφάλματα. Ε, ας το καταλάβουμε αυτό, ας το ομολογήσουμε, ε, τους θέλουμε. Και θα πρέπει να έχουμε περισσότερες δυνατότητες επικοινωνίας, εργαστήρια, σεμινάρια, πώς θα συμπληρώνουν τα έντυπα και πώς λειτουργούν οι διαδικασίες. Το βασικό είναι ότι είμαστε σταγόνα στον ωκεανό από αυτά που είπατε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΑΕΠ της δηλαδή, είναι 14-3. 2% δίνουμε ε, συνολικά στην έρευνα και την ανάπτυξη. 280 δις είναι αυτά συνολικά. Τα μισά είναι ιδιωτικά κονδύλια, 140 δις καινοτομίας και επιστήμης. Τα υπόλοιπα 140 είναι από τις χώρες μέλη. 140 δις ετησίως είναι το σύνολο αλλά του προϋπολογισμού. Αν διαιρέσεις τα 80 εκατομμύρια διεπτά είναι 10 δις το χρόνο από τον ορίζοντα. Δηλαδή από τα 140 βρισκόμαστε στα 10 δις ετησίως. Έχετε απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβουμε γιατί γίνονται αυτές οι συζητήσεις σε πολλές χώρες για το PDP, ότι κανένας δεν θέλει να βάλει ένα ευρώ παραπάνω. Γι' αυτό είναι το πρόβλημα. Νομίζω, ελπίζω να απάντησα λίγο στις ερωτήσεις σας. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Βιόλα Φων Κάρμα. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Σας ευχαριστώ και εσάς και την ομάδα σας για μια πραγματικά πολύ εμπεριστατωμένη δουλειά. Θα ήθελα να μου δωσετε λίγη, λίγο follow-up σε σχέση με τα όσα είπε η κυρία Χολμάγερ. Ναι, όχι μόνο την ποσότητα των μελετών, αλλά και τους τίτλους και ίσως και τους λόγους για τους οποίους δεν έχουν δημοσιευθεί. Γιατί νομίζω ότι εκεί είναι κάπως περίπλοκο το ζήτημα. Θα ήθελα λοιπόν να έχω μια γενικότερη εικόνα. Είστε... Έχετε δίκιο. Πήγαμε στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Τεχνολογία και την Καινοτομία, το επισκεφθήκαμε και πολύ σωστά είπατε κι εσείς αυτοί οι νέοι ερευνητέ είναι το μέλλον μας και θα πρέπει να μείνουν στη θέση τους, να χρηματοδοτούνται περισσότερο. Επίσης να είμαστε πιο φιλικοί προς την ε, ε, χρηματοδότηση ακόμα και σε project τα οποία έχουν πολλούς κινδύνους σε συνδυασμό με νεοφυείς επιχειρήσεις, με μικράς ε, ε, επιχειρήσεις και με ενδιαφέρει πολύ το μοντέλο χρηματοδότηση που θα ακολουθήσουμε γιατί στο συγκεκριμένο ίδρυμα λέει μέχρι 25% της έρευνας θα χρηματοδοτείται είτε από το Horizon 2020 είτε από κάτι άλλο αλλά χρηματοδοτούνται και από άλλα ταμεία. Θα ήθελα να μου πείτε λοιπόν πόσα λαμβάνουν από άλλες ευρωπαϊκές πηγές, ταμεία, προγράμματα, για να δούμε την ανταγωνιστικότητα, τη βιωσιμότητα του Ιδρύματος, για να δούμε πώς τα χρησιμοποιούν για να μοχλεύσουν από τη βιομηχανία, άλλες επενδύσεις και επίσης με εξέπληξε το γεγονός πως οι ερωτήσεις που υποβάλλω κρίνονται πλέον απόρριτες. Έχω στείλει ερωτήσεις όχι μόνο σε μία επιχείρηση ή για μία επιχείρηση, αλλά τα κοιτάμε τους εταίρους μας από τρίτες χώρες, θα ήθελα να πείτε ποιες είναι οι ασφαλιστικές δικλείδες που έχετε συμπεριλάβει στις συμβάσεις των ερευνητών με τρίτους χώρες έτσι ώστε να μην γίνει κατάχρηση ή βιομηχανική εκμετάλλευση εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί για την εταιρεία που σας έγραψα και ίσως για κάποιες άλλες η ανησυχία μου είναι πως χρειαστούν κάποιες βελτιώσεις για το επόμενο πρόγραμμα. Αν έχετε κάνει οτιδήποτε έκτοτε μια και ίσως κάποιες χώρες να... και κάποια ερευνητικά κέντρα να χρησιμοποιήσαν με ασφαλμένο τρόπο ή να καταχράστηκαν αυτή τη χρηματοδότηση ενώντας, μεταφέροντας ε, εκτός. Ε, ο Επίτροπος. Θα ήθελα να σας πω ότι θα σας στείλω όλες τις πληροφορίες σε γραπτή μορφή. Έχετε βεβαίως το δικαίωμα να μάθετε τα πάντα για τις μελέτες. Δεν έχω τίποτα να κρύψω από αυτού. Απλά δεν τα έχω μαζί μου, δεν έχω τις πληροφορίες. Όμως θα δώσω εντολή στην ομάδα μου να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις. Θα σας δείξουν όλες τις μελέτες, γιατί υπάρχουν, για ποιο λόγο. Όσον αφορά το ε, η δεν είναι σήμερα υπό την ευθύνη μου. Όπως ξέρετε υπάγεται ε, στον ε, συνάδελφο που είναι αρμόδιο την εκπαίδευση το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα της Τεχνολογίας. Εκεί υπάγεται, αλλά ένα από τα σημαντικότερα μέτρα το οποία ε, δεν αναφέρθηκε όμως από τον κυρία Ουρσουλα Φαντελένη είναι να δώσει την ε, Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας στον ίδιο Επίτροπο και αυτό ε, είναι σωστό. Έτσι λοιπόν, όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα της Τεχνολογίας, θα σας στείλω τα στοιχεία με όλους τους αριθμούς. Όμως πιστεύω ένα από τα πράγματα που πήγε πολύ καλά στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Τεχνολογίας είναι η κοινότητα ε, πληροφόρησης, το KICS ε, και εκεί υπάρχει μια ανάμιξη ε, του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και νομίζω ότι αυτό θα καταλαμβάνει ένα μεγάλο κομμάτι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας, αυτό που φτιάξαμε μαζί. Νομίζω στην καινούργια δομή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτό θα δουλέψει πάρα πολύ καλά και θα σας στείλω τα σχετικά στοιχεία. Όσον αφορά τώρα την εταιρεία που δεν αναφέρατε, στη γενικότερη ερώτησή σας, Νομίζω ότι ένα από τα θέματα που δεν κάναμε καλά και που εκεί πρέπει να βελτιωθούμε είναι ότι ναι πράγματι είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις χώρες του κόσμου αλλά χρειαζόμαστε αμοιβαιότητα ε, με όλες τις χώρες, ό,τι και αν είναι κάθε χώρα. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση της εταιρεία που αναφέρεται, ο αγώνας με τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν περισσότερο για να διασφαλίσω ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείε που βρίσκονται στην Κίνα μπορούν να απευθυνθούν και σε κιναζικά εθνικά κονδύλια και να τα λαμβάνουν. Ε, κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών επιτύχαμε μία συμφωνία επί χάρτου, αλλά η πραγματικότητα όμως ε, δεν είναι αυτή. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι ναι, Πρέπει όμως ε, πρώτα απ' όλα να διαφυλάξουμε την αμοιβαιότητα που δεν υπάρχει σήμερα. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι υπάρχει ένα γεγονός ότι είμαστε ανοιχτοί σε άλλες χώρες ε, και αυτή είναι μια γενικότερη απάντηση και Επίσης, ε, πάρα πολλές πληροφορίες που παίρνουμε από διάφορες χώρες που αφορούν στην επιστήμη, την τεχνολογία, ε, στον τρόπο με τον οποίο εργάζονται. Αυτά είναι πολύ θετικά για την Ευρώπη. Μπορούμε δηλαδή ε, να δούμε το θέμα από διαφορετική επίσης σκοπιά. Και όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα ε, και αυτά ε, υπάρχουν τέτοια θέματα με τις ευρωπαϊκές εταιρείες, διότι το δικό μου το σύνθημα ήταν να είμαστε πάντα σε ανοιχτό περιβάλλον. Εάν τα κονδύλια είναι δημόσια, οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν την πληροφορία για να επιτύχουν την καινοτομία. Άρα δηλαδή όταν οι άνθρωποι ε, παρισφρέουν στα, στις επιχορηγήσεις μας, θα πρέπει να μπορούν να δημοσιεύουν δημοσιεύουν ε, τα στοιχεία τους, ε, γιατί αυτό επιθυμούν να το γνωρίζουν και οι φορολογούμενοι. Και τα δεδομένα, τα στοιχεία να είναι επίσης δημοσιοποιήσιμα. Και μετά να μπορεί κανείς να πει ότι να, αυτή η ιδέα της εταιρεία πρέπει να προστατευτεί. Όμως ε, η επιλογή default ότι η εταιρεία ε, είτε έρχεται από την Κίνα είτε τις ΗΠΑ, πρέπει να εντάσσεται μέσα σε ένα ε, ανοιχτό σύστημα, γιατί έχει αποδειχτεί ότι η ανοιχτή καινοτομία δουλεύει καλύτερα από την κλειστή. Ακόμα και εάν υπάρχει ένα πορώδες σύστημα καλύτερο αυτό από το να είναι κλειστό. Το ένα είναι να ανοίξουν ε, και να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία και το άλλο είναι να προστατεύονται οι ιδέες. Εγώ πάντα έλεγα ανοιχτές, διαθέσιμες πληροφορίες, αλλά να προστατεύονται οι ιδέες. Γιατί αν δεν προστατεύονται οι ιδέες δεν θα υπάρχουν και επιχειρήσεις. Άρα δηλαδή ε, πρέπει να υπάρχει κάποια ισορροπία. Ε, τώρα, ε, ρήτρε και δικλείδες ασφαλείας έναντι τρίτων χωρών. Όλα αυτά θα πρέπει να υπάρχουν για να υπάρχει ασφάλεια, αλλά τις περισσότερες φορές δεν είναι καν απαραίτητα όλα αυτά, γιατί υπάρχει αμοιβαιότητα στην οποία αναφέρθηκα προηγουμένως. Συμφωνείτε? Καλώς. Ε, ο κύριος Κούς, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμε, κύριε Επίτροπε. Λυπάμαι που σας γυρίζω την πλάτη. Είμαι υποχρεωμένος. Αλλιώς δεν θα μπορέσω να μιλώ στο μικρόφωνο. Ε, μια ερώτηση έχω. Με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολούθησα αυτά που είπατε και τις ιστορίες σας και πολύ με εντυπωσίασαν αυτά και το θέμα το κάνετε και πιο προσιτό. Ε, έχω μια ερώτηση. Μιλήσατε για την απλούστευση, simplification και μας είπατε ότι θα μπορούσε αυτό να αποτελέσει μια λύση. Πώς θέλετε ακριβώς να το κάνετε αυτό. Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεσπίζει όλο και περισσότερους κανόνες και περιπλέκει τον κόσμο ακόμα χειρότερα για αυτά που θέλουμε εμείς να κάνουμε. Με όλο και περισσότερους κανόνες που στηβάζονται. Ε, πώς θέλετε εκεί να επιτύχετε την απλούστευση. Έχετε δίκιο. Ιδιαίτερα για την επιστήμη θα ήταν πάρα πολύ επιθυμητό αυτό ε, και καλό ήταν να το έχουμε ως ε, ε, προσδοκία και επιδίωξη, αλλά πώς θα το κάνετε αυτό. Πολύ συναρπαστική ερώτηση για τον Επίτροπο. Απάντηση. Όταν αρχίσαμε τη δουλειά μας το 2014, ε, μπήκαμε στο πρώτο κύμα της απλούστευσης, όπως το ονομάσαμε, που δεν ήταν ακριβώς το πρώτο, γιατί το πρώτο βήμα ήταν ε, το Horizon 2020. Όλο το πρόγραμμα ήταν πιο απλό. Σε αυτό το πρώτο κύμα, λοιπόν, τι θέλαμε να κάνουμε, να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο, γιατί ξέραμε το εξής, ότι... Υπάρχει κάτι που ξέρουμε. Όταν είναι περίπλοκοι οι κανόνες, πολλαπλασιάζονται και τα σφάλματα. Αυτό το λέει και η λογική και η πραγματικότητα. Και ανέκαθεν επέμενε το ελεκτικό συνέδριο στην απλούστευση των κανόνων. Από εκεί ξεκινήσαμε εμείς και είπαμε ας απλουστεύσουμε κάτι ε, που να είναι το εξή. Αν θέλετε επιδότηση, ε, δύο ε, συντελεστέ έχετε. 75% ή 100%. Αν είστε ερευνητής, αμυγής είναι 100%. Αν είστε μικρομεσαία επιχείρηση και τα λοιπά καινοτόμα, 75%. Ένα άλλο πρόβλημα που οδηγεί σε μεγάλη σύγχυση είναι το έμεσο κόστος. Υπάρχει το, τα, οι δαπάνες προσωπικού και το έμεσο κόστος. Δηλαδή, όταν πηγαίνεις σε ένα συνέδριο, ξέρω εγώ πρέπει να αγοράσεις γραφική ύλη, ε, χαρτί. Ε, Χρειαζόντουσαν έντυπα επί εντύπων για να γίνει αυτό. Και είπαμε ας το αλλάξουμε αυτό. Ό,τι και να γίνει, 25% του άμεσου κόστους θα είναι το έμεσο και θα σας το καταβάλουμε. Ε, εκεί δεν μπορείτε να κάνετε λάθος, γιατί είναι ένα κατά αποκοπήν ε, πόσο. Επίσης, υπήρχαν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στις συμφωνίες για τις επιδοτήσεις. Ε, μια συμφωνία για το α πρόγραμμα, μια άλλη συμφωνία για κάτι άλλο και ε, είχαμε πελαγώσει. Γι' αυτό είπαμε ότι ε, θα γίνει ενιαία αυτή η διαδικασία. Έχουν γίνει βήματα. Απλούστευση είναι πραγματικά ο σωστός όρος, γιατί γίνεται απλούστερη η διαδικασία. Αλλά καμιά φορά υπάρχουν κάποιες συνέπειες ε, που δεν ε, τις είχαμε υπολογίσει και δεν είναι και σκεμμένες όταν προσπαθείς να απλουστεύσεις κάτι και χρειάζεται αναθεώρηση, στάθμιση, τι κάναμε, πώς το κάναμε. Πάντω έχουμε πετύχει πολλά. Το ελεγκτικό συνέδριο τι έκανε. Όταν ξεκίνησα εγώ, ανέλυαν τις συναλλαγές του προγράμματος πλαίσιο 7 και θα ερχόντουσαν εδώ και θα έλεγαν ε, ναι, αλλά δεν κάνατε αυτά στην απλούστευση. Ναι, γιατί δεν είναι συνέπεπτε χρονικά, γιατί ανέλυαν ένα παρελθόν ε, πρόγραμμα ερευνητικό. Τώρα πραγματικά πιστεύω ότι θα μπούμε και ελπίζω σε ένα νέο κύμα πλουστεύσεων. Εγώ δεν θα είμαι εδώ για να το ζω, αλλά θα τα παρακολουθώ απ' έξω. von ECR ist niemand. Το ECR απουσιάζουν και από την ΚΟΕ κύριος Φλάναγκαν επίσης. Έχω όμως εγώ να σας κάνω ερώτηση, όχι προς εσάς κύριε Επιτροπέ, αλλά προς το ελεγκτικό συνέδριο. Στην περασμένη του έκθεση, το ελεγκτικό συνέδριο τόνισε πάρα πολύ την τεχνική βοήθεια, το technical assistance. Τι εννοείτε, πώς θέλετε εδώ να διευρυθεί. Γι' αυτό που ρώτησε η κυρία Πένκοβα, σε χώρες που έχουν μεγάλες δυσκολίες να συμμετέχουν σωστά στο πρόγραμμα, στα προγράμματα. Τι θα πρότεινε το ελεγκτικό συνέδριο, τι θα υποστήριζε ε, τι θεωρεί ιδιαίτερα θετικό έτσι ώστε να δημιουργηθεί η συνειδητοποίηση στις χώρες αυτές αλλά και η ικανότητα συμμετοχής στα προγράμματα ή στα πλαίσια της έρευνας και της ανάπτυξης και της καινοτομίας να βελτιωνόμαστε. Δεύτερη ερώτηση, πάλι και εγώ θα ρωτούσα για την απλούσταυση στον, ε, τον Επίτροπο. Κύριε Κούς, δεν είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, περιπλέκει τα πράγματα. Εμείς τα περιπλέκουμε. Γιατί εμείς είμαστε τελικά οι νομοθέτες, εμείς κάνουμε τις προτάσεις, εμείς ασκούμε κριτική και πάντα υπάρχει αντίδραση στην όποια δράση. Άρα εμείς ε, φτιάχνουμε ένα πιο περίπλοκο κόσμο. Και σας ερωτώ, πού βλέπετε ε, συγκεκριμένες δυνατότητες απλούστευσης γιατί πολύ συχνά βλέπουμε δαπάνες προσωπικού που δεν είναι επιλέξιμες και θεωρούνται προβληματικές, ε, που είναι κόστος που δεν μπορεί να καλυφθεί, γιατί ε, ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται είναι πολύ περίπλοκος ως κατασκεύασμα. Εγώ έχω ασχοληθεί στο παρελθόν ε, και πραγματικά αν είσαι μικρομεσαία επιχείρηση ή κάποιος που για πρώτη φορά κάνει την αίτηση, είναι κικαιώνας, τεράστια πρόκληση. Ε, πού βλέπετε λοιπόν χώρο εκεί για απλούστευση και πού θα είχε νόημα να γίνει κάτι τέτοιο. Και πάλι μια ερώτηση προς το ελεγκτικό συνέδριο. Η αναφορά βάση επιδόσεων, αυτό το performance, η ε, performance reporting. Αν δούμε τι γίνεται στην έρευνα και την επιστήμη, αυτό τι σημαίνει. Είναι δύσκολο. Γιατί όταν είσαι ερευνητή, ψάχνει κάτι, δεν ξέρει το τελικό αποτέλεσμα, ποιο θα είναι και πόσο επιτυχέ. Πώ μπορείτε να έχετε εκεί δείκτε εκ των προτέρων για να μετράτε την επιτυχία ή και την ενδεχόμενη αποτυχία. Όταν ερευνά κάτι και ψάχνει ερευνητή, μπορεί και να αποτύχει. Δεν σημαίνει ότι θα το βρει πάντα αυτό. Και όταν αρχίζει κάτι να ψάχνει, δεν <laughs> καταλήγει πάντα εκεί που θέλει, όταν το θέλει. Ε, και δεν τηρείς και τις προθεσμίες πάντα. Εκεί στην έρευνα λοιπόν και την καινοτομία και την επιστήμη τι μετράτε ως απόδοση και τι αναφέρετε στις εκθέσεις μετά. Thank you, for, for your questions. I think... Uh, Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις αυτές. Θα ξεκινήσω εγώ και θα δω αν θα προσθέσει κάτι ο Επίτροπος. Για την τεχνική βοήθεια Να σας πω πως ε, πρόσφατα εγκρίναμε το ετήσιο πρόγραμμα για το 2000 για το Horizon 2020 και εδώ έχουμε συμπεριλάβει και μια ειδική έκθεση για τη διεύρυνση του Horizon 2020 και εκεί νομίζω ότι θα απαντήσουμε κάποιες ερωτήσει που έκαναν οι ευρωβουλευτές. Δηλαδή, ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση και τι πρέπει να γίνει. σε κάποιο βαθμό το σημείο αυτό το έχουμε τοποθετήσει σε μία από τις συστάσεις μας, όπου η σύστασή μας είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει μία εκστρατεία ενημέρωσης μέσω σεμιναρίων, μέσω ημερίδων στα κράτη-μέλη, Και αυτό χρειάζεται ακόμα πιο πολύ αν προσπαθεί κάποιος να προσελκύσει νεότερους και πιο καινούριους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα. Από κάποια κράτη, με συγχωρείτε, πρέπει να ρωτήσω Αυτός που τους ενοχλεί ο ήλιος. Θέλετε να κλείσουμε τελείως τα ρολά ή συμφωνείτε με το να αφήσουμε να περνάει λίγο ήλιος. <laughs> so the majority is for sun. <laughs> Οι περισσότεροι λοιπόν θέλουν και λίγο ήλιο. Σας ευχαριστώ. Ah, ah. Με συγχωρείτε που σας ε, διέκοψα για αυτά τα θέματα. Εγώ πάντα θέλω περισσότερη διαφάνεια, οπότε καταλαβαίνετε ήλιο για να δώσει διαφάνεια. Για την τεχνική βοήθεια νομίζω ότι είπα ό,τι μπορούσα και με μεγάλη χαρά βλέπω ότι στην ε, ειδική αυτή έκθεση αναφερόμαστε στο ετήσιο πρόγραμμα και θα σας δώσουμε συγκεκριμένες ε, απαντήσεις όταν θα έρθει η κατάλληλη στιγμή. Για την ε, έκθεση, για τα αποτελέσματα, είστε Έχετε δίκιο. Αν αντιμετωπίσει κανείς ε, το σύστημα αυτό με τους δείκτες απόδοσης και δει και το κεφάλαιο 3 της ετήσιας έκθεσης, θα καταλάβει πως δεν ικανοποιείται απόλυτα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το σύστημα έτσι όπως υπάρχει. Στην τρέχουσα έκθεση, αν κοιτάξετε το τέλος, το τέλος του κεφαλαίου, του μιλάμε για κάποιους δείκτες οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν φέτος για να αξιολογήσουμε τις ε, επιδόσεις και την απόδοση διαφόρων ε, έργων και κυρίως ποια ήταν ε, τα, ποιοι ήταν οι στόχοι και ποια ήταν τα αποτελέσματα. Κοιτάξαμε project τα οποία ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί για να δούμε αν το κόστος ευθυγραμμίζεται με την πρόοδο που αναφέρεται, με το ρυθμό εφαρμογής, γιατί πολλές φορές έχουν ε, πληρωθεί περισσότερα από ό,τι έχουν επιτευχθεί. Και τέλος, κοιτάμε και σε ένα, δίκτυο που είναι πολύ σημαντικός και ανέφεραν κάποιοι συνάδελφοι αυτό της ε, διάχυσης του αποτελέσματος. Κοιτάξαμε λοιπόν περιπτώσεις που διαδόθηκαν μερικώ μόνο τα αποτελέσματα. Αυτοί είναι κάποιοι δείκτες, σα δίνω κάποια παραδείγματα. Έχουμε και άλλο ένα στοιχείο για την απόδοση που είναι το εξής. Εμείς έχουμε ξεκινήσει ένα πιλωτικό πρόγραμμα για την αναφορά στην απόδοση Τη απόδοση, δηλαδή του χρόνου, το ελεκτικό συνέδριο θα παρουσιάσει μια διαφορετική έκθεση για την απόδοση τη Ευρωπαϊκή Δράση. Και ένα από τα θέματα που θα θελήσουμε να δούμε σε με λεπτομέρειε είναι αυτό του Horizon 2020. Το έχουμε βάλει στο μάτι γιατί είναι δύσκολο, γιατί είναι μεγάλη πρόκληση, γιατί έχουμε πολλές ερωτήσεις για το πώς και πόσο αποδοτικό είναι. Για το θέμα της απλούστασης έχουμε μια γενική σύσταση σχετική. Καταλαβαίνω λοιπόν πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να προσπαθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Αν θέλετε τώρα πιο συγκεκριμένα παραδείγματα για τη σύσταση αυτή θα μπορούσα να αναφερθώ σε ένα μέτρο, δηλαδή να εγκαταλείψουμε την απέτηση υπολογισμού ωριαίου ε, κόστους για προσωπικό το οποίο ε, δουλεύει αποκλειστικά και μόνο για τα ευρωπαϊκά project. Είναι μια λίγο τεχνική, τεχνητή απέτηση και βέβαια ε, υπάρχει κίνδυνος να καταπατήσει κανείς ε, το κανόνα της διπλής οροφής στη χρηματοδότηση. Πρέπει λοιπόν να αποφύγουμε τέτοιου είδους κινδύνους, να μην έχουμε δηλαδή παράλληλα συστήματα τα οποία θα εμφαρμόζονται ταυτόχρονα και να καταργήσουμε με τον τρόπο αυτό ένα κομμάτι του προβλήματος. Ένα ακόμα παράδειγμα είναι η ανάγκη ξεκαθαρίσματος ε, κατά πόσο είναι επιλέξιμες επιπλέον αμοιβέ ε, για το project. Αυτό δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρο. Για τους δικαιούχους βέβαια. Και πολλές φορές κάνουν λάθη. Για να μην έχουμε λοιπόν δραματικές αλλαγές, αυτό που κάνουμε είναι ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δει τι χρειάζεται να βελτιωθεί σε συγκεκριμένο σημείο. Δεν χρειάζεται δηλαδή μια επαναστατική αναπροσαρμογή του συστήματος, αλλά να αναμορφωθεί με στοχευμένο τρόπο έτσι ώστε να ξεπεραστούν τα προβλήματα τα οποία οδηγούν τους ε, δικαιούχους σε σφάλματα. Και ε, σφάλματα τα οποία δεν μπορούν να βρουν ε, οι ελεγκτικές διαδικασίες με αποτέλεσμα να καταλήγουν σε εμάς. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Ο επίτροπο τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, σχετικά με την πρώτη σας ερώτηση για το πόσο δύσκολο ε, είναι να εκτιμήσεις το, επιλέξιμο, το ε, μη επιλέξιμο κόστος, να κάνεις μια διάκριση. Προσπαθήσαμε να κάνουμε κάτι καινούριο και προσβλέπουμε και στη βοήθεια του ελεκτικού συνεδρίου. Είναι αυτό το σύστημα με το καταποκοπή ποσών αντί να βλέπουμε και να μετράμε αν είναι επιλέξιμο, τι είναι και δεν είναι, δίνεις εκεί ένα ποσό. Υπάρχει πρώτη φάση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το πρώτο στάδιο και θα επανέλθουμε αργότερα όταν θα έχουμε περισσότερα στοιχεία. Ε, δεν ξέρουμε ποτέ τι συνέπειες ε, ε, δεν είχαμε υπολογίσει και στις οποίες δεν ε, προσβλέπαμε να έχει. Ε, θα τα ξαναπούμε. Για τους δείκτες τώρα. Για τους δείκτες είναι δύο διαφορετικά πράγματα εδώ. Το, έχει, το ένα έχει να κάνει με τη βασική και τη θεμελιώδη έρευνα και το άλλο έχει να κάνει με την καινοτομία. Για τη θεμελιώδη έρευνα φυσικά δεν ξέρεις πού θα καταλήξεις ούτε από τώρα σε 50 χρόνια. Γνωρίζεις όμως ότι ένας πάρα πολύ καλός ερευνητής που κάνει πολύ σπουδαίες ε, δημοσιεύσεις, ε, τον ε, παραπέμπουν πολλές φορές, τον αναφέρουν στη βιβλιογραφία. σε δημοσιεύματα και σε δημοσιεύσεις που είναι πάρα πολύ χρήσιμα και για το ελεκτικό συνέδριο. Κάποιο σαν τον Σερ Πίτερ Ράτκλιφ, που τώρα βέβαια είναι νομπελίστας, αλλά πριν πάρει τον Νόμπελ είχε εντυπωσιακή ε, ποσότητα δημοσιεύσεων. Και είναι αρκετά περίεργο ε, ότι αυτό για τις επιχειρήσεις είναι ε, πιο δύσκολο. Οι επιχειρηματίες αποτυχάνουν ξανά και ξανά και κάποια μέρα πετυχαίνουν. Πώς θα χρηματοδοτήσεις κάποιον που θα αποτύχει αλλά κάποια μέρα μπορεί και να πετύχει και να το βοηθήσει σε αυτή την πορεία για να κάνει κάτι θαυμάσιο. Ε, και πάλι επανέρχομαι στο παράδειγμα. Χρηματοδοτήσαμε μια εταιρεία που λέγεται InFarm. Δεν θυμάμαι πόσα τους δώσαμε, ένα εκατομμύριο ή ούτε καν. Και ξαφνικά μοχλεύσανε 88 εκατομμύρια από τον ιδιωτικό τομέα, από επενδυτές. Και αυτό ενδεικτικό είναι, οι δείκτες, σε πάση περιπτώσει. Πάντα υπάρχουν οι δείκτες, αλλά είναι σχετικοί και αυτοί. Είναι μία ψηφίδα μόνο δεν θα πρέπει να προσανατολιζόμαστε ούτε εσείς, ούτε εμείς, ούτε το ελεγκτικό συνέδριο σε δείκτες. Να βλέπουμε και την ανθρώπινη πλευρά, να ξέρουμε ποιοι είναι οι άνθρωποι στους οποίους επενδύουμε ε, και καμιά φορά θα αποτύχουν. Αλλά το σημαντικό, Πρόεδρε, είναι ότι είναι λιγότερες οι αποτυχίες και περισσότερες οι επιτυχίες όταν κάνουμε τον απολογισμό μας. Ε, αυτή είναι η ζωή, λέει η Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Επίτροπε, έχετε άλλες ερωτήσεις να υποβάλλετε. Από ό,τι βλέπω όχι. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα καλύτερα σας ευχόμαστε και σας ευχαριστούμε πολύ για την ε, πολύ καλή σας ε, δουλειά και λυπούμαστε πάρα πολύ που φεύγετε. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή αλλά ειλικρινά ε, μας άρεσε πάρα πολύ η δουλειά σας, η συνεργασία με την Επιτροπή και ευχαριστούμε πάρα πολύ ε, για τη δουλειά που κάνατε, που σεβαστήκατε πάρα πολλές από τις συστάσεις μας, τις απόψεις μας και που ε, το, τα δικά μας τα προγράμματα έρευνας και καινοτομίας τα καταστήσατε αποτελεσματικότερα, καλύτερα, με βέλτιστες πρακτικές και παράλληλα προσπαθήσατε να συμπεριλάβετε και περισσότερα κράτη-μέλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, σεβόμαστε ιδιαίτερα εσάς και μέσω ημών και τη γενική σας διεύθυνση. So, now we have to wait a little bit on, uh, Τώρα θα πρέπει να περιμένουμε λίγο για να έρθουν όλοι οι υπόλοιποι. 5 λεπτά διάλειμμα. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ähm, wir dürfen wieder starten. Ich äh, begrüße. Äh, λοιπόν, καλωσορίζω τον κύριο Πιατρορούσο, μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου η συνεργάτη σα είναι πάρα πολύ καλή όταν αναφέρομαι σε κάποιον από τον δείχνει και με το δάχτυλο για να ξέρω ποιο είναι. Ε, θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω να τοποθετηθείτε και μετά ο κύριο Σεντόφσκι και κατόπιν θα ακολουθήσουν και ευχαριστώ πολύ που τα έχουμε τόσους πολλούς ε, γενικούς γραμματείς ε, που ήρθαν κοντά μας. Ε, χαίρομαι που βρήκατε το χρόνο και μας κάνατε την τιμή σήμερα. Χαιρόμαστε που θα ακούσουμε τις σα και μετά θα σας κάνουμε ερωτήσεις και θα ξεκινήσει η συζήτηση. Αγαπητέ κύριε Πιέτρο Ρούσο, παρακαλώ πολύ, έχει το λόγο.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 Κυρία Πρόεδρε, αγαπητά μέλη της Επιτροπής, είναι χαρά για μένα που μπορώ να σας παρουσιάσω σήμερα το κεφάλαιο 10 της ετήσιας έκθεσης του ε, συνεδρίου. Εκεί έχουμε την αξιολόγηση για τις διοικητικές δαπάνες, αξιολόγηση ε, όλων των ευρωπαϊκών ε, θεσμών. Το 2018 οι πληρωμές στο πλαίσιο του τομέα υπαριθμών 5 ανήλθαν σε 9,9 εκατομμύρια ευρώ ή αν θέλετε περίπου το 6,3% του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αξιολόγηση το 2018 είναι θετική και οι δαπάνες για την δίκηση δεν έχουν ε, σφάλματα. Ε, φέτος ε, κάναμε δειγματοληπτικό έλεγχο 45 συναλλαγών, εκ των οποίων 9 αφορούσαν άλλους θεσμούς. Τρεις συναλλαγές για το Συμβούλιο, δύο συναλλαγές για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και μία συναλλαγή για κάθε μία Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Επιτροπή των Περιφερειών, ε, τον επόπτη, ε, τον Ευρωπαϊκό Επόπτη της Προστασίας Δεδομένων και τον Ευρωπαϊκό και την Ευρωπαία διαμεσολαβήτρια. Όσον αφορά άλλους θεσμούς, ε, ε, δεν βρήκαμε σφάλματα στις αναλλαγές και γι' αυτό δεν έχουμε συγκεκριμένες ε, παρατηρήσεις για τους άλλους θεσμούς. Κυρία Πρόεδρε, ε, κύριε Συγητά, αγαπητά μέλη της Επιτροπής, ε, τελειώντας θα ήθελα να ευχαριστήσω το προσωπικό του συνεδρίου ε, για τη δουλειά του όλα αυτά τα χρόνια και προφανώς και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Και εμείς, λέει η Πρόεδρος, ε, τώρα, το λόγο έχει ο εισηγητής, ο κύριος Τόμας Τεντόφσκι Εγώ θα μιλήσω τσέχικα, γιατί μερικές φορές είναι δύσκολο για μένα να μπω σε λεπτομέρειες και δεν είμαι σίγουρος ότι θα κατανοήσουν ε, όλοι τα αγγλικά μου, όλες τις λεπτομέρειες που θέλω να πω, ε, εφόσον μιλώ για κάποια συγκεκριμένα θέματα που αφορούν στην απαλλαγή. Λοιπόν, στα τσέχικα τώρα αξιότιμε αξιότιμα μέλη του ελεγκτικού συνεδρίου, αξιότιμη γενική γραμματής, αξιότιμοι συνάδελφοι. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω το ελεγκτικό συνέδριο για τη δουλειά που μας παρουσίασε και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί όπως και κατά τα προηγούμενα έτη το ελεγκτικό συνέδριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι πληρωμές το 2018 ε, δεν περιλάμβαναν πολλά σφάλματα και επίσης ότι τα συστήματα ελέγχου ήταν αποτελεσματικά. Για τους άλλους θεσμούς ε, το ελεγκτικό συνέδριο ε, δεν κατέληξε στο να εντοπίσει μεγάλες ελλείψεις. Ε, δηλαδή η διαχείριση σε άλλους θεσμούς το 2018 ήταν ικανοποιητική, αποτελεσματική και οι θεσμοί ήθελαν να ελαχιστοποιήσουν τις δαπάνες τους και το κόστος για το προσωπικό να το κρατήσουν σε επίπεδο 2017, που τα κατάφεραν. Βέβαια δεν ήταν εύκολο αυτό για τους υπόλοιπους θεσμούς, γιατί ήταν πολύ σημαντικό να διατηρήσουν κάποιες ε, βασικές θέσεις. Ε, πρόκειται για τη συνέχεια ε, κάποιοι θεσμοί που έπρεπε να περιορίσουν τις ε, θέσεις απασχόλησης, εκεί ήταν πολύ δύσκολο να περιορίσουν το προσωπικό. Γι' αυτό εκτιμώ ιδιαίτερα τη δουλειά που κάνατε. Και τελειώνοντας θέλω να συγχαρώ όλους τους ε, θεσμούς για τα αποτελέσματα τα οποία παρουσίασαν το 2018 και σας εύχομαι για το 19 τόσο καλά αποτελέσματα έτσι ώστε να μπορούμε και πάλι να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν ένα πολύ καλό παράδειγμα για το πώς πρέπει κανείς να, ε, να χειρίζεται τον ενωσιακό προϋπολογισμό. Ωραία. Τόμας, πολύ ωραία. Και τώρα, πριν λάβουν το λόγο οι σκιώδεις ξεκινάμε με το ε, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, Γενικός Διευθυντής, κύριος Πλάκο. Ε, ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και ε, με χαρά να σας δώσουμε και το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εσάς και τον εισηγητή που μας δώσετε τη δυνατότητα να συμμετέχουμε εδώ για την απαλλαγή, για τον προηγούμενο προλογισμό. Ο γραμματέας μας δεν είναι εδώ, οι γραμματέας μας δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή, αλλά εκπροσωπείται από ε, τον επικεφαλής ε, του γραφείου της και να σας πω πως για μας ήταν ε, το 2018 μια έκτατη χρονιά γιατί είχαμε μεγάλη ένταση δικαστικής εργασίας. Είχαμε ένα ρεκόρ προσφυγών Πάνω από 1.500 ε, υποθέσεις κλείσαμε, που ήταν και αυτό ρεκόρ. Και σε σχέση με το 2017 είχαμε μία ε, αύξηση ε, του 11% και είχαμε και 1.600 περίπου νέες υποθέσεις που ήταν ο αριθμός ο υψηλότερος στην ιστορία του θεσμού μας. Αυτή λοιπόν η... αυτός ο όγκος εργασίας δικαστικής συνοδεύεται από μια μείωση του χρόνου διεκπαιρέωσης των υποθέσεων. 15,7 μήνες ε, λοιπόν ε, στο δικαστήριο και 17 ε, και 12 με συγχωρείτε για το πρωτοδικείο. Και αυτά εξηγούνται από το γεγονός πως είχαμε αλλαγές στον κανονισμό μας και το γεγονός πως πολλά θέματα ανταγωνισμού το 2017 επιλύθηκαν. Είχαμε λοιπόν πολύ εντατική δικαστική εργασία και να σας πω πως είχαμε και στο δικαστήριο θέματα με δική μας ε, πρωτοβουλία μεταξύ ε, του Πρωτοδικείου και του Δικαστηρίου του 2018 έτσι ώστε να έχουμε ποιοτική δικαιοσύνη, αποδοτική και αποτελεσματική. Πρώτα απ' όλα άνοιξε η πλατφόρμα η πολύ γλωσσή και ασφαλής του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου που επιτρέπει στα κράτη-μέλη και δηλαδή στα ανώτατα και στα κυρωτικά δικαστήρια των ε, κρατών μελών, όπως επίσης και στο ΔΕΚ, να ανταλλάσσουν με ασφαλή τρόπο ε, πληροφορίες, αποφάσεις και να κάνουν και κάποιες ε, έρευνες για δικαστικά θέματα στο παρελθόν, εκτός από τα απόρριτα ε, έγγραφα, είχαμε και κάποια άλλα, τα οποία είχαμε δημοσιεύσει στο ίντερνετ και τώρα βρίσκονται και αυτά σε τούτο το δίκτυο. Το δεύτερο, στο οποίο ήθελα να σταθώ, είναι η πρωτοβουλία του 10 από 1η Ιουλίου του 2018 για να έχουμε ανώνυμη δικαστική πληροφορία που δημοσιοποιείται για τα προδικαστικά ερωτήματα για φυσικά πρόσωπα και την ε, υποκατάσταση των ανθρώπων από αρχικά, των ονομάτων των ανθρώπων που εμπλέκονται με αρχικά κάτι το οποίο επιτρέπει να ενισχύσουμε την προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων. Τρίτον, πρόοδος στην χρήση της ε, εφαρμογής κούρια με πάνω από 1.500 χρήστες που άνοιξαν λογαριασμό και από 1η Δεκεμβρίου του 2018 είναι υποχρεωτική η χρήση αυτής της εφαρμογής για τις ανταλλαγές μεταξύ των γραμματέων του δικαστηρίου και των εκπροσώπων των ε, διαδίκων. Ένα τέταρτο σημείο είναι το 2018 το project για την χρήση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης που είχε σκοπό να αντικαταστάσει την πληθώρα ε, των εφαρμογών που χρησιμοποιούσαμε μέχρι σήμερα έτσι ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική η ίδια εκπαιρέωση και βέβαια τα όσα είχαμε στην έκθεση του 14, την έκθεση 14 για το 2017. Για τη διοικητική μας δράση να σας πω πως το 2018 ξεκινήσαμε μία μεταρρύθμιση των ε, διοικητικών μας δομών. Πλέον έχουμε τρεις γενικές διευθύνσεις και όχι τέσσερις, έτσι ώστε να έχουμε κάποια συνέργεια και να εξορθολογήσουμε τη ροή εργασιών, έτσι ώστε να βελτιώσουμε και την συνεισφορά ε, στην δικαστική εργασία αυτών των διευθύνσεων δεν είχαμε παρατηρήσει από το, ελληνικό, το συνέδριο για το σημείο αυτό. Άρα λοιπόν η, αυτό ενισχύει την ιδέα πως τα οικονομικά μας τα διεκπαιρεώνουμε με απόλυτη κανονικότητα. Η διαχείριση πόρων είναι πάρα πολύ ε, στενή. Εκτέλεση πληρωμών 99,2, ε, ποσοστό απασχολησιμότητας 97%. Άρα λοιπόν αυτά ε, και είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εξαιρετική δουλειά του δικαστηρίου επίσης, που είναι διεθνώς ε, γνωσμένου κύρους. Και έρχομαι τώρα στο ελεκτικό συνέδριο το ίδιο, στον κύριο Εντουάρδο Γκαρσία Ρουίθ. Ή τα λέω καλά. γιατί πάντα μπερδεύομαι γιατί είναι τρία ονόματα. Εγώ φταίω, όχι εσείς και δεν τα πετυχαίνω με τη σωστή σειρά κάθε φορά. Ε, την άλλη φορά ε, θα τα αφήσω στην Ισαμπέλ Γκαρθία να τα πει που τα ξέρει τα Ισπανικά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμη Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Το 2018 το ελεγκτικό συνέδριο συνέχισε τις εργασίες του ε, πιστοποίησης, ελέγχουν της νομιμότητας, ε, της τυπικής διαχείρισης και της καλής διαχείρισης. 72 έγγραφα δημοσιεύσαμε, 6 αιτήσει εκθέσεις μεταξύ αυτών και 35 ειδικέ εκθέσεις. Και για πρώτη φορά, και νομίζω ότι είναι σημαντικό να το πούμε, ε, δημοσιεύσαμε μία μόνο έκθεση που περιλαμβάνει αποτελέσματα του οικονομικού ελέγχου που κάναμε στους εξωτερικούς οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η ενοποιημένη έκθεση θα διευκολύνει ε, την ανάγνωση και την ανάλυση των αποτελεσμάτων. 6.500 ημέρες ε, ελέγχου κάναμε σε όλα τα κράτη-μέλη και στα 28 και επιθεωρήσεις σε 26 τρίτες χώρες. Ε, τώρα, κάναμε εκθέσεις για διάφορα θέματα που σας ενδιαφέρουν και το κοινοβούλιο σα, άρα και τον Ευρωπαίο πολίτη. Ανανεώσιμε πηγές ενέργειας στην Ήπεθρο, ε, σύμφωνο σταθερότητα και ανάπτυξη στο πρόγραμμα Erasmus συν ατμοσφαιρική ρήπανση, κέντρα αριστεία και έρευνας, μηχανισμό για τους πρόσφυγες στην Τουρκία. Ε, επίσης, το 2018 προχωρήσαμε ε, στους ελέγχους που κάνουμε για τη δήλωση αξιοπιστίας. Ε, τώρα αλλάζει, ξέρετε, η μεθοδός μας, μεταρρυθμίζεται και θέλουμε να είμαστε σε θέση να λαμβάνουμε καλύτερα υπόψη τους εσωτερικούς ελέγχους που γίνονται στα κράτη-μέλη και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τρόπο ώστε να μπορούμε να εντοπίζουμε καλύτερα τα προβλήματα και να αυξήσουμε και να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα των ελέγχων. Για τη διαχείριση ήταν καλοί οι δείκτες. Να σας δώσω ένα παράδειγμα κάναμε μια έρευνα μεταξύ των χρηστών των εκθέσεών μας, το 87% θεώρησαν τη δουλειά μας χρήσιμη και 78% ε, θεωρούσαν ότι είχαν θετικό αντίκτυπο σε ό,τι αφορά την κάλυψή μας ε, στα social media έχει αυξηθεί και σε ό,τι αφορά τις συστάσεις εδώ μετριάζεται κάπως ο αντίκτυπος και μετράμε εκεί. Το 24% των συστάσεων που έχουμε ε, απευθύνει το 2014 σε ειδικέ εκθέσεις έχουν ήδη εφαρμοστεί. Αυτό δείχνει ότι προσπαθεί το ελεγκτικό συνέδριο να έρθει πιο κοντά στον πολίτη και να βοηθήσει να βελτιωθεί η αξιοπιστία του πολίτη στο ευρωπαϊκό εγχείρημα. Το ελεγκτικό συνέδριο ε, με αυστηρότητα ε, χειρίζεται τα δημόσια οικονομικά του με κάλυψη 98% με θετικές επιθεωρήσεις εσωτερικές και εξωτερικές. Ο εσωτερικός ελεγκτής ε, έκανε μια εκτίμηση για τα έξοδα ταξιδίου και παράστασης των μελών του ελεκτικού συνεδρίου το έτος αυτό. Γιατί ένα παλιό μέλος ε, του ελεκτικού συνεδρίου είχε μια υπόθεση η οποία στάλει στην Όλαφ. Υπήρχε επίση και μια ε, ε, περίπτωση απάτης, αλλά είναι μεμονωμένη η περίπτωση αυτή και το ελεγκτικό συνέδριο έχει εντείνει ε, τους ελέγχους για να προλαμβάνουμε τέτοια φαινόμενα στο μέλλον. Επίσης, βελτιώθηκε η ασφάλεια των εγκαταστάσεων για το προσωπικό. Έχουμε περιβαλλοντική πιστοποίηση και ε, βελτιώσαμε και την ε, προαγωγή των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις. Βέβαια, απέχουμε πόρο από την ισορροπία φύλου που θέλουμε ε, στις ελεγκτικές υπηρεσίες και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση αυτή. Συνοψίζω, το 2018 το ελεγκτικό συνέδριο ανταποκρίθηκε στην αποστολή του, βοηθώντας το Κοινοβούλιο και βοηθώντας στη βελτίωση της διαχείρισης και στη λογοδοσία Είμαστε δρακόντιοι στη διαχείρισή μας και όπως σας είπα ε, έχει αυξηθεί και η ποιότητα και η ποσότητα των εκθέσεων μας. Θα θέλαμε εδώ να τονίσουμε το σημαντικό ρόλο που έπαιξε το προσωπικό μας, οι ελεγκτές, οι μεταφραστές, ε, οι ε, πληροφορικάροι, το τεχνικό και διοικητικό προσωπικό για να φτάσουμε σε αυτή την έκβαση και το αποτέλεσμα του επιτυχές. Ε, θα βρείτε στα αντίστοιχα έγγραφα περισσότερες προφορίες και φυσικά είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση τυχόν έχετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα αρχόμαστε στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Πρώτα απ' όλα επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μου δίνετε εδώ να παρουσιάσω τις εργασίες της ΟΚΕ. Να σας πω πως ε, δεν είχαμε σημαντικά ασφάλματα, έτσι είπε το ελεγκτικό συνέδριο και εκτέλεση 98,7%. Είμαστε δηλαδή το πιο αποτελεσματικό από όλα τα όργανα εστιάσαμε πολύ στο ψήφισμα το οποίο ενέκρινε το Μάρτιο για την απαλλαγή του 17 του Κοινοβούλιο και σε κάποια παραδείγματα είπαμε η ενίσχυση της πολιτικής και διοικητικής συνεργασίας με την Επιτροπή Περιφερειών και το Κοινοβούλιο οι εκστρατείες και η προώθηση του περιβάλλοντος εργασίας με σεβασμό, ο δεοντολογικός κώδικας για τα μέλη και η έγκριση μιας στρατηγικής για την πολιτική της πληροφορικής. Για την πολιτική μας εργασία είχαμε μια σημαντική συμβολή στις νομοθετικές εργασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 115 γνωμοδοτήσεις που εγκρίθηκαν, ε, γνωμοδοτήσεις και εκθέσεις με τα κέντρα ε, Going Local που μας επιτρέπουν να είμαστε σε επαφή με την κοινωνία των πολιτών στα κράτη-μέλη. Για την πολιτική επικοινωνία, ο αριθμός επισκεπτών έφτασε τους 10.000, 1% λοιπόν αύξηση. Είμαστε στο Twitter, στο Facebook και θα ανοίξουμε και πρόσφατα και σύντομα Instagram και έχουμε πολλούς χιλιάδες επισκέπτες καθημερινά. Για την πολιτική συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πέραν των παραδοσιακών επαφών που έχουμε μεταξύ των Προέδρων Τμήματων και των Ισχυτών με τους ομολόγους του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου, είχαμε την κοινή δήλωση ο κύριος Νταλή με τον κύριο Ταγιάννη το Δεκέμβριο του 2018 με σκοπό να ευαισθητοποιήσουν την κοινή γνώμη για την ψηφοφορία που έπρεπε να γίνει στις ευρωπαϊκές εκλογές και σε επαφές που γίνονται στα πλαίσια της διάσκεψης προέδρων. Συνεργασία και στο διοικητικό κλάδο με σημαντική προόδο σε θέματα ασφάλειας, όπως επίσης και διερμηνίας. Και κυρίως στο δεύτερο αυτό, να σας πω πως οι εργασίες προετοιμασίας μας επέτρεψαν φέτος να υπογράψουμε μία συμφωνία για την παροχή υπηρεσιών που καλύπτει τα δύο, μας θεσμικά, τα δύο αυτά όργανα. Επίσης, προσπαθούμε να εξεύρουμε συνέργεια για το θέμα της μετάφρασης με, άλλες, με άλλα όργανα, με, το, με την έψο για το Foresight και με το Γραφείο Δημοσιεύσεων. Αποτελεσματικότητα διοικητική σε συνεργασία με την Επιτροπή των Περιφερειών τα έχουμε καταφέρει. Έχουμε ένα μοντέλο χρηστής διαχείρισης δημόσιου οργανισμού και πρέπει να σας πω ότι μαζί κάνουμε ε, την πληροφορική και την μετάφραση. Με ε, σημαντική εξοικονόμηση δαπανών. Θα μπορούσαμε βέβαια να κάνουμε κάτι παραπάνω και έχουμε μια συνεχή εξερεύνηση με τους εξωτερικούς μας συνεργάτες έτσι ώστε να συντονίζουμε και τις ιατρικές μας υπηρεσίες κτλ όπως επίσης και με το προσωπικό που υποστηρίζει τις αίθουσες συνεδριάσεων. Για αυτά λοιπόν έχουμε μια χρηστή διαχείριση σύμφωνα με το σύστημα EMAS, λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του περιβάλλοντος στην κατανάλωση ενέργειας, φυσικού αερίου και χαρτιού. Θέματα τα οποία ε, έχουμε προσπαθήσει με κάποιους δείκτες να ε, μειώσουμε την κατανάλωση με πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα για το μέλλον. Επίσης, σεβασμό στο χώρο εργασίας. Μία εκστρατεία ξεκίνησε το 2019, λέγεται Respect at Work και είναι μια σειρά πρωτοβουλειών και δράσεων για την ευαισθητοποίηση και για να επενθυμίσουμε πόσο σημαντικό είναι το περιβάλλον εργασίας στην οποία, στο οποίο θα πρέπει να γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και εδώ θα ήθελα να υπογραμμίσω πως η πολιτική μας αρχή έχει ένα συγκεκριμένο εργαλείο, ένα κώδικα διοντολογικό ανανεωμένο από το Μάρτιο πέρσι που υπενθυμίζει πως θα πρέπει να γίνεται σεβαστή η αξιοπρέπεια του εργαζομένου στον χώρο εργασίας. Γεωγραφική ισορροπία. 18% των εκπροσώπων κάτω από το 20% που θα θέλαμε. Έχουν πετύχει αυτό το στόχο, αλλά ελπίζουμε ότι σύντομα και εμείς θα τα καταφέρουμε. Δυστυχώς, το θέμα της ισότητας, αντίθετα στο θέμα της ισότητας των φύλων, έχουμε ε, τα καλύτερα αποτελέσματα από οποιοδήποτε όργανο. 54% στις μεσαίες θέσεις και 50% στις ανώτερες ιεραρχίες καταλαμβάνονται από γυναίκες. Είμαστε ικανοποιημένοι λοιπόν από τα αποτελέσματα αυτά. Προσπαθούμε πάντα να ασκούμε κριτική στις δικές μας επιδόσεις και πάντα προσπαθούμε να εμψυχωθούμε και να εμπνευστούμε από ό,τι κάνουν τα υπόλοιπα όργανα έτσι ώστε να βελτιωθούμε περισσότερο. Θα κλείσω εδώ, δεν θέλω να φάω το χρόνο σας, αλλά θα απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση έχετε να μου κάνετε ή και σε παρατηρήσεις. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσίασή σας καθώς και για το μέσο όρο της ισότητας που έχετε πετύχει. Ευχόμαστε τα αντίστοιχα και για τα άλλα θεσμικά όργανα. Πάμε τώρα λοιπόν στην Επιτροπή των Περιφερειών. Πέδρο Σερβία Μαρτίνεθ. Για να τον παρακαλέσω μας κάνει την ειδική του παρουσίαση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρία Χολμάιερ. Και ευχαριστώ πολύ που προφέρατε σωστά και το όνομά μου. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που μου απευθυνέται να έρθω σήμερα εδώ και ξεκινώ ευχαριστώντας τον συζητή τον κύριο ε, Σεχόφσκι, ε, με τον οποίο και εγώ ξεκίνησα με τον κύριο και μια πολύ καλή συνεργασία ε, και προβλέπω να συνεχιστεί. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι σας ομιλώ σήμερα ως ε, προσωρινός Γενικός Διευθυντής. Είμαι από τον Αύγουστο. Ο προκάτοχός μου ε, θα είναι εδώ και κατά την επόμενη χρονιά. Κυρίε και κύριοι, η διαδικασία της απαλλαγή είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για να εξετάσει κανείς λιγάκι αυτά τα οποία έχει πετύχει από κοινού. Και είναι και ένα τρόπο για να στρέψει το βλέμμα ε, και σε αυτό που μπορεί να βελτιωθεί. Θα ήθελα να εστιάσω την προσοχή μου σε τρία θέματα στρατηγική. Πρώτον, τα κοινά προγράμματα ε, για το 2019. Δεύτερον, η Συμφωνία Συνεργασίας ε, που υπογράψαμε πριν από πέντε χρόνια και τρίτον ε, τα επιτεύγματα για οικονομικές, οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους. Όσον αφορά τις ευρωπαϊκές εκλογές, κατά τη διάρκεια του 2018 ε, αναπτύξαμε πάρα πολλές προσπάθειες, οι δικές μας ομάδε συνεργάστηκαν με αυτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να διευκολύνουν το ε, μεγαλύτερο βαθμό συμμετοχή σε κάθε εκλογική περιφέρεια. Εμείς στηρίξαμε τις συζητήσεις με τους πολίτες σε όλες τις πόλεις και τις περιφέρειες της Ευρώπης. Επίσης, ε, τις ε, πρωτοβουλίες μας τις αναπτύξαμε με βάση αυτά που μας προτείνατε. Είχαμε υψηλά ποσοστά συμμετοχής, κυρίως ανάμεσα στους νέους. Και μαζί με σας επιθυμούμε τώρα να συνεχιστεί αυτή η θετική εμπειρία, κυρίως ε, κινητοποιώντας ε, τους νέους πολιτικούς, ε, τα, τους δημοτικούς συμβούλους κάτω των 40 ετών. Από κοινού το 18 και το 19 ε, αναπτύξαμε ε, συζητήσεις σε 23 χώρες, πάνω από 200 ε, τοπικές συναντήσεις με πάρα πολλούς συμμετέχοντες και σε πάρα πολλές περιφέρειες και πόλεις. Αυτά δείχνουν ότι είμαστε υπεύθυνοι και για τα επόμενα πέντε χρόνια. Την προηγούμενη εβδομάδα πάνω από 1.600 επαγγελματίες, επικοινωνιολόγοι ε, εδώ και στα δικά μας τα γραφεία είπαν ότι πρέπει να υπάρχουν κοινέ δράσεις. Αυτό έγινε στα πλαίσια της 10 ης Eurocom που οργανώνεται από κοινού ε, με την Επιτροπή των Περιφερειών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, και άλλους θεσμούς και και ξεκίνησαν εργασίες με τον κύριο Κάρας. Είχαμε λοιπόν ε, μια μεγάλη πολιτική συμμαχία. Τον Φεβρουάριο του 2014 το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή υπέγραψαν μια συμφωνία για πολιτική συνεργασία και εσείς ήσασταν ανάμεσα σε εκείνους ε, που πιέσατε και σε ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Χολμάρ. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο τα δικά μας ε, τα μέλη και εσείς ως ευρωβουλευτέ αγωνίζεστε όλοι από κοινού για να υπάρχει σωστή χρηματοδότηση και σωστές επενδύσεις στο επόμενο πουδουπού. Οι μας, οι πρόεδροι και οι πολιτικές ομάδες έχουν αυξήσει την ποσότητα και την ποιότητα της δουλειάς τους. Η δουλειά μας πλέον ακολουθεί τον νομοθετικό κύκλο ε, χάρη ε, του στρατηγικού σχεδιασμού. Και πάλι ξεκινήσαμε όλα αυτά και με τα νέα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνεργαζόμαστε με τους νέους ευρωβουλευτές σε μία σειρά επιτροπών. Ευχαριστώ παραδείγματος τον κύριο Σεντεχόφσκι για την βοήθεια που προσφέρει ε, στην Επιτροπή ΣΥΒΕΞ. Αυτό το αποκαλούμε ενεργό επικουρικότητα η Επιτροπή επιθυμεί μαζί με το Κοινοβούλιο να ε, εφαρμοστεί καλύτερα η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Και ως απόδειξη για την αποφασιστικότητά μας, η Επιτροπή έχει συστήσει ένα πιλωτικό δίκτυο ε, σχετικά με την εφαρμογή της ε, ενωσιακής νομοθεσίας. Τα αποτελέσματα θα τα μοιραστούμε μαζί σας. Αυτό θα γίνει αυτή την εβδομάδα για πρώτη φορά όπου θα καλωσορίσουμε τον πρόεδρο της ΑΚΟ, τον κύριο Ταγιάννη, ε, ε, στη δική μας τη συνδιάσκεψη περί επικουρικότητας. Αξιότιμα μέλη, θα ήθελα να τελειώσω ε, δίδοντας κάποια στοιχεία για τον προϋπολογισμό μας. Εμείς σταθεροποιούμε τους πόρους μας περίπου το 1% έχουμε κάνει εξοικονόμηση στα πλαίσια της συνεργασίας, όπως ήδη υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας. Αυτή η συνεργασία μας επιτρέπει σημαντική εξοικονόμηση, όπως αναφέρθηκε ήδη, στην πολιτική της πολυγλωσίας, στη χρήση των αιθουσών, στη συντήρηση των κριτηρίων, στην πληροφορική με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε μια διοικητική συμφωνία που μας έχει επιτρέψει να βελτιώσουμε τη συνεργασία σε πολλούς τομείς, στις μελέτες, στη διερμηνία, ε, στην ασφάλεια, στην πληροφορική παρότι ε, χάσαμε περίπου το 9% των πόρων μας το 2013, ε, προσπαθήσαμε να προσφέρουμε υψηλό επίπεδο ε, στα μέλη μας. Το πρόγραμμα δράσης μέχρι το 2021 για τις ίσες ευκαιρίες. Δίδουμε επιπλέον σημασία στην πληροφορική, νέα μέτρα για την τηλεκινητικότητα και τε, τηλεεργασία μάλλον. Και τέλος θέλω να υπογραμμίζω ότι μας ενδιαφέρει η βιώσιμη ανάπτυξη περιορίζοντας το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you very much. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας και την καλή συνεργασία. Και τώρα ερχόμαστε στην Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια Τζεζίρα Ντανιέλου. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Είναι η δεύτερη φορά που έχω την τιμή να απευθύνομαι στην Επιτροπή σας εξ ονόματος της κυρίας Έμιλι Οράιλι, ε, της ε, διαμεσοδη... Ε, ε, με συνοδεύει ο κύριος Αλεσάνδρο Ντελμπον, τμήματάρχης για το προσωπικό και τα οικονομικά. Θα σας ενημερώσω για τις βασικές μας δραστηριότητες, τις έρευνες και μετά τα εσωτερικά. Για τις έρευνες εξακολουθούμε να εφαρμόζουμε τη στρατηγική της διαμεσολαβήτριας προς το 2019 που είχε τη συντριπτική υποστήριξη του Κοινοβουλίου στην αρχή της τρέχουσας θητείας. Στόχος είναι να έχουμε ε, μεγαλύτερη ε, προβολή αντίκτυπο και ε, αποτελεσματικότητα ε, για τους πολίτες παντού για να καταπολεμήσουμε την κακοδιαχείριση. Ε, εξακολουθούμε να έχουμε αποτελέσματα. Αυξάνεται ο φόρτος εργασίας μας γιατί οι πολίτες στην Ευρώπη κατανοούν ότι μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Αυξήθηκαν οι καταγγελίες σε ιστορικό επίπεδο 880 ή 40%. Δεύτερον, ε, ως συνέπεια της αύξησης αυτής το 2018 ανοίξαμε έναν αριθμό ρεκόρ ερευνών 482 σε σύγκριση με τις 437 του 2017. Από αυτές τις έρευνες που ανοίξαμε 55 ήταν ε, για το δημόσιο συμφέρον δηλαδή ε, είχαν ε, αντίκτυπο ε, πέραν της μεμονωμένης υπόθεσης. Ε, τρίτον, για την προβολή εξακολουθούν να αυξάνονται οι ακόλουθοι στο Twitter, Instagram και στα υπόλοιπα μίντια. Είμαστε πολύ μικροί, αλλά ε, έχουμε πολλαπλασιαστές τους ακολούθους και ανθρώπους που ασκούν επιρροή, έτσι ώστε το μήνυμά μας να διαδίδεται. Να σας δώσω μερικά παραδείγματα για να καταλάβετε τι αντίκτυπο έχουν κάποιες από τις έρευνές μας. Για παράδειγμα, ομάδες εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με τις δικές μας συστάσεις έχει αναθεωρήσει σε μεγάλο βαθμό τη διαδικασία αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με πιο ε, διαφανή διαδικασία επιλογής, ε, πολιτική για τη σύγκρουση συμφερόντων, εγγραφή στο Μητρό Διαφάνειας ε, για εργαζομένους αυτό, μάλλον αυτοπασχολούμενους και εκπροσώπους οργανώσεων που διορίζονται σε ομάδες εμπειρογνωμόνων. Πρόσβαση στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας. Αυτό το είχε ζητήσει ε, πρώτα μια βελγική ΜΚΟ ε, για να γνωρίζει ε, ποια είναι τα λόμπι που πιέζουν την ευρωπαϊκή έρευνα σε θέματα αμυντικά. Το θέμα ήταν πώς απάντησαν οι αρμόδιες αρχές. Εδώ χρειάζεται βελτίωση ε, και έγινε ε, αυτή η βελτίωση μετά από όσα ζητήσαμε. Ε, πάνω από 800 ασκούμενοι στα ΣΓΕΡ της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης πληρώνονται ανά τον κόσμο στις αντιπροσωπείες μας. Έχουμε βελτιωμένη διαφάνεια στις εμπορικές διαπραγματεύσεις, ο κώδικας διαντολογίας των επιτρόπων έχει ενισχυθεί. Οι διαπραγματεύσεις ε, για τον Brexit είναι ένα παράδειγμα ε, διαπραγματεύσεων με υψηλό επίπεδο διαφάνειας. Έρχομαι τώρα στη στρατηγική δουλειά που κάνουμε. Έχουμε ξεκινήσει πέντε στρατηγικές ε, πρωτοβουλίες και κλείσαμε δύο στρατηγικές έρευνες και πάλι μερικά παραδείγματα. Η προώθηση της αξιοπρέπειας ε, ε, στην εργασία, στην ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση έβγαλε τα κατάλληλα συμπεράσματα και τις βέλτιστες πρακτικές για το πώς να προλαμβάνονται περιπτώσεις παρενόχληση και πώς να αντιμετωπίζονται. Επίσης, η πολυγλωσία θα πρέπει να βοηθηθούν ε, τα θεσμικά ε, όργανα ε, να βρουν μια ισορροπία ανάμεσα στις ανάγκες να σέβονται τη γλωσσική πολυμορφία και την αναγνώριση ότι υπάρχουν περιορισμοί στους πόρους. Ε, βρήκαμε λύσεις στο 81% των περιπτώσεων και 85% στις υποθέσεις δημοσίου συμφέροντος. Ε, αυξάνονται αυτά τα στοιχεία, είναι σημαντικό ε, γιατί όταν συμμορφώνονται στις αποφάσεις αυτές αυτό βοηθάει και το ευρύτερο κοινό. Έρχομαι τώρα στα εσωτερικά θέματα. Είμαστε μια μικρή μονάδα, άρα θα πρέπει να εξακολουθήσουμε να είμαστε δημιουργικοί για να βελτιώνεται η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητά μας. Χωρί να είναι αυτό, μόνο αυτό σκοπός, αλλά επειδή θέλουμε να απελευθερώσουμε όσο γίνεται περισσότερους πόρους για να ενισχύσουμε τη δυνατότητα που έχουμε να κάνουμε έρευνες. Ε, πρώτον, αντιμετωπίζοντα τις ε, καταγγελίες των πολιτών εγκαίρω, και αυτό είναι για μας ύψιστη προτεραιότητα. Ε, ε, να σας παρουσιάσω ορισμένες βελτιώσεις που πετύχαμε το 2018 από την αποτελεσματικότητα. Κλείσαμε περισσότερες υποθέσεις από ποτέ, 534 σε σύγκριση με τις 348 ε, το 2017. Ο μέσος χρόνος διεκπεραίωσης των ερευνών εξακολουθεί να μειώνεται. Το 18 ήταν 255 ημέρες ενώ το 2017 ήταν 266, ενώ το 2016 ήταν 340 ημέρες κλείσαμε 57% όλων των ερευνών εντός εξαμήνου και 18, 88% ε, εντός 18 ε, μήνου, που είναι πέρα από τους στόχους ε, των βασικών δικτών επιδόσεών μας. Το Φεβρουάριο κινήσαμε μια διαδικασία ταχείας διεκπαιρέως, fast track, για αντιμετώπιση των καταγγελιών που έχουν να κάνουν με πρόσβαση σε δεδομένα. Είναι πολύ θετικός ο απολογισμός. Οι αποφάσεις λαμβάνονται τρεις φορές γρηγορότερα από ό,τι στο παρελθόν, κατά μέσο όρο 44 εργάσιμες, ενώ το 16 ήταν κατά μέσο όρο και το 17 134 εργάσιμες. Επίσης, φτάνουμε σε απορρόφηση του προπολογισμού της τάξης του 95,3% και πάλι αύξηση. Ε, εξακολουθούμε να επενδύουμε ε, στην εκπαίδευση που προσφέρουμε, ε, πράγμα που εκτιμά πάρα πολύ το προσωπικό μας. Έχουμε ιδιαίτερα θετικά σχόλια για την υποχρεωτική κατάρτιση ε, σε ό,τι αφορά την πρόληψη ε, της παρενόχλησης και για το προσωπικό και για ε, τους μάνατζερ. Έχουμε τώρα υπαλλήλους δεοντολογίας και επιτροπή συνδιαλλαγής. Τέλος, εξακολουθούμε να ψάχνουμε τρόπο να ενισχύσουμε την οικονομική μας αποτελεσματικότητα. Όπως επανέλαβα, είμαστε μικροί ως θεσμός, αλλά χρησιμοποιούμε ε, πολλά ε, εργαλεία, συμβάσεις, υπηρεσίες και ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Ε, το 2018 ε, εγκρίναμε το MIPS που είναι το εργαλείο που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διαχειρίζεται τις αποστολές. Ε, θέλουμε να μειώσουμε επιπλέον τα έξοδα για τη μετάφραση μέσω περαιτέρω διοργανικής συνεργασίας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω τώρα ή αργότερα σε κάποιες ερωτήσεις σας. Αν θέλετε να σας δώσουμε και άλλα στοιχεία μετά το τέλος συνεδρίας. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ ακριβή τα στοιχεία που μας δώσατε. Και τώρα τελευταίος κατά σειρά είναι ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων. Ο κύριος Λεωνάρντο Σεβέρα Νάβας. Παρακαλώ. Thank you, Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε που μας δώσατε την ευκαιρία να πάρουμε το λόγο ενώπιόν σας εκπροσωπώντας τον επόπτη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η Μάριαν και ο Κιμ ε, εδώ θα με βοηθήσουν να κάνω ό,τι μπορώ για να απαντήσω τις δικές σας ερωτήσεις να σας πω πως ε, στο λίγο χρόνο που έχουμε μπορώ να πω δύο λόγια για την εντολή του δικού μας, ε, της δικής μικρής μας ε, υπηρεσίας και για τις προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε το 2018 και θα μιλήσω και για την συνέχεια που δώσαμε στην απόφαση απαλλαγής για το 2017. Το 2018 εμείς μεγαλώσαμε γιατί μας ανατέθηκαν όλο και περισσότερα καθήκοντα και η προστασία των δεδομένων απέκτησε και μεγαλύτερη σημασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και εκτός. Είμαστε ακόμα το μικρότερο όργανο. Έχουμε μόνο 87 άτομα προσωπικό το 2018 με προϋπολογισμό μόλις 14,5 εκατομμύρια ε, που διαφέρει πολύ από τα 9 δις που κάποιος ε, ανέφερε ως διοικητική δαπάνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα βασικά μας καθήκοντα είναι η εποπτεία της διαδικασίας προστασίας και διαχείρισης προσωπικών δεδομένων από ευρωπαϊκούς θεσμούς και όργανα. Κάνουμε καταρχήν λοιπόν έρευνες και επιθεωρήσεις, μερικές φορές αυταπαγγέλτος και μερικές φορές λόγω ε, καταγγελιών και το κάνουμε και ε, εμείς από την πλευρά μας για να αυξήσουμε ε, την ε, αναγνωρισιμότητα και την ευαισθητοποίηση για τα θέματα αυτά, παρακολουθώντας τις εξελίξεις ε, με ένα δικό μας ενεργό τρόπο. Έχουμε λοιπόν και τους ομολόγους μας της προστασίας προσωπικών δεδομένων στα άλλα όργανα, με τους οποίους είμαστε με, συνεχή, σε συνεχή επαφή. Από το 2017 και, και μετά καλύπτουμε την Eurojust, τη Europol, όπως επίσης και το Γραφείο της Ευρωπαϊκής Συγκέντρωσης Θέλουμε λοιπόν να έχουμε ισχυρή πολιτική προστασίας δεδομένων στα ευρωπαϊκά όργανα και δεύτερον ε, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να βοηθήσουμε τον νομοθέτη στη χάραξη πολιτικής προσφέρουμε με επίσημα και ανεπίσημα σχόλια συμβουλές και πολλές φορές μας καλούν τα δικαστήρια να παρέμβουμε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, είναι πολύ εξοικειωμένο με, τη δική μας, με τις δικές μας συμβουλές και είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες για την εκτίμηση της οποίας χαίρουμε εδώ και κυρίως ε, στο πόσο η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ Ελευθεριών ε, σέβεται ε, τις δικές μας συστάσεις. Συνεργαζόμαστε και με άλλους διεθνείς αντίστοιχους οργανισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων, είτε μας αρέσει όχι, τα προσωπικά μας δεδομένα φεύγουν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, φτάνουν πολύ μακριά και είναι σημαντικό αυτά να προστατεύονται και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τέλος, και μετά την ε, υπογραφή και την εφαρμογή του ε, GDPR, του κανονισμού αυτού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, παρακολουθούμε να υπάρχει ομοιόμορφη και ενιαία προστασία των δεδομένων αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, ποιε είναι οι βασικέ προκλήσει για το 2018. Να σα πω πω το 18 χρονιά ήταν μια χρονιά πολύ διαφορετική από όλε τι άλλε λόγω της ε, ε, έγκρισης του κανονισμού για την προστασία των δεδομένων ήταν η χρονιά των προσωπικών δεδομένων. Μεγάλη πρόκληση για μας. Σας είπα, είμαστε ο μικρότερος ε, θεσμός και χρειάστηκε να ανδρωθούμε ε, με έναν τρόπο δύσκολο, μεγάλο το έργο, το κάναμε επιτυχημένα μπορώ να πω. Και ο Τζοβάνι Βουταρέλη που είναι ο υπόπτης μας και ο οποίος δυστυχώς ε, πέθανε πέρσι το καλοκαίρι, ήταν ο μεγάλος ηγέτης ο οποίος οργάνωσε μια διεθνή διάσκεψη για την, ε, για την προστασία των δεδομένων με τους εξηματούχους για το θέμα αυτό, με πάνω από χίλιους προσκεκλημένους από παντού στον κόσμο που ήρθαν εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τεράστια πρόσκληση, επαναλαμβάνω, για ένα τόσο μικρό θεσμό όπως εμείς. Και το κάναμε ε, για να ε, ε, παγιώσουμε την ηγετική θέση που έχει η Ευρώπη στην προστασία των δεδομένων. Σαν να μην έφτανε αυτό το Δεκέμβριο. Παρουσιάστηκε και ένας νέος κανονισμός που εφαρμόζεται στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και υπηρεσίες και χρειάστηκε όλοι να ε, προσαρμόσουμε τις διαδικασίες μας σε αυτή τη νέα νομοθεσία. Και πρέπει να πω από τις πολλές αλλαγές που έγιναν, περάσαμε από τους δύο επόπτες σε έναν, από την 5η Δεκεμβρίου του 2018. Κάτι πολύ σχετικό, γιατί τώρα εσείς πρόκειται να διορίσετε το νέο υπόπτη. Και είναι σημαντικό το άτομο που θα επιλέξετε να γνωρίζει το πώς ε, λειτουργούν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Όταν θα διορίσουν τον επικεφαλής της, υπηρεσία μας. 91,5% έχουμε ε, εκτέλεση προϋπολογισμού. Καλώς είναι, γιατί είχαμε πολλά στοιχεία αβεβαιότητας και για το τελευταίο σημείο που είναι η απαλλαγή και την απόφαση και το, τη συνέχεια που δόθηκε. Έχετε την έκθεσή μας, θα ήθελα απλώς να τονίσω πως το να είναι κανείς μικρός είναι δύσκολο. είναι δύσκολο να εφαρμόσουμε όλες τις συστάσεις και κυρίως αυτές που είναι σχετικές με την ισότιμη εκπροσώπηση εθνικοτήτων όταν είμαστε όλοι όλοι 80, το να έχουμε και από τα 27 κράτη-μέλη εκπροσώπους είναι δύσκολο. Θα κάνουμε όμως ό,τι μπορούμε για να ακολουθήσουμε αυτές τις συστάσεις και είμαστε πολύ χαρούμενοι που το ελεγκτικό συνέδριο δεν ανέφερε βρήματα για την αξιοπιστία των λογαριασμών μας και για να κλείσω θα σας πω πως παρόλο που είμαστε πάρα πολύ μικροί και έχουμε το μικρότερο προϋπολογισμό, εμείς τις δημοσιονομικές μας υποχρεώσεις τις λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη και χαιρόμαστε πάρα πολύ για το ότι συνεχίζετε να μας στηρίζετε ε, εμάς και όλους τους συναδέλφους που εργάζονται στον χώρο της προστασίας προσωπικών δεδομένων στην Ευρώπη. Θα απαντήσω με χαρά στις ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Και εμείς ε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ε, περιστατωμένες οι εισηγήσεις σας ε, και να δώσω τώρα το λόγο στον εισηγητή μας ε, για να κάνει τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο ακριβής και αντικειμενικός γίνεται. Αλλά θα είμαι και αυστηρός. Και σε κάποιες ερωτήσεις που θα κάνω ε, θα είμαι ε, πιο αναλυτικός, κυρίως ε, θα αφορούν οι ερωτήσεις αυτές θέματα όπου δεν ήσασταν σαφείς. Η Επιτροπή αυτή έχει μία σχέση με τους άλλους θεσμούς που ήταν πάντα πολύ καλή, τουλάχιστον όσο είμαι εγώ Ευρωβουλευτή στο Κοινοβούλιο και ελπίζω αυτό να παραμείνει και στο μέλλον. Ξεκινάω με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και εδώ νομίζω ότι εκφράζω την άποψη των περισσότερων μελών της Επιτροπής. Υπάρχει κάτι που δεν μας αρέσει και αυτό αφορά στο ότι εδώ και εννέα χρόνια δεν μπορούμε να δώσουμε απαλλαγή στο Συμβούλιο γιατί το Συμβούλιο δεν συνεργάζεται μαζί μας ε, και δεν μας δίδει τις ε, πληροφορίες που επιθυμούμε. Σήμερα ε, ούτε καν ήρθε ο Γενικός Γραμματέας υπόψη όλων, προς υπόψη όλων. Εμείς θέλουμε ε, μία λύση ε, η οποία θα μας επιτρέψει να λάβουμε μία σωστή απόφαση ε, με βάση τεκμηριωμένες πληροφορίες. Χαιρετίζω αυτά που είπαν οι κυρίες Γιώροβα και Χάν κατά την ακρόαση είπαν ότι είναι πρόθυμες να εξετάσουν αυτό το πρόβλημα ε, και να ε, προσφέρουν μεγαλύτερη διαφάνεια στις συζητήσεις του ε, Συμβουλίου για τον προϋπολογισμό. Θέλουμε όμως να γνωρίζουμε πώς ακριβώς το Συμβούλιο εφαρμόζει τον προϋπολογισμό και μέχρι ποιου βαθμού. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να σας πω ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις έχουν ήδη ξεκινήσει και ελπίζω το στομό των ετών να καταλήξουμε σε συμπέρασμα. Και τώρα, σε άλλους μεμονωμένους θεσμούς, όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ε, χαίρομαι πάρα πολύ που φέρατε και τη συνάδελφό σας και την καλωσορίζω θερμά. Τρεις πολύ σύντομες ερωτήσεις. Η ε, ασφάλεια και η ταχύτητα των ε, ροών της πληροφορικής είναι πολύ σημαντικές και ερωτώ, έχετε επιτύχει βελτίωση όσον αφορά την App ή Κούρια και τι ακριβώς ε, συμβαίνει με την, ε, το ολοκληρωμένο management του φάλων που ε, συνεργάζεται στενά με την Ικούρια και αυτό το συστήσαμε και το συστήνει μια ειδική έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Επίσης, διαπιστώνουμε ότι χρειαζόμαστε σαφείς κανόνες για να μπορούμε να διασφαλίσουμε την ισότητα των ευκαιριών. Και ερωτώ το ε, συνέδριο έχει ασχοληθεί με τους κανόνες περί υποστήριξης. Είναι οι κανόνες που αφορούν τους χρηματοδότες. Είπατε επίσης ότι το 2018 είχατε 274 ασκούμενους, αλλά μόνο λίγοι εξ αυτών πήραν χρήματα για την πρακτική τους άσκηση. Είπατε ότι το 2018 αναθεωρήσατε και μεταρρυθμίσατε το σύστημα των ασκούμενων, ότι θέλετε να χρηματοδοτείτε περισσότερους, αλλά εξακολουθείτε να προσφέρετε πολλές ε, θέσεις ε, πρακτικής εξάσκησης χωρίς χρηματοδότηση. Γι' αυτό ερωτώ το συνέδριο, τι θα κάνει στο μέλλον ή ε, όσον αφορά στο μέσο ποσό, το οποίο δίνει το ελεγκτικό συνέδριο στους ασκούμενους ως αμοιβή. Με αυτό τι θα γίνει. Επίσης, ε, σας συγχαίρω, ελεγκτικό συνέδριο, ότι ασχολείστε με, το, με τον ηθικό κώδικα και το ηθικό πλαίσιο όσον αφορά τις σεξουαλικές ε, παρενοχλήσεις ε, και τον εκφοβισμό. Εδώ βέβαια θα ήθελα να κάνω και μία ερώτηση προς το ελεγκτικό συνέδριο. Γνωρίζουμε όλοι ότι η Όλαφ διεξάγει έρευνες και την τελευταία χρονιά έστειλε μία έκθεση. Πρόκειται για παρατυπίες εκ μέρους που αφορούν σε ένα μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου. Αυτές οι παρατυπίες αφορούν κάποιες διοικητικές διαδικασίες. Ερωτώ λοιπόν με αυτές τις ε, περιπτώσεις ε, τι ακριβώς θα γίνει, τι ακριβώς κάνει το ελεγκτικό συνέδριο για να παρεμποδίσει παρεμφερείς ε, περιπτώσεις. Και επίσης θέλω να ερωτήσω τι θέλει να κάνει το συνέδριο πολύ συγκεκριμένα για να εμποδίζει να υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Ε, χαίρομαι που έχετε αυξήσει το σύστημα των ψηφιακών ελέγχων και χαίρομαι που ο Γενικός Γραμματέας πρόκειται να εγκρίνει ε, τις ε, δαπάνες αποστολών για τα μέλη του ελεγκτικού συνεδρίου. Σημαίνει άραγε αυτό ότι αυτές οι δαπάνες θα ελέγχονται τώρα με την ίδια ακρίβεια όπως και άλλες δαπάνες. Και τώρα, όσον αφορά τις έρευνες για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Πρόκειται για τον ε, έλεγχο ε, των δαπανών ταξιδιών ε, κάποιων μελών του ελεγκτικού συνεδρίου ε, πρόκειται επίσης για τον ε, στόλο αυτοκινήτων του ελεγκτικού συνεδρίου και τη χρήση αυτού του στόλου. Νομίζω αυτό ήταν μια σημαντική πρόοδος του ετήσιου προγράμματος και θέλω να ρωτήσω τι ακριβώς έχει γίνει σε αυτή την περίπτωση. Υπάρχουν άραγε κάποια ε, αποτελέσματα που μπορείτε να μας ανακοινώσετε όσον αφορά τον στόλο αυτοκινήτων του ελεγκτικού συνεδρίου. Χαιρόμαστε ε, που έχει τεθεί κάποιο ανώτατο όριο στις ε, πληρωμές και το ανώτατο αυτό όριο τώρα πλέον ε, είναι χαμηλότερο. Παλαιότερα το ανώτατο ήταν 15.000 χιλιόμετρα, τώρα είναι 10.000 χιλιόμετρα. Έχετε όμως και άλλες διατάξεις που να αφορούν στη χρήση αυτού του στόλου αυτοκινήτων. Και τελευταία ερώτηση για το ελεγκτικό συνέδριο. Χαίρομαι που το ελεκτικό συνέδριο δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του ε, τις ε, ε, δηλώσεις οικονομικού συμφέροντος των μελών και αυτές τις δηλώσεις μπορεί να τις ελέγξει η κοινή γνώμη, όποιος επιτιμεί. Όμως Μήπως ε, προτίθεστε να βελτιώσετε περαιτέρω αυτές τις δηλώσεις οικονομικού συμφέροντος των μελών σας. Περνάμε τώρα στην ε, Επιτροπή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και χαίρομαι για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε πάρα πολλούς ε, τομείς εντάθηκε η παρουσία σας, έχει γίνει πιο ορατή. Θα μπορούσατε να γίνετε πολύ καλό παράδειγμα προς μίμηση για άλλους θεσμούς. Και η Επιτροπή των Περιφερειών και αυτή τα τελευταία δύο χρόνια ε, είναι πιο ορατή και αυτό το χαιρετίζω. Ε, κάποιες ερωτήσεις. Το 2018 υπήρξαν ε, κάποιες περιπτώσεις παρενόχλησης στον χώρο εργασίας. Στον ηθικό κώδικα, στον κώδικα συμπεριφοράς, έχετε κάνει κάποιες αλλαγές που να αφορούν στα μέλη. Επίσης, από ό,τι φαίνεται, έχετε περιορίσει τον αριθμό των ανθρώπων που προσέρχονται σε συνεδριάσεις και ρωτώ την ε, στρατηγική σας σφιγμομετρήσεων τι αναθεωρήσατε, πού ακριβώς επιτύχατε περικοπές και εξοικονόμηση. Και άλλη μια ερώτηση ε, προς αυτή την Επιτροπή. Έχετε περιγράψει τη διαδικασία επιλογής του Γενικού Γραμματέα και υπάρχουν πληροφορίες ότι λόγω αυτής της ε, επιλογής έχετε επιβεβαιώσει ε, κάποιες αιτήσει για ενημέρωση. Και λέτε επίσης ότι ε, κανείς δεν έχει διαμαρτυρηθεί για τη διαδικασία επιλογής. Όμως παρόλα αυτά ερωτώ, δεν θέλετε να αναθεωρήσετε το, ε, τη διαδικασία επιλογής ε, του Γενικού Γραμματέα. Παραδείγματο χάρη στη διαδικασία αυτή θα μπορούσε να συμμετέχει και ένα ανεξάρτητο μέλος. επιπλέον. Όταν συμμετέχει κάποιος που είχε σημαντική θέση στην Επιτροπή, ο συγκεκριμένος αυτός άνθρωπος αποκλείται αυτόματα από τη διαδικασία. Νομίζω ότι αν κάνετε κάποιες μεταρρυθμίσεις ε, θα βελτιωθεί η διαφάνεια της διαδικασίας επιλογής. Τελευταία ερώτηση αφορά στην ε, διοικητική συνεργασία ανάμεσα στη δική σας την Επιτροπή και την Επιτροπή των ε, Περιφερειών. Έχετε κάποιες βελτιώσεις, ανέπιες ναι, και τι είδου πρόοδο περιμένετε αν τελικά προκύψει μια νέα συμφωνία. Στην Επιτροπή των περιφερειών. Θέλω να ε, καλωσορίσω τον κύριο Μαρτίνες. Αυτή τη στιγμή έχει την ε, θέση ε, του μεταβατικού γενικού γραμματέα, του εκτελούντος χρέη και χαιρετίζω κατά πάσα τον μελλοντικό γενικό γραμματέα αυτής της Επίτροπης. Και περνάω σε ένα θέμα που μας απασχόλησε πάρα πολύ κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απαλλαγής των τελευταίων ετών. Επρόκειτο για μία περίπτωση όπου ε, την επισημαίνει την περίπτωση αυτή ο πρώην εσωτερικός ελεγκτής. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Επιτροπή ε, δέχτηκε την πρόταση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ε, αμελητή Τέτοιο ερώτημα κατά πόσον θα ε, προκύψει μια νέα επιτροπή για την ε, αναπηρία. Ε, συστήθηκε αυτή η επιτροπή και αποφάνθηκε ότι η ασθένεια του πρώην εσωτερικού ελεγκτή ανάγεται αδιαμφισβήτητα στην άσκηση των καθηκόντων του. Εγώ λοιπόν ρωτώ τελικά τι θα γίνει πώς θα το αντιμετωπίσει το θέμα η Επιτροπή των Περιφερειών, γιατί θέλουμε να κλείσει αυτή η υπόθεση το συντομότερο δυνατόν όλοι έχουμε καταλάβει πόσο ε, σημαντικά ήταν όλα αυτά που έκανε ο εσωτερικό ελεγκτής γιατί μας ενημέρωσε για αδυναμίες αλλά πραγματικά αυτή η περίπτωση ε, τραβάει χρονικά πάρα πολύ και ε, νομίζω ότι θα ήταν λάθος πριν από την απαλλαγή του 2019 να ασχοληθούμε και πάλι με την ίδια περίπτωση. Υπάρχει και το θέμα της παρενόχλησης ενός μέλους. Η διαμεσολαβήτρια ε, πρότεινε να υιοθετήσουμε κάποιους ε, κανόνες ε, που ανάγονται βέβαια σε αποφάσεις του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρόκειται και πάλι για περιπτώσεις παρενόχλησης και ρωτώ τι ακριβώς επιτύχατε και μετά η εκστρατεία για το μέλλον της Ευρώπης. Οργανώστε περίπου 200 εκδηλώσεις. Σε αυτές τις εκδηλώσεις συμμετείχαν πολλά μέλη. Μπορείτε λοιπόν να μας περιγράψετε τα αποτελέσματα αυτών των εκδηλώσεων. Τι έφεραν συγκεκριμένα, τι δεν έφεραν, πόσοι συμμετείχαν σε αυτές τις εκδηλώσεις, πόσοι εργαζόμενοι και θα ήθελα επίσης να γνωρίζω κατά πόσον τα κονδύλια, τα χρήματα που δαπανίζονται για αυτές τις δαπάνες τεκμηριώνονται ως δαπάνες. Και τέλος, στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Σας συγχαίρω γιατί αυτός είναι ο μόνος θεσμός ο οποίος περιέκοψε τον προπολογισμό του σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, κατά περίπου 70.000 ευρώ. Όμως ε, το ε, Κοινοβούλιο ε, θέλει να ληφθούν υπόψη και νέες εξελίξεις, νέα γεγονότα. Το 2008 υπήρξε μία μεταρρύθμιση και τώρα έχει υπάρξει και άλλη μία. μπορείτε λιγάκι να μας την περιγράψετε, γιατί πρόκειται κυρίως για τα καθήκοντα, το προσωπικό και τον προεπολογισμό. Αυτό που μου άρεσε ήταν η ε, παρουσίαση των ε, εργασιών του Ευρωπαίου ε, Επόπτη στην ιστοσελίδα που χωρίζονται σε διάφορα κεφάλαια, διαφάνεια, ηθική και πολλά άλλα. Και βεβαίως Υπάρχουν εκεί και πάρα πολλές ε, σελίδες, αλλά γιατί δεν προβλέπετε και ένα κεφάλαιο για τις, ε, τους εσωτερικούς κανόνες. Ε, θα μπορούσε να είναι ένα είδος ηθικού πλαισίου. Σας ερωτώ λοιπόν τι ακριβώς προτίθεστε να κάνετε από αυτού σε σχέση με όλα αυτά που ανέφερα και κυρία Πρόεδρε τελειώνω σιγά σιγά αλλά θέλω να σας πω ότι υπάρχουν ε, πάρα πολλοί θεσμοί, 7 είναι αυτοί που ήρθαν εδώ ε, και γι' αυτό και εγώ χρειάστηκα περισσότερο χρόνο. Ήθελα λοιπόν ε, σε κάποιες ερωτήσεις να είμαι λίγο πιο διεξοδικός, πιο αναλυτικός, ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων. Το 2018 ήταν πολύ σημαντική χρονιά γι' αυτόν λόγω του PDPA. λόγω του GDPR, με συγχωρείτε. GDPR, α ναι, για την οδηγία περί προστασίας δεδομένων. Και θα ήθελα επίσης να γνωρίζω ε, ο Ευρωπαίος ε, επόπτης πώς ακριβώς ελέγχει την εφαρμογή των κανόνων και τι είδους επιπτώσεις έχουν όλα αυτά στο προσωπικό και στην, ε, στα προσόντα του προσωπικού. Γνωρίζω παραδείγματο χάρη ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτύχουμε την ισορροπία ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες και αυτό σε ένα θεσμό που είναι αρκετά περιορισμένος. Θα ήθελα λοιπόν ε, να ρωτήσω, εσείς έχετε στρατηγική περισσότερες των δύο φίλων που να την εφαρμόζετε, γιατί αυτό το είχατε πει την προηγούμενη χρονιά και τελικά τους στόχους αυτής της στρατηγικής τους επιτυγχάρετε ή όχι. Αγαπητοί συνάλφοι, χαίρομαι πάρα πολύ για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει, χαίρομαι που θα μου δώσετε απαντήσεις σε ερωτήσεις μου και λυπάμαι πάρα πολύ που μακρηγόρησα, αλλά ε, ίσως... Ε, ε, κάποιες ερωτήσεις που ετέθησαν ε, να είναι σημαντικές για τους αδέλφους. Ε, χαίρομαι για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Εσείς είπατε ότι ήρθατε εδώ για να μας ακούσετε και εμείς όμως ακριβώς έτσι το βλέπουμε. Εμείς οι βουλευτές είμαστε εδώ για να ακούσουμε εσάς, τις απόψεις σας, να σας βοηθήσουμε στη δουλειά σας που την εκτιμούμε τόσο πολύ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σδεχόφσκι. αφήσατε και καμιά ερώτηση για τους άλλους, τους και συγγητές. Τα είπατε όλα. Για να δούμε τι έχουν να πούν οι σκιώδεις πρώτα και μετά ε, ε, να απαντήσουν οι θεσμοί. Θα δώσω το λόγο στον εαυτό μου, γιατί είμαι σκιώδης εισηγήτρια των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Και το πρώτο που θέλω να κάνω είναι γενικά σχόλια για όλους τους ε, θεσμούς. Στην απαλλαγή του 2018 διαπίστωσα ότι έγιναν πρόοδοι ε, και θετικά βήματα σε όλα τα θεσμικά όργανα, όπως είναι η ευαισθητοποίηση στην παρενόχληση, η ενδεχόμενη σύγκρουση φερόντων, η προστασία των ε, καταγγελόντων. Όλα αυτά βοηθούν και συστηματοποιούν και δρεώνουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Ε, είχα κάποιες ερωτήσεις να κάνω, απάντησαν όμως ήδη Γενική Γραμματής, γι' αυτό δεν θα μακρηγορήσω τόσο όσο ο κύριος Δεχόφσκι. Παρόλο που είπε στην αρχή ότι δεν θα μακρηγορήσει και ζήτησε το, το πρωί από εμά να είμαστε σύντομοι. Ε, σε ό,τι αφορά το Συμβούλιο, συμφωνώ με τον κύριο εισηγητή Οπότε δεν πρόκειται να σχολιάσω τίποτα παραπάνω. Ε, για το δεύτερο θεσμικό όργανο που είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Μου φάνηκε ενδιαφέρον αυτό που άκουσα, ότι είναι το πρώτο θεσμικό όργανο που έχει κάνει ε, ε, τα open space γραφεία ατομικά μετά από ένα ερωτηματολόγιο που είχε κυκλοφορήσει. Τι ήταν αυτό που σας οδήγησε τα open space να τα ξανακάνετε ατομικά γραφεία. Είχατε χρόνο να εκτιμήσετε αν επέφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα. 1.120 ευρώ παίρνουν οι υπότροφοι στα ΣΓΕΡ στο Λουξεμβούργο. Φτάνουν αυτά τα λεφτά για το Λουξεμβούργο. Για μια αξιοπρεπή διαβίωση. Για ποιο λόγο ε, δεν ε, δημοσιεύει τις, το πόθεν και στο μελόν του το δικαστήριο ενώ το κάνουν τα άλλα ε, ευρωπαϊκά όργανα. Πηγαίνω στο ελεγκτικό συνέδριο. Τι γίνεται με την έρευνα του μέλους του ελεγκτικού συνεδρίου που βγήκε στη δημοσιότητα το 2017 για την ισομερή εκπροσώπηση. Λέει ο Γενικός Γραμματέας ότι εργάζεστε προς την κατεύθυνση της βελτίωσης. τι μέτρα λαμβάνετε. Τι κάνει το ελεγκτικό συνέδριο για να προσελκύει ε, νέους υπαλλήλου και τελευταίο με πόσα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια έχετε συνάψει συμφωνίες ε, για να τους ε, εκπαιδεύετε τους φοιτητές σε θέματα ελέγχου των ευρωπαϊκών οικονομικών. Τώρα έχω ερωτήσεις για την Επιτροπή των Περιφερειών και για την ΟΚΕ μαζί. Βάσει του Συμφώνου Συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2018. Το Κοινοβούλιο, όπως και τα άλλα χρόνια, έχει δώσει επιπλέον μεταφραστές ε, γιατί έτσι αντισταθμίζεται η μείωση του προσωπικού της μετάφρασης της ΟΚΕ και της Επιτροπής των Περιφερειών. Πώς αξιολογούν αυτή την ιδιάζουσα κατάσταση και οι δύο γενικοί ε, γραμματείς. Στη συμφωνία με το Κοινοβούλιο. Αυτή, αυτή υπογράφηκε το 2016 και εκπνέει τέλη του έτους. Τουλάχιστον στα χαρτιά είναι ενθουσιασμένα και τα δύο αυτά θεσμικά όργανα, οι δύο επιτροπές. Γιατί όμως δεν υπάρχουν ποσοτικά στοιχεία, πόσες οικονομίες έχετε κάνει μετά από τη συμφωνία αυτή. Έχει ληφθεί καμιά απόφαση για την ανανέωση του συμφώνου αυτού. Σε ό,τι αφορά τη συμφωνία που υπεγράφει το περασμένο Αύγουστο, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ανταλλαγή κτηρίων. Θεωρείτε ότι τα αποτελέσματα αυτά της επιμελητίας ε, αποζημιώνουν την οικονομική απώλεια. Αναφέρονται και ε, τα δύο θεσμικά οργανά για το χώρο εργασίας του μέλλοντος. Τι είναι αυτό το workplace of the future, τι εννοείται. Και μια ερώτηση συγκεκριμένα για την ΟΚΕ. Έχετε πρόθεση να διευρύνετε την εκπαίδευση για την πρόληψη της παρενόχλησης στο χώρο εργασίας στα μέλη της ΟΚΕ και μια ειδική ερώτηση δεν είναι ακριβώς ερώτηση για την Επιτροπή των Περιφερειών θα ήθελα να σας ρωτήσω για την υπόθεση Μακόη αλλά σήμερα λάβαμε μια επιστολή που έλεγε ότι η πρώτη συνεδρίαση της ε, συνδιαλλαγής συμφιλίωσης θα γίνει στις 4 Δεκεμβρίου. Να περιμένουμε να δούμε τι θα βγει από τη συνεδρίαση αυτή. Και έρχομαι τώρα στην Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια. Η συμβασιούχοι είναι το 20% του προσωπικού του θεσμικού οργάνου σας. Και συνταξιούχοι καλύπτουν πάγιες ανάγκες όμως. Υπάρχει καμιά δυνατότητα να βελτιωθεί ο τύπος τη σύμβαση του προσωπικού αυτού που είναι όλο και πιο μόνιμο. Φαντάζομαι γνωρίζετε τα mail που έχουμε λάβει πολλοί βουλευτές με ε, ρητές ε, κατηγορίες που στρέφονται κατά της κυρίας Οράιλη, της διαμεσολαβήτριας ε, θεωρείτε σκόπιμο να δώσετε καμία εξήγηση. Νομίζω προσφέρεται εδώ η ευκαιρία αυτή. Και τέλος, τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Το 40% του προσωπικού σας είναι συμβασιούχοι. Για ποιο λόγο δεν ανησυχείτε ε, από την ε, επισφάλεια την εργασιακή αυτών των εργαζομένων και θα χάνετε και τεχνογνωσία και εμπειρογνωμοσύνη. Γιατί όταν εκπνέει η εξαετία των συμβασιούχων θα πρέπει να επενδύεται ξανά σε εκπαίδευση νέου προσωπικού. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου. Και να περάσουμε τώρα στον κύριο Πέξα. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα καταρχήν να σας πω πως μου δώσατε την ευκαιρία να κάνω ερωτήσεις και γι' αυτό σας ευχαριστώ. Ε, πραγματικά ε, είναι μια μεγάλη ευκαιρία και θα ξεκινήσω με την πιο συγκεκριμένη ερώτηση, η οποία είναι η εξής. Ε, στρέφομαι προς το 10. Μιλώ για το για τις προσλήψεις προσωπικού και επίσης για τα προβλήματα προϋπολογισμού που α, αντιμετωπίζετε. Τι σκοπούς έχετε <coughs> και ποια είναι η διάρκεια μιας υπόθεσης η οποία φτάνει στο ΔΕΚ. Ποια είναι η τάση για το πόσο χρόνο χρειάζεται για την τραπ... Για την ΕΤΕ λοιπόν, ε, τι συνέβη. Με ποιο τρόπο επενδύει τα ευρωπαϊκά χρήματα. Ε, ε, Και έχω ακόμα μια γενική ερώτηση. για την εξοικονόμηση πόρων στο διοικητικό επίπεδο. Ε, για παράδειγμα, εξοπλισμός, γραφείου κτλ. χαρτικά. Υπάρχει τρόπος να μειωθούν οι δαπάνες σας αυτές. Επίσης για τη μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου, μήπως λιγότερα ευρωπαϊκά ταξίδια. Ε, αυτό θα μείωνε και τις ε, ταξιδιωτικές δαπάνες και τα οδηπορικά. Αυτά αφήνω χρόνο για να κάνουν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Κούς, τι Ο κύριος Κούτς έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω άλλες ερωτήσεις. Καλύφθηκα. Ευχαριστώ πολύ. Pues entonces pasamos a la señora Η κυρία Πέκοβα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Μία ερώτηση σε σχέση με τα όσα συζητούσαμε. Ε, κόστος ε, μεταφορών και απευθύνομαι προς την Ευρωπαϊκή ΟΚΕ. Επειδή έχει να κάνει αυτό με την βελτιστοποίηση του κόστους, πώς μπορείτε εσείς να κάνετε μία πρόβλεψη για το ενδεχόμενο κόστος έτσι ώστε η δαπάνη να είναι η χαμηλότερη δυνατόν. Δηλαδή πώς εξασφαλίζετε τη σχέση κόστους ωφέλους σε αυτή τη γραμμή προπολογισμού. Λοιπόν, ας ακούσουμε τις απαντήσεις. Θα δίνω εγώ το λόγο σε καθέναν από εσά έτσι ώστε να έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε. Να περάσουμε λοιπόν από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταρχήν. Ε, Ευχαριστώ, κύριε Γκαρθία Μουνιό. Ας αρχίσουμε από τις ερωτήσεις που έκανε ο εισηγητής. Τρεις ερωτήσεις έκανε για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η πρώτη αφορά την ταχύτητα στην επικοινωνία και στις βελτιώσεις ε, στη, ε, ως προς το χαρτί και τα έγγραφα με την ηλεκτρονική εφαρμογή ή κούρια και το σύστημα το ολοκληρωμένο διαχείρισης. Ε, το βασικό στοιχείο το είπα στην αρχή. Ποιο είναι ε, η εφαρμογή αυτή ή κούρια που είναι ένα σύστημα πληροφορικής για ανταλλαγή ε, εγγράφων μεταξύ των γραμματέων ε, των διαφόρων δικαιοδοτικών οργάνων. Ε, από τη μια δηλαδή έχουμε υποβολή των εγγράφων και ταυτοποίησή τους. Από την 1η Δεκεμβρίου 2018 είναι υποχρεωτική αυτή η εφαρμογή στο δικαστήριο και είναι και σημαντική πρόοδος διότι η χρησιμοποίηση αυτής της πλατφόρμας την οποία κατά τα άλλα καλωσόρισαν και τον υποχρεωτικό χαρακτήρα ε, το Συμβούλιο και οι εκπρόσωποι των κρατών μελών. Ε, τώρα έχουμε μια πιο άμεση ανταλλαγή εγγράφων. Ε, μπορούμε να εξοικονομήσουμε φυσικά και χαρτί με πολύ θετικό αντίκτυπο και δημοσιονομικό αλλά και περιβαλλοντικό και ε, ελαφρύνεται και ο διοικητικός φόρτος για τη ε, γραμματεία μας ε, που έχει να χειριστεί ένα πολύ μεγάλο όγκο χαρτιών και να το κωδικοποιεί κάθε φορά. Λοιπόν, έχει βελτιωθεί το σύστημα και χρησιμοποιείται και με τρόπο πιο εντατικό. Ε, στο έχει στόχο να αντικαταστηθεί από το ενιαίο σύστημα ε, διαχείρισης των υποθέσεων που είναι ευρύτερο από το σημερινό γιατί εκεί θα ενταχθούν και εργαλεία παρακολούθησης των υποθέσεων όχι μόνο μια ηλεκτρονική πλατφόρμα ανταλλαγών και καταρχήν θα είναι μια δικτυακή πύλη ε, για τα ε, μέρη που ενέχονται στη δίκη. Στη συνέχεια, τα μέτρα που λαμβάνουμε ε, για την ισότητα ε, σε χορηγίες, sponsoring. Ε, εμείς δεν κάνουμε τέτοιες χορηγίες για κάποια γεγονότα, εκδηλώσεις, γι' αυτό δεν έχουμε και αντίστοιχου κανόνες. Η ε, τρίτη ερώτηση ε, είχε να κάνει με τις έμιστες ή άμιστες θέσεις ε, άσκησης. Το 2018 ελήφθη όμως μια νέα απόφαση για ένα νέο καθεστώς πρακτικής άσκησης και προβλέπονται και έμιστες θέσεις που στο παρελθόν δεν ε, ε, σε, σε γραφεία που δεν υπήρχαν παλαιότερα. Οπότε έχουμε ε, και στα γραφεία των δικαστών και στο μέλλον θα αυξηθούν οι έμιστες θέσεις περισσότερο από ό,τι ε, το 2018. Ε, είναι γεγονός ότι προβλέπονται ακόμα από την απόφαση αυτή ε, θέσεις άμυστες πρακτικής άσκησης στα γραφεία των δικαστών, αλλά θέλουμε να διατηρηθεί ακόμα αυτή η δυνατότητα γιατί πολλές φορές οι ασκούμενοι έχουν υποτροφία. γιατί υπάρχουν και κάποιες διατάξει διατάξεις διαδικαστικού χαρακτήρα που αφορούν την πρόσβαση ε, και το οποίο δικαιούται να υποβάλει υποψηφιότητα με πολύ συγκεκριμένες ε, διάρκειες. Ε, Αυτό το σύστημα στο μέλλον θα παραμείνει όμως να είναι στην μειοψηφία παρά στην πλειονότητα των θέσεων. ερώτηση των σχεδόν εισηγητών, ε, τη σκιώδου εισηγήτρια, για το open space που ρωτήσατε για στους χώρους εργασίας. Ε, μία υπηρεσία, ε, η Διεύθυνση Τεχνολογίας Πληροφορίας, ενδιαφέρθηκε ε, στην αλλαγή των γραφείων, για την εφαλλαγή των γραφείων που είχαν γίνει χώροι συλλογική εργασίας, αυτά τα open space, και στόχος ήταν να ε, αναδιατάξουμε τα γραφεία μετά από έρευνα που έγινε, δημοσκόπηση στο προσωπικό, ε, το οποίο είχε εκφράσει δυσφορία και δυσαρέσκεια με την κατάσταση αυτή του open space. Αυτό η μέρη οφειλόταν σε προβλήματα και δυσκολίες συγκέντρωσης, ε, θερμοκρασία στα γραφεία, ε, και επειδή αυξήθηκε σημαντικά ο φόρτος εργασίας και στη συνέχεια μειώθηκε και το προσωπικό στις υπηρεσίες αυτές, ε, συστήθηκε ομάδα εργασίας ε, που ε, εξέτασε το θέμα και κατέληξε ότι καλό θα ήταν όχι να επανέλθουμε στην παρελθούσα κατάσταση, αλλά να επιλέξουμε μια νέα φόρμουλα. Να έχουμε βέβαια ατομικά γραφεία, αλλά πιο μικρά από ό,τι στο παρελθόν και ένα μεικτό σύστημα να υπάρχουν και συλλογικοί ειδικοί χώροι για συνεδριάσεις, για συναντήσεις, αντί να υπάρχει ένας ενιαίος χώρος open space ανοιχτός όπου να εργάζονται όλοι. Ε, ε, οι ασκούμενοι παίρνουν μια υποτροφία, μια, ένα είδος μισθού, 1120 ευρώ συγκεκριμένα. Το δικαστήριο συνεισφέρει επίσης τα οδηπορικά ε, των ασκουμένων. Αρκεί αυτό για, σε σχέση με το επίπεδο ζωής στο Λουξεμβούργο. Έγινε μια συγκριτική μελέτη ε, και είδαμε τι δίνουν τα άλλα θεσμικά όργανα. Ε, στόχος είναι να είμαστε κάπως ευθυγραμμισμένοι και με τους υπολείπους. Θα δούμε. <laughs> Πώς θα εξελιχθεί το βιωτικό επίπεδο στο Λουξεμβούργο και μπορεί να χρειαστεί αναθεώρηση ε, του ποσού αυτού για να γίνει αυτό αρκεί μια απλή απόφαση του Γενικού Γραμματέα. Γιατί αυτό δεν το ορίζει κάποιο ειδικό γενικό καθεστώς. Ε, μπορεί να γίνει με μια απόφαση πιο γρήγορα και πιο εύκολα. Σε ό,τι αφορά τη δήλωση των πόθεν έσχεση οικονομικών συμφερόντων των μελών του δικαστηρίου, όντως δεν έχουμε την πρόθεση να τα δημοσιεύουμε. Ε, είδαμε τι γίνεται στα ανώτατα δικαστήρια των κρατών μελών ε, καθόλου διαδεδομένη δεν είναι αυτή η πρακτική της δημοσιοποίησης. Έχει και μια ιδιαιτερότητα το δικαστήριο, ε, απέτηση ανεξαρτησίας των δικαστών και των δικαιοδοτικών οργάνων και θεωρούμε ότι η δημοσίευση των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων ενώ δεν προσφέρει επιπλέον εγγύησεις ε, αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων. Θα μπορούσε να είναι όμως πηγή ε, ε, άσκησης πίεσης που θα έθετε σε κίνδυνο την ανεξαρτησία των δικαστών. Σε ό,τι αφορά το νέο προσωπικό σε σχέση με τον προπολογισμό, δεν ξέρω αν κατάλαβα πολύ καλά τη διερμηνία. Δεν κατάλαβα τι με ρωτήσατε. Είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω όποτε θέλετε, για να σας διευκρινίσω. Και τελευταία ερώτηση που είχε να κάνει με τη διάρκεια ε, διεκπαιρέωσης μιας υπόθεσης. Στην αρχή σας έδωσα τα στοιχεία κατά μέσο όρο το 18 ε, στο δικαστήριο και στο διοικητικό ε, δικαστήριο, το πρώτο βάθμιο. Εκεί η μέση διάρκεια των διαδικασιών είναι σαφώς χαμηλότερη ε, από την προηγούμενη, ε, πριν τη μεταρρύθμιση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι, γιατί το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τώρα και το διοικητικό και τα δύο μαζί διεκπερώνουν πολύ περισσότερες υποθέσεις και είναι και πολλές οι πρωτοβουλίες για να παραμένει λογική η διάρκεια όπως ορίζει το άρθρο 47 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ. Το ελεγκτικό συνέδριο. Έχετε το λόγο. Θα ξεκινήσω με την ερώτηση που έγινε για την υπόθεση που έστειλε το ελεγκτικό συνέδριο στην Όλαφ για ένα πρώην μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου και βρισκόμαστε στο εξή σημείο. Έχουμε ήδη ανακτήσει τα χρεωστή τους καταβληθέντα 153.000 ευρώ και αυτή τη στιγμή η υπόθεση έχει πάει στο δικαστήριο, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η Όλαφ έστειλε στην εισαγγελία στο Λουξεμβούργο τα σχετικά στοιχεία έτσι ώστε το πρώην μέλος να χάσει ε, την προστασία τη δικαστική και να ε, λογοδοτήσει και ο εσωτερικός μας έλεγχος κατέληξε, ευχαριστώ πάρα πολύ, ε, στο ότι ήταν μια μεμονωμένη περίπτωση, έχει αρθεί ασυλία, δεν είναι μια πιο διευρυμένη απάτη. Ο εσωτερικός έλεγχος επίσης κατέληξε πως η ελέγχη που κάναμε για την λειτουργία των συστημάτων είναι επαρκής και ο Γενικός Γραμματέας από εδώ και στο εξής εγκρίνει όλες τις αποστολές οι οποίες ελέγχονται όπως και όλες των υπαλλήλων του ελεγκτικού συνεδρίου είναι το σύστημα που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το σύστημα MIPS που έχει αυτοματοποιημένους ελέγχους ε, κατασταλτικούς ε, και ε, προληπτικούς και έδειξε αυτό πως δεν είχαμε σφάλματα ή λάθη γιατί όλες οι αποστολές όλες των, ε, όλου του ελληνικού συνεδρίου δημοσιεύονται στο ίντερνετ και αυτό για να ενισχύσουμε και τη διαφάνεια. Τώρα για το πρόγραμμα εργασίας να σας πω πως για το 2020 οι προτεραιότητες θα είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, η ανάπτυξη και η σε ευκαιρίες, η ασφάλεια, η μετανάστευση και η ενιαία αγορά. Εγκρίναμε πρόσφατα το πρόγραμμα εργασίας για την επόμενη χρονιά και πρέπει να σας πω πως όπως πάντα ο πρόεδρος του ελεγκτικού συνεδρίου θα έρθει εδώ στην επιτροπή σας για να σας παρουσιάσει το πρόγραμμά μας. Εγώ θα σας στείλω επίσης το πρόγραμμα εργασίας που θα εγκρίνουμε για να μπορέσετε κι εσείς να το έχετε διαθέσιμο. Τώρα για τις δηλώσεις που έχουν γίνει για τα οικονομικά συμφέροντα των μελών του ελεκτικού συνεδρίου δημοσιεύονται στο ίντερνετ όπως σας είπα και φέτος έγινε μία αναθεώρηση ε, ε, τύπου peer review με τους ομολόγους μας από την Κροατία και την Πολωνία για το σύστημα ακεραιότητας και ηθικής ε, ε, του δεοντολογίας του ελεγκτικού συνεδρίου και στην έκθεση αυτή συμπεριλαμβάνεται η αναθεώρηση αυτών των δηλώσεων και εξέταση αυτών για να δούμε αν μπορούν με κάποιο τρόπο να βελτιωθούμε. Έχουν και το σχέδιο δράσης το οποίο θεωρούμε ότι θα καταφέρουμε με τον τρόπο αυτό να φέρουμε σε πέρας για τα μέτρα ε, για την ισότητα του δικαστήριο έχει αυτή τη στιγμή εγκρίνει ένα πρόγραμμα ισότητας ευκαιριών, το οποίο θα στείλουμε μαζί με τα προηγούμενα και το οποίο αποτελείται από μία σειρά μέτρα, για παράδειγμα επιμόρφωση, ευαισθητοποίηση, ιδιαίτερη προσοχή ε, στην κατάρτιση των γυναικών έτσι ώστε να αναλάβουν διευθυντικές θέσεις και το στοιχείο αυτό θα λαμβάνει υπόψη σε όλες τις διαδικασίες, για παράδειγμα πρόληψης, προαγωγής, για να είμαστε σίγουροι πως δεν υπάρχει καμία παρεκτροπή ή κανένα πρόβλημα σχετικό με την ισότητα των φύλων. Το πρόγραμμα αυτό γίνεται σε στενή συνεργασία με, το σχετικό, με τη σχετική υπηρεσία στο Βίλνιους. Θα σας στείλω και αυτό το κείμενο και είμαστε στη διάθεσή σας για να απαντήσουμε ε, σε σχόλια δικά σας ή σε κάποιες προτάσεις οι οποίες επιθυμείτε εσείς να κάνετε για να βελτιώσουμε αυτό το σχέδιο δράσης. Άκουσα και μία ερώτηση για το κατά πόσο είμαστε ελκυστικό θεσμικό όργανο. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε. Δηλαδή καμιά φορά κάνουμε και ακροβατικά για να το πετύχουμε και δεν είναι εύκολο. Εμείς δηλαδή λέμε πόσο πως προσφέρουμε ε, ε, μια ε, καριέρα διαφοροποιημένη στους ελεγκτές μας. Έχουμε προγράμματα υποδοχής και ένταξης για όποιον έρχεται. Έχουμε εκπαιδευτικές δυνατότητες. Ένα κάμπους στο οποίο τους καλούμε να επισκεφθούν το ελεκτικό συνέδριο και τους δίνουμε όλων των ειδών τις ευκαιρίες για να τους προσελκύσουμε, αλλά δεν είναι εύκολο. Γιατί? Γιατί, ξέρετε, πως θα πρέπει να ανταγωνιστούμε με τους μισθούς της Βρυξέλλες και όπως ξέρετε κι εσείς έχουμε τον ίδιο συντελεστή διορθωτικό στο Λουξεμβούριο και στο Βρυξέλλες και παρόλα αυτά, παρόλο που έχουμε τους ίδιους μισθούς, είναι πολύ πιο ακριβό το Λουξεμβούργο και κυρίως ε, ε στο θέμα της στέγης. Ένα πρόβλημα το οποίο προσπαθούμε συνέχεια να αντιμετωπίσουμε και δεν είναι κατά πόσο είναι, μα αλλά είναι θέμα κοινωνικής δικαιοσύνης. Ο ελάχιστος μισθός στο Λουξεμβούργο είναι πιο υψηλός από αυτό που προσφέρει ένας ευρωπαϊκός θεσμός στους εργαζόμενους. Αυτό το διορθώσαμε με πολλή προσπάθεια, πολλές δυσκολίες και ήθελα να σας το αναφέρω γιατί πρέπει να το γνωρίζετε. Θεωρούμε πως είναι άδικο και δεν θα πρέπει να γίνει αυτό αποδεκτό. Δεν μπορούμε να θεωρούμε πως άνθρωπος ο οποίος εργάζεται στα ευρωπαϊκά όργανα θα έχει χαμηλότερο μισθό από τον ε, ελάχιστο μισθό που θεωρούν ε, απαραίτητο ε, αρχές για τους εργαζόμενους στη χώρα τους. Τώρα, για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια να σας πω το εξή. Έχουμε και ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο για να μπορούν να επιμορφωθούν ε, στο Πανεπιστήμιο του Νανσί οι ε, ελεγκτές μας είναι ένα ε, μάστερ σε δεύτερο επίπεδο στην οικονομία και ένα μάστερ στη στατιστική μπορούν να πάνε και κάνουμε και θερινικά μαθήματα ανοιχτά σε όλους τους υπαλλήλους μας, σε όλους τους ελεγκτές δηλαδή και σε όποιον ενδιαφέρεται για θέματα ελεγκτικά. Αυτό πηγαίνει, μπορεί κανείς να πάει και στο Πανεπιστήμιο της Πίζα στην Ιταλία με ανάλυση δεδομένων και ε, εργαλεία πληροφορικής. Επίσης, έχουμε και μία αντίστοιχη ε, δράση με το Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας. Συμφωνίες, λοιπόν, και ε, το Πανεπιστήμιο στην Πρίζ. Έτσι, λοιπόν, χρησιμοποιούμε τους καθηγητές και την εμπειρία που έχουν αυτά τα διάφορα πανεπιστήμια. Προσφέρουμε και υποτροφίες, μπορούν να πάνε σε διάφορα ε, πανεπιστήμια, αλλά έρχονται και από πανεπιστήμια, από τη Σορβόνη, από την Καστίγια Λαμάντσα και από άλλα πανεπιστήμια. Για τον έλεγχο της ΕΤΕ, περιορισμένη εντολή, γνωρίζετε κι εσείς πως έχει η ΕΤΕ δικούς της ελεγκτές για τους δικούς της ε, πόρους, ίδιους πόρους. Εμείς απλώς περιορίζουμε την εντολή μας στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται ε, τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το ΕΦΣΙ για παράδειγμα. Και στις εκθέσεις μας, στο ελεγκτικό μας πεδίο συμπεριλαμβάνουμε και αυτά τα κονδύλια από την ΕΤΕ. Αυτή τη στιγμή συζητάμε μαζί τους την ανανέωση αυτή τη τριμερού συμφωνία, που είναι η συμφωνία μεταξύ Κομισιών Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και ημών για να έχουν και τη νομική κάλυψη αυτή η έλεγχη. Για την ερώτηση για την εξοικονόμηση σε ταξίδια και οδηπορικά είναι ένα θέμα το οποίο είναι επίκαιρο. Το λαμβάνουμε υπόψη και σε αποστολές που κάνουμε και που δεν χρειάζεται να γίνουν ε, το έχουμε λάβει υπόψη. Κάνουμε βίντεο διασκέψεις και τηλεδιασκέψεις και μάλιστα πρέπει να σας πω πως ο αριθμός αποστολών και ταξιδιών που κάνουν οι ελεγκτές μας και κυρίως προς τις Βρυξέλλες έχουν μειωθεί. Όποτε μπορούμε, κάνουμε λοιπόν τηλεδιάσκεψη και κάνουμε όλο και περισσότερες. Ευχαριστώ. Muchas Ευχαριστώ πολύ. Και θα περάσουμε τώρα στην ε, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Έχετε το λόγο κύριε Μπρουνέτη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ομαδοποιήσω τις απαντήσεις γιατί ε, έτσι μπορούμε να εξοικονομήσουμε λίγο χρόνο. Θα ασχοληθώ πρώτα με την παρενόχληση. Και επαναλαμβάνω αυτό που είπα προηγουμένως για τα συγκεκριμένα μέτρα που έχει λάβει το θεσμικό μας όργανο. Καταρχάς, ε, προληπτικά, έχουμε μια εκστρατεία που ονομάζεται «Σεβασμό στη δουλειά», «Respect at work». Αυτό πλαισιώνει και το διοικητικό πλαίσιο που έχει πολύ ε, σαφείς ε, διατάξεις για το σεβασμό. Επίσης υπάρχουν και σύμβουλοι εμπιστοσύνης. Ήμασταν οι πρώτοι που τους θεσμίσαμε, είχαμε πέντε, τώρα είναι έξι τα μέλη μας έχουν κώδικα δεοντολογίας όπου απερίφραστα ορίζεται η υποχρέωση να γίνεται σεβαστή η αξιοπρέπεια ε, στο χώρο εργασίας. Εγκρίθηκε το Μάρτιο και κάθε φορά που έχουμε κάποιες καταγγελίες, κάθε φορά επαναλαμβάνω, αυτές διεκπεραιώνονται με βάση τον ε, κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης και τον ιστορικό κανονισμό και τη διδολογία. Επίσης, ε, στην ανανέωση που θα γίνει του χρόνου το φθινόπωρο, ε, θα προσθέσουμε και αυτή τη δυνατότητα εκπαίδευση στο μελό μας. Πολύ καλή ιδέα πέρα από το σεβασμό δηλαδή θα πρέπει να μάθουν τι σημαίνει να εργάζονται σε ένα περιβάλλον πολυπολιτισμικό και πολύγλωσσο. Ε, σε ό,τι αφορά την επιλογή ε, του Γενικού Γραμματέα και του ανώτατου προσωπικού. Ε, η απάντηση είναι στην ερώτηση 34. Είμαστε περήφανοι πρέπει να σας πω για τις διαδικασίες μας. Είναι πάρα πολύ διαφανείς και αποτελούν πρότυπο, ε, παράδειγμα προς μίμηση για τα άλλα θεσμικά όργανα. Εδώ και 10 χρόνια κάθε φορά που χειρεύει η θέση του Γενικού Γραμματέα δημοσιεύεται, προκυρήσεται η θέση στην επίσημη εφημερίδα σε όλες τις γλώσσες. Το Προεδρία μας που είναι το πολιτικό όργανο ορίζει ένα αριθμό μελών ε, που διαπιστώνει και εγκρίνει την προκήρυξη, ε, ότι χειρεύει η θέση και προκηρύσσεται και ε, στα social media. Στη συνέχεια έχουμε ένα πάνελ που ορίζεται πάλι από το Προεδρείο, τα μέλη της Επιτροπής Εξεταστικής και οι επιλαχόντες αυτοί υποψήφοι πηγαίνουν ε, σε ένα κέντρο αξιολόγησης που είναι στην έψω ουσιαστικά που παρέχει αυτές τις υπηρεσίες. Και μετά ε, ε, υπάρχει και άλλη συνέντευξη με τον υποψήφιο και τελική επιλογή. Αυτό τηρουμένο των αναλλαγιών με κάποιες παραλλαγές εφαρμόζεται και στις θέσεις διευθυντών στις ανώτατες βαθμίδες της διοίκησης. ρωτήσατε πώς μπορούμε να ελέγξουμε και να μειώσουμε τις δαπάνες των μελών της ΟΚΕ. Εδώ θα ήθελα να θυμίσω κάτι. Τα μέλη μας δεν είναι οι υπάλληλοι μας. Ε, δουλεύουν στους οργανισμούς τους τα κράτη-μέλη έρχονται στις Βρυξέλλες μόνο για να συμμετέχουν στην νομοθετική αυτή ε, ε, δραστηριότητα. Αλλά επειδή έχουν και άλλη θέση, υπάρχουν δύο στοιχεία τα οποία εμείς δεν ελέγχουμε. Το πρώτο είναι η νομοθετική, το νομοθετικό χρονοδιάγραμμα. Έρχονται τα αιτήματα σε εμά όταν μας διαβάζουν κείμενα οι νομοθέτες. Το δεύτερο στοιχείο, και το συνδέω ήδη αυτό και με μια ερώτηση που έγινε προηγουμένως, ότι έχουμε τα ίδια κτίρια με την Επιτροπή των Περιφερειών. Εδώ γίνονται πολλές οικονομίες, αλλά εμείς δεν είμαστε κύριοι του ε, ε, ημερολογίου, του, του χρονοδιαγράμματός μας. Θα πρέπει ένα χρόνο πριν να προβλέπουμε τις αίθουσε και όλη την επιμελητία. Αυτό επηρεάζει έτσι κι αλλιώς ε, την ευελιξία. Τι συμβαίνει λοιπόν και έχουμε ένα προϋπολογισμό για τα οδηπορικά των μελών και την διαμονή τους που είναι γύρω στο 15% του συνολικού προϋπολογισμού. 5% είναι για τη διαμονή. Τι κάνουμε για να προγραμματίσουμε και να προσπαθούμε να ελέγχουμε αυτές τις δαπάνες. Έχουμε ένα πρόγραμμα software που είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο και ακριβές για τις δαπάνες και τώρα να θεωρείται κιόλας και έχουμε και μια ευρεία πολιτική απέναντι στα μέλη. Ε, τους ε, καλούμε να χρησιμοποιούν ε, πιο οικονομικό τρόπο κράτησης αεροπορικών εισιτηρίων από νωρίς, εκ των προτέρων, διασταυρούμενες, ακόμα και εταιρείε χαμηλού κόστους. Το 20% ε, των ταξιδιών, των αεροπορικών γίνονται ε, είτε σε οικονομική θέση είτε με εταιρείε σε low cost. Υπάρχουν οι τεχνολογικές δυνατότητες ε, αυτή τη στιγμή ε, όμως που δεν μας επιτρέπουν να έχουμε διερμηνία εξ αποστάσεως και τηλεδιασκέψεις, ε, θα πρέπει να είναι παρόντα στον ίδιο χώρο τα μέλη μας για να μπορούν να συζητούν, να ανταλλάσσουν απόψεις και να αποφαίνονται για τα νομοθετικά κείμενα. Ε, έγινε ερώτηση για την εξωτερήκευση της μετάφρασης και αν είμαστε ικανοποιημένοι ή όχι. Από πλευράς ποιότητας, όταν εξωτερικεύεις, είσαι πάντα λίγο πιο απαιτητικός και αν μπορώ να χρησιμοποιήσω μια έκφραση έτσι όχι πάρα πολύ κομψή, είμαστε συγκρατημένα ικανοποιημένοι. 20% ήταν η εξωτερικεύση, αλλά ε, αυτό εξαρτάται και από το φόρτο εργασίας. Αν μειώνεται η νομοθετική δραστηριότητα, μειώνεται και η μεταφραστική δραστηριότητα, αναγκαστικά και τούμπαλιν. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να έχουμε κάποιους εσωτερικούς μεταφραστές, μια δυνατότητα όταν υπάρχει φόρτο εργασίας. Ε, γενικά Εντάξει, αλλά θα πρέπει να κάνουμε προσπάθειες για να εξωτερικεύσουμε ακόμα περισσότερο, να αναθέτουμε εξωτερικά. Βεβαίως, μιλώ υπό την αίρεση των όσων θα πούν οι συνάλληλοι από την Επιτροπή των Περιφερειών. Euh, Έρχομαι τώρα στη συνεργασία με την Επιτροπή των Περιφερειών αναφερθήκαμε στις οικονομίες που έχουμε από αυτή τη συνεργασία, της ε, απαντήσεις. Για τις δύο επιτροπές αυτό ανέρχεται σε 20 εκατομμύρια. Δεν είναι ευκαταφρόνητο το ποσό. Έχει να κάνει με τεχνικά θέματα αλλά και οικονομίες στο προσωπικό. Είναι αρκετά καλό παράδειγμα και, και σημαντικό που δείχνει με ποιο τρόπο μπορούν να εργαστούν τα θεσμικά όργανα όταν σέβονται τα χρήματα των φορολογουμένων και πώς μπορούν να κάνουν σημαντικές οικονομίες. Εμείς έχουμε δεσμευτεί βέβαια να κάνουμε περισσότερα. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή με τη Συμφωνία Συνεργασίας. Η σημερινή συμφωνία εκπνέει ε, στις 31 Δωδεκάτου. Ήδη προετοιμάζεται η επόμενη ανανέωσή της και ενίσχυσή της σε ορισμένα σημεία και προς το παρόν έχει αποφασιστεί να ανανεωθεί η συμφωνία αυτή μέχρι τα τέλη του 2020. Βέβαια θα πρέπει επίσημα να πάρουν την απόφαση και οι πολιτικοί θύνοντες ε, πρόεδροι για να δούμε πώς μπορούμε καλύτερα ακόμα να συνεργαστούμε. Πάντως, ε, είναι σημαντική η πρόοδος που έχουμε κάνει. Κάποιες μονάδες μετάφρασης προβλέπεται να ε, συγχωνευτούν. Στην αρχή ήταν δύο ζεύγοι ε, μονάδων ε, τμήματων, τώρα είναι εννέα παρακαλώ. Επίσης πρέπει να σας πω ότι ε, σε ό,τι αφορά τη συνεργασία μας, η μεγαλύτερη φετινή επιτυχία είναι ότι τα δύο θεσμικά όργανα συμφώνησαν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την ε, ε, ενεργή υποστήριξη του Επιτρόπου Τιγκέρ, να ανταλλάξουμε δύο κτίρια μας με το κτίριο Βαν Μάρλαντ, που ήταν ένα παλιό κτίριο του Κοινοβουλίου για όσους είναι συνομιλικοί μου. Βέβαια, αυτό ε, ε, ε, σημαίνει οικονομίες, αλλά απώλεια εμβαδού. 10.000 τετραγωνικά χάνουμε. Δηλαδή 200 γραφεία. Euh, σύμφωνα με τον τρόπο με τον οποίο μοιραζόμαστε τα γραφεία με την Επιτροπή των Περιφερειών. Όταν μιλάμε για το χώρο εργασία του μέλλοντος, φυσικά είναι ένα θέμα που μας προβληματίζει και μα απασχολεί να δούμε πώς μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε το μειωμένο χώρο, μετατοπίζοντας εσωτερικά χωρίσματα, γιατί δεν είναι τύχη, ε, αυξάνοντας ε, τους χώρους ε, που μοιράζονται οι εργαζόμενοι ή αυξάνεται και ο αριθμός των ε, εργαζομένο σε τηλεεργασία, καθώς το επιτρέπουν αυτό οι νέες δυνατότητες τεχνολογίας και της πληροφορική. Είμαι στη διάθεσή σας για τυχόν ε, περισσότερες ερωτήσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, Επιτροπή των Περιφερειών, κύριε Σερβίγια Μαρτίνες, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα μου επιτρέψετε καταρχήν να σας ευχαριστήσω για τα εισαγωγικά σας σχόλια γενικότερα, για τη σημασία ε, που έχει η Επιτροπή μας και για τη στήριξη που μας έχετε προσφέρει για να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα όλων των θεσμικών οργάνων. Είμαστε πολιτικό όργανο ε, και δεν μπορούμε παρά να συμμεριζόμαστε ε, τα λεγόμενά σας. Εάν μου επιτρέψετε, στις ερωτήσεις της δικές σας θα απαντήσω παράλληλα με τις ερωτήσεις που μας έκανε ο εισηγητής και θα δώσω κάποια στοιχεία έτσι ώστε μετά εσείς να καταλήξετε στα συμπεράσματα που πρέπει. Το λέω λοιπόν για τον εισηγητή γιατί ενδεχομένως δεν τα γνωρίζει. Μετά την προηγούμενη απαλλαγή είχαμε την ε, απόφαση του δικαστηρίου το 2018 ε, για την προηγούμενη ε, Επιτροπή ε, για τις ε, αναπηρίες καινούρια με γιατρό από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ευχαριστούμε τις υπηρεσίε του Κοινοβουλίου που παρίσταται στις συνεδριάσεις αυτής της Επιτροπής που ασχολείται με τις ανικανότητες και τις αναπηρίες και το Μάιο του 2019 αυτή η Επιτροπή αποφάσισε πως η ασθένεια ήταν επαγγελματικής ε, προέλευσης. Το Προεδρείο και ο Γενικός Γραμματέας ενέκριναν την απόφαση της επιστροφής και της οικονομικής αποζημίωσης των ποσών ε, στον πρώην ελεγκτή. Ο πρώην ελεγκτής, όπως γνωρίζετε κι εσείς, ζητά επιπλέον αποζημίωση και επιστροφές. Εσείς είστε η Επιτροπή Ελέγχου των Προπλογισμών και ζητάτε από τη δική μας Επιτροπή να μπει σε μία ε, διαδικασία διαμεσολάβησης με ένα μέλος και αυτή τη στιγμή εσείς τυχαία έχετε λάβει το αποτέλεσμα που είναι η συγκεκριμένη απάντηση του Προέδρου μας που έδωσε συγκεκριμένη ημερομηνία κατά την οποία οι δικές μας πολιτικές αρχές και η δική, και η μας διοίκηση παρουσία ενό μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα συναντηθεί με αυτόν τον πρώην ελεγκτή. Ελπίζουμε πως με τον τρόπο αυτό θα λυθεί μια και καλή αυτό το θέμα. Γενικά ο εισηγητής μας ρώτησε τι γίνεται με άλλου είδους, ε, τέτοιου είδες ε, περιπτώσεις όχλησης. Ε, νομίζω ότι δεν έχουμε άλλες περιπτώσεις παρενόχλησης, οι άλλοι αναφέρθηκαν. Να προσθέσω μόνο πως 4 Δεκεμβρίου ή 5 στην Ολομέλειά μας θα εγκριθεί ένας ε, δεοντολογικός κώδικας για τα μέλη της Επιτροπής μας με πολύ λεπτομερείς διατάξεις για να αποφευθεί ε, οποιαδήποτε περίπτωση ενδεχόμενης παρενόχλησης από μέλος της Επιτροπής προς προσωπικό της Επιτροπής μας. Πολύ λεπτομερής, πολύ αυστηρός, πολύ ε, στην ίδια γραμμή με τα όσα ισχύουν εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για τα υπόλοιπα θέματα, ο συνάδελφος Τζανλούκα Μπρουνέτη από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή απάντησε δεν θα φέρω οποιαδήποτε αντίρρηση και αντίθετα θα πω ότι αυτό το 20 με 25% της εξωτερήκευσης ε, της ε, εξωτερικής ανάθεσης μετάφρασης γίνεται. Το ζήτημα είναι τι θα γίνει με τη νέα επιτροπή. Και αν συνεχίσετε να δουλεύετε στον ίδιο ρυθμό. Αν αυξήσετε εσείς το ρυθμό σας και χρειαστεί εμείς να, να υποβάλουμε περισσότερες γνωμοδοτήσεις, τότε και οι μεταφραστές θα πρέπει να κάνουν περισσότερη δουλειά και αυτό το 20 με 25% δεν ξέρω αν θα είναι αρκετό. Η ανανέωση συμφωνίας δεν υπάρχει τίποτα εδώ να σχολιάσω, παρατείνεται γιατί λειτουργεί σωστά και στις ενδεχόμενες βελτιώσεις ε, θα τις δούμε με μεγαλύτερη άνεση Άρα λοιπόν εκεί δεν έχω κάτι να πω. Ό,τι είπε ο συνάδελφος. Το ίδιο ισχύει για τα πλέον εκτήματα τα συγκεκριμένα. Μπορούμε να τα ποσοτικοποιήσουμε και να πούμε 20 εκατομμύρια και θα μπορούσαν αυτά να πολλαπλασιαστούν. Να μπούμε και σε μια συζήτηση, αλλά προφανέστατα επειδή έχουμε αυτά τα κοινά ε, ε, αυτό το κοινό προσωπικό και τα κοινά κτίρια και εγκαταστάσεις ε, νομίζω ότι είναι πάντα πλεονέκτημα για όλους. Κάναμε και μία εκτίμηση της ακίνητης περιουσίας για το 2020 με 2022 η αξία παραμένει ε, η ίδια, η ανταλλαγή με το κτίριο συνεχίζεται και με τη Βαμέρλαν και με το άλλο κτίριο που έχουμε ανταλλάξει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αν μου επιτρέψετε το περίμπεφημο νέο σύστημα εργασίας θα το αφήσω αργότερα, γιατί είναι κυριολεκτικά κάτι πάρα πολύ περίπλοκο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το δουλεύει 10 χρόνια, δεν έχει ακόμα καταλήξει συγκεκριμένα ε, εδώ και 10 χρόνια το κοιτάει, είναι αυτά τα τρία β, τα οποία ακόμα δεν έχουν βρει μια λύση, αλλά θα δούμε τι μπορεί να κάνει η νέα τεχνολογία ή η ψηφιακή στρατηγική ή τηλεεργασία, όλα αυτά μπορεί να μας βοηθήσουν για να χρησιμοποιούμε, χρησιμοποιούμε καλύτερα τους χώρους που έχουμε στη διάθεσή μας. Ε, por la defensora del pueblo, señora Danielo, tiene la palabra. Σας Ευχαριστώ πολύ. Ε, είχα πολλές ερωτήσεις ε, και θα τις εξετάσω με τη σειρά. Ε, ξεκινάω με τις ερωτήσεις που ήρθαν από τον εισηγητή για το νέο καταστατικό. Αυτός είναι ένας τομέας ειδικής νομοθετικής πρωτοβουλίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η διαδικασία ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα Είχαμε τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ακολούθησε μετά τη νομική άποψη του Συμβουλίου, το οποίο πρέπει να συνενέσει στη διαδικασία. Η δική μας θέση είναι ότι εμείς ε, δεν ε, ζητάμε τίποτα, αλλά είμαστε έτοιμοι, όπως συνέβη και κατά το παρελθόν, να προσφέρουμε οποιαδήποτε ε, πληροφορία είναι απαραίτητη, όχι μόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και στους τρεις θεσμούς, όσον αφορά τις τεχνικές τυχές της εργασίας μας. Ε, η διαμεσολαβήτρια εμφανίστηκε στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και αυτή των αναφορών και τώρα αυτό ίσως είναι πιο σημαντικό γιατί έχουμε ε, την άποψη του Συμβουλίου και της Επιτροπής, άρα δηλαδή είμαστε στη διάθεσή σας ε, σε οποιοδήποτε επίπεδο. Τώρα, το άλλο ερώτημα. Ε, βεβαίως και πρέπει να ανταλλάσσουμε τις βέλτιστες πρακτικές, να τις ε, διαθέτουμε στον ηθικό τομέα να υπάρχουν αυτές στην ιστοσελίδα μας. Είμαστε ανοιχτοί σε αυτό. Η δική μας ιστοσελίδα περιλαμβάνει ήδη τις ε, εσωτερικές μας πολιτικές, αλλά είναι καλύτερα να υπάρχει και καλύτερη οργάνωση. Και μπορώ να σας πω ότι από τότε που ξεκίνησα, πριν από ένα χρόνο περίπου, κάτι παραπάνω, έκτοτε αναθεωρώ όλες τις εσωτερικές πολιτικές, γιατί πιστεύω ότι για ένα γραφείο όπως είναι αυτό του διαμεσολαβητή είναι πολύ σημαντικό ε, να είμαστε ενημερωμένοι κυρίως σε θέματα ηθικής. Ε, βρίσκομαι στα μέσα αυτής της δουλειάς. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι είναι μια θαυμάσια ιδέα την οποία και θα συζητήσω με τους συνεργάτες μου. Ε, κατόπιν είμαι ευγνώμων κυρία Πρόεδρε για την ερώτηση ε, που αφορά τους συμβασιούχους διότι κατ' ουσίαν αντικατοπτρίζει μια προτεραιότητά μας και έχουμε υποβάλει ε, μια λεπτομερή πρόταση στην Επιτροπή Προϋπολογισμού του Συμβουλίου και προφανώς και του Κοινοβουλίου όπου ισχυριζόμαστε ότι σε ένα μικρό γραφείο όπως είναι το δικό μας το να είναι το 20% συμβαχιούχοι που εργάζονται πολύ στενά με τους μόνιμους και πολύ συχνά ε, κάνουν την ίδια την παρεμπερή δουλειά. Αυτό δεν είναι και πολύ καλό γιατί πολύ εύκολα μπορεί να οδηγήσει σε απογοήτευση. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε καταθέσει λεπτομερή πρόταση στην αρχή προϋπολογισμού να αλλάξει αυτό το 20% των συμβασιούχων ε, να είναι κανονικές, ε, οργανικές οι θέσεις ή μόνιμες ή όπως το προτιμά η αρχή προϋπολογισμού, να είναι ε, προσωρινή ή με σύμβαση. Ε, τους ε, συμβασιούχους που έχουμε τώρα θα τους παίρνουμε μόνο αν χρειαστεί, αν δηλαδή κάποιοι υπάλληλοι φεύγουν ε, για λόγους τοκετού ή οτιδήποτε άλλο. Ε, να σας δώσω και άλλες λεπτομέρειες, αλλά πραγματικά ελπίζω ότι η αρμόδια αρχή προϋπολογισμού θα τοποθετηθεί θετικά στο αίτημά μας, το οποίο περιλαμβάνει ε, πολύ λίγες επιπρόσθετες δαπάνες, γιατί κατ' ουσίαν ε, τους, ε, τις συμβάσεις παρετούμεθα αυτών και προτείνουμε κάποιες επιπρόσθετες μόνιμες θέσεις. Άρα δηλαδή δεν θα υπάρχουν ε, επιπτώσεις στον προϋπολογισμό. Και η τελευταία ερώτηση Πράγματι είναι πολύ λυπηρή η κατάσταση, σωστό αυτό που είπατε ε, και πρέπει να επιβεβαιώσω ότι είμαστε ε, στα μέσα μιας εκστρατείας παραπληροφόρησης, έτσι την ορίζουμε. Υπάρχουν ε, ανώνυμα email τα οποία στέλνονται σε έναν ανώνυμο σερβερ κωδικογραφημένα, κωδικοποιημένα και αξ' έχουμε μετρήσει ότι περιλαμβάνουν κατ' ουσίαν τρεις επιθέσεις. Στη μία επίθεση παρουσιάζουν ε, λανθασμένα την έρευνα σχετικά με το προσωπικό. Στην άλλη επίθεση αναφέρονται στις επιπτώσεις της δουλειάς του Ευρωπαίου ε, διαμεσολαβητή και στην τρίτη επίθεση εκεί ε, προβαίνουν σε ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς ε, για κάποια γεγονότα που αφορούν το γραφείο μας. Όσον αφορά τις επιπτώσεις, ε, εγώ προσπάθησα στην ομιλία μου να παρουσιάσω πολλά θέματα που έχουν σχέση με τις επιπτώσεις που προκύπτουν από τη δουλειά μας. Έχουμε και την ετήσια έκθεση ε, που σήμερα εγκρίθηκε από την Επιτροπή Αναφορών με συντριπτική πλειοψηφία. Έτσι λοιπόν ε, όσον αφορά τις θετικές προεκτάσεις της δουλειάς μας. Ε, εμείς έχουμε υψηλό ποσοστό συμμόρφωσης, 81% και ε, άλλο ένα αντίστοιχο 85% για περιπτώσεις δημοσίου. Υπάρχουν ε, κάποιες περιπτώσεις που είναι πολύ σημαντικές γιατί έχουν στόχο να αλλάξουν την οτροπία του, της διοίκησης. Ε, δεν έχουμε άμεσα αποτελέσματα, αλλά ακόμα και στις περιπτώσεις όπου πρώτα ο θεσμός αρνείται τις συστάσεις του ε, διαμεσολαβητή, βλέπουμε όμως ότι υπάρχει μια, μια κινητικότητα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην θέσπιση ενός νέου κώδικα για τους επιτρόπους. Ε, θα μπορούσα να αναφέρω πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις, αλλά αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι πέρα από τις άμεσες αλλαγές, όπου οι θεσμοί συμμορφώνται σε πολύ ψηλό επίπεδο, το όφελος για τους ε, πολίτες και για ευρύτερα ακροατήρια όπου αυτοί που οι θεσμοί συμμορφώνονται και η πόρτεση είναι προς όφελος ε, το, του πολίτη, υπάρχει και μία αργή μετακίνηση στην οτροπία της διοίκησης. Ε, ευαίσθητες περιπτώσεις όπου αρνητική η πρώτη αντίδραση, αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε μια αργη μετακινηση στην οτροπια της διοικησης ε περιπτώσει, περιπτωσεις οπου αρνητικη η πρωτη αντιδραση αλλα παρολα αυτα βλεπουμε μια κινητικοτητα Και για να επανέλθω στο ερώτημα, εγώ πραγματικά το βρίσκω πάρα πολύ δύσκολο να ισχυρίζεται κανείς ότι η ε, προεκτάσεις της δουλειάς του, της διαμεσολαβήτριας ε, είναι περιορισμένες. Κατόπιν έχουμε, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη ψέματα, αλλά ας πούμε για ε, παραπλάνηση σε σχέση με κάποια γεγονότα που αφορούν στο γραφείο μας. Ένα από αυτών είναι ότι το γραφείο μας εξαρτάται από νομικές συμβουλές. Δεν είναι έτσι όμως. Έχουμε 120 περιπτώσεις που ερευνούνται και με αυτές ασχολούνται άνθρωποι που είναι δικηγόροι. Άρα δηλαδή αυτό είναι μόνιμο στο γραφείο μας ότι εξετάζουμε τη νομική συμμόρφωση. Μερικές φορές ε, προσλαμβάνουμε ε, ταλαντούχους νέους που δεν είναι ε, δικηγόροι, αλλά δεν είμαστε και δικαστήριο, θα ήταν και σχεδόν υπερβολικό να επιτρέπουμε να προσληφθεί σε εμά κάποιος μόνο εφόσον είναι δικηγόρος. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα ε, λάθος ισχυρισμοί που αφορούν ε, την ίδια τη διαμεσολαβήτρια, ε, την υποφαινόμενη δηλαδή, αναφέρονται σε κάποια στοιχεία της καριέρας μου. Και επίσης υπάρχει και χρήση μιας εσωτερικής έρευνας που δεν ε, έχει ε, δεν έχουν κοινοποιηθεί αυτά τα email Θα μπορούσα να σας αναφέρω κάποια παραδείγματα. Ε, το site αναφέρει αρνητικά ε, στατιστικά δεδομένα. Ε, γίνεται λόγος για το ποσοστό των στατιστικών δεδομένων προσθέτοντας ουδέτερες απαντήσεις, δηλαδή δεν έχω άποψη ή καμία απάντηση. Και βεβαίως φτάνουμε σε ένα πολύ υψηλό ποσοστό αρνητικών δηλώσεων. Μπορώ να σας αναφέρω συγκεκριμένα τις σελίδες όπου όλα αυτά ε, περιλαμβάνονται ε, στις έρευνες. Και θα ήθελα επίση να πω ότι δεν αναφέρουν καθόλου προφανώς, γιατί αυτό είναι και ο στόχος των email, δεν αναφέρουν ότι η έρευνα για το προσωπικό περιλαμβάνει πολύ ε, θετικά παραδείγματα. Παράδειγμα, το 75% είναι ευχαριστημένο με το εργασιακό περιβάλλον, το 67% είναι ευχαριστημένο με την ανταλλαγή πληροφοριών, το 57% ε, θέλει να ε, συμβάλλει σε βελτίωση του γραφείου. Όλα αυτά είναι αξιοσημείωτα διότι έχω κάνει παλαιότερα εμπειρία με έρευνες προσωπικού ε, που οργανώνονται από συνδικάτα, από επιτροπές προσωπικού. Βεβαίως ε, αντιμετωπίζονται ως ένα εργαλείο για να εντοπιστεί η απογοήτευση. Είναι λοιπόν αξιοσημείωτο το ότι έχουμε ε, πολλά και θετικά σχόλια ακόμα και σε μία έρευνα την οποία διεξάγει η Επιτροπή Προσωπικού. Δεν θέλω να ε, σας κουράσω, ε, να επαναλάβω μόνο ότι ε, πολύ ευχαριστώ να σας πω πολλές λεπτομέρειες που αφορούν το τι περιλαμβάνουν αυτά τα email, τα οποία όπως σας είπα εμείς τα θεωρούμε ως μια κλασική εκστρατεία παραπληροφόρησης και παραπλάνησης που αφορά ε, δημοκρατικές εκλογικές διαδικασίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Τέλος, στον επόπτη για την προστασία των δεδομένων, ο κύριος Νάβας. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι ήδη αργά, όλοι είναι πολύ κουρασμένοι. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να μιλήσω ισπανικά. Μια και έχουμε ευρωβουλευτή από την Ισπανία στην Προεδρία. Ευχαριστώ λοιπόν τον εισηγητή για τα θετικά του λόγια που υπογράμμισε τις ε, προσπάθειες που κάνουμε όλοι εμείς οι θεσμοί για να εκπληρώσουμε τις και να συμμορφωθούμε με τις υποχρεώσεις μας. Όντως έτσι γίνεται και πραγματικά τον ευχαριστώ που το αναγνωρίζει και θα ήθελα να ευχαριστήσω και το ελεγκτικό συνέδριο για τη δουλειά που κάνει για όλους μας που είναι πολλές φορές αφανής αλλά σημαντική για να έχουμε τη σωστή διαχείριση των διαθέσιμων πόρων. Τέσσερις ερωτήσεις έγιναν, θα τις απαντήσω επιγραμματικά. Νέα καθήκοντα. Τρία νέα καθήκοντα μέσω της νέας νομοθεσίας. Ε, γραμματεία σε ένα νέο οργανισμό, δηλαδή 25 άτομα. οργάνωση της εποπτείας των υπηρεσιών του πρώην τρίτου πυλώνα, Europol που είναι το Ευρωπαϊκό FBI να υποπτεύουμε την ε, βάση δεδομένων των αστυνομικών δεδομένων μου τεράστια πρόκληση και με τη νέα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων που ετέθησε εφαρμογή το 2018 έχουν νέες υποχρεώσεις, νέα καθήκοντα Πρέπει δηλαδή να κοινοποιούν ε, ε, διαρροές ε, δεδομένων στο υποπτικό όργανο. Αυτό συμβαίνει συχνά. Και τώρα πια μπορούμε να επιβάλλουμε πρόστιμα, για παράδειγμα, στα θεσμικά όργανα και επίσης να βοηθάμε τους αξιωματούχους για την προστασία δεδομένων των θεσμικών οργάνων στα καθήκοντά τους. Τώρα, σε δημοσιονομικό επίπεδο εμείς ζητήσαμε διεύρυνση μάλλον αύξηση 25% του προσωπικού για το 19 και το 2020, γιατί κάναμε μία μελέτη για το ποια ήταν η γενικότερη αύξηση των ε, πόρων μετά το GDPR ε, στις ε, υπηρεσίες προστασίας των προσωπικών δεδομένων σε εθνικό επίπεδο. Βρήκαμε ότι κάνανε γύρω στο 25% και είπαμε κάτι αντίστοιχο και εμείς. Ελπίζουμε πως τον προπολογισμό του 2020 θα ληφθεί αυτό υπόψη και θα μας δοθεί η αύξηση που ζητήσαμε. Μιλήσατε για το ηθικό πλαίσιο, το ιδεοντολογικό πλαίσιο. Για μας είναι ουσιαστικό. Θεωρούμε πως η ιδεοντολογία αποτελεί τη βάση όλων των ε, προσπαθειών που κάνουμε και όταν λείπει αυτή η ηθική διάσταση ξεκινά τα προβλήματα. Έχουμε λοιπόν αξιωματούχο για το συγκεκριμένο ε, που παρακολουθεί ε, τη διοντολογική συμπεριφορά του προσωπικού μας και προετοιμάζει μία έκθεση μια φορά το χρόνο τουλάχιστον για μια ειδική συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του οργάνου μας. Λειτουργεί καλά, είναι μια πρακτική την οποία θα ήθελα να συστήσω και στους υπόλοιπους. Επίσης για την ερώτηση που έγινε, γιατί έχουμε τόσο υψηλό ποσοστό συμβασιούχων, 40%, θα το πω ανοιχτά. έχει να κάνει με την κρίση και το πάγωμα το προϋπολογισμό όλων των ευρωπαϊκών οργάνων ε, τα τελευταία χρόνια. Αυτό. Για μας που ήμασταν στην φάση της ανάπτυξης, ο μόνος τρόπος με τα λίγα κονδύλια που είχαμε να συνεχίσουμε να γεμίζουμε τα γραφεία ήταν με συμβασιούχος που είναι πιο φθηνή από τους μόνιμους υπαλλήλου. Αυτή είναι η κατάσταση. Πέρσι κάναμε αυτή τη μεγάλη ε, διεθνή διάσκεψη και χρειάστηκε να ενισχύσουμε προσωπικά το προσωπικό μας για να καλύψουμε κάποιες ανάγκες. Εν πάση περιπτώσει συμφωνούμε και εμείς πως η κατάσταση αυτή είναι κακή, πως δεν είναι βιώσιμη. Και γι' αυτό προσπαθούμε να μειώσουμε αυτό το ποσοστό σε κάτι πιο λογικό. Οργανώσαμε δύο διαγωνισμούς μέσω έψω, πολύ πολύ δουλειά, αλλά το κάναμε για να μπορούμε να προσλάβουμε περισσότερους μόνιμους υπαλλήλου για να πέσουμε από το 40% στο 25% των συμβασιούχων το 2020. Και μετά θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε μειώνοντας αυτά τα ποσοστά. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Και για να κλείσουμε θα ξαναδώσω το λόγο στον εισηγητή, στον κύριο Σδεχόφσκι. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους ε, που ε, δαπανίσατε το χρόνο σας για να συζητήσουμε για το θέμα της απαλλαγής ε, για το 2019. Νομίζω ότι είναι το 2018. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί εμείς είμαστε εταίροι σας, δεν θέλουμε να σας επιτιθέμεθα, δεν είμαστε εχθροί. Και το λέω εδώ Είμαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πέντε χρόνια και συμμετείχα ε, σε όλες τις συζητήσεις απαλλαγής για άλλους ε, θεσμούς και πρέπει να σας πω ότι σήμερα και δεν είναι ότι είμαι μόνο εισηγητής, όχι μόνο γι' αυτό, αλλά σήμερα πραγματικά ήταν η καλύτερη ατμόσφαιρα που επικράτησε ποτέ σε τέτοιου είδου συζητήσει. Είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία και συζήτηση και γι' αυτό να πάτε ήσυχοι στο σπίτι σας, ε, να φροντίσετε τον εαυτό σας και τις οικογένειές σας. Είναι το πιο πολύτιμο που έχετε στη ζωή σας. Και αν κάποιος μπορεί να σε επικρίνει, νομίζω ότι ε, δεν μπορεί να σας επηρεάσει σε τελική ανάλυση. Σας εύχομαι τα καλύτερα. Σας ευχαριστώ και όλους εσάς για την τόσο ζωηρή συζήτηση και το διάλογο αυτό. Εγώ χρειάστηκε να προεδρεύσω εδώ, αλλά με τόσους Ισπανούς αισθάθηκα στο σπίτι μου, σαν την πατρίδα μου. Κυριάρχησαν τα Ισπανικά εδώ, σε τη συνεδρίαση αυτή. Θέλω να σας πω ότι η επόμενη συνεδρία θα γίνει στις 18 Νοεμβρίου από τις 3 μέχρι τις 6.30. Σας ευχαριστώ πολύ ε, και όπως και όλα τα μέλη της Επιτροπής. Καλό σας βράδυ.